Señorías, buenos días. Vamos a dar comienzo a la sesión de, de esta mañana, cuyo orden del día anunciaré. Ας ξεκινήσουμε τη σημερινή μας συνεδρίαση, την πρωινή συνεδρίαση. Την ημερήσια διάταξη φαντάζομαι την έχετε. Θα μου τη δώσει τώρα η γραμματεία. El primer punto del orden del día hace referencia al sistema común. Το πρώτο σημείο της ημερησίας διατάξεως αναφέρεται στο ΦΠΑ. Ο κύριος Κάσακ είναι ο εισηγητής, είναι στο δρανό του, του δίδω το λόγο. Thank you, Mr. Chairman, and good morning to, all my colleagues. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ναι, πράγματι. Αυτή είναι μια οδηγία η οποία τώρα έχει σωματωθεί στην υγεία και δεν χρειάζεται, νομίζω, να παρουσιαστεί γιατί πρόκειται για απλούστευση και εναρμόνιση των κανόνων για το ΦΠΑ. Έχει δοθεί στο κράτη-μέλη αυτή η πρόταση για την απλούστευση των κανόνων μέσα στα πλαίσια ιδίως των κανόνων που ισχύουν για την αποστολή των τιμολογίων. Ο στόχος είναι να απλουστευτεί η νομοθεσία και οι διοικητικές διαδικασίες στον τομέα του ΦΠΑ. Δεύτερον, να αρθούν τα νομικά εμπόδια της εσωτερικής αγοράς για τα τιμολόγια ΦΠΑ. Τρίτον, να απλουστευτεί η ενημέρωση των υποχρεώσεων ε, που θα μειώσει το διοικητικό κόστος και τέλος να εθαριθούν οι, οι να αναλάβουν το κόστος για την απλούστευση και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα των τεχνολογίων αυτών. Η Κομισιόν ίση μια σειρά κανόνων εναρμονισμένων, μειώνοντας τις εναλλακτικέ ε, που είχαν τα κράτη-μέλη και προβλέποντας επίσης ε, ηλεκτρονικά θυμολόγια με τους ίδιους όρους όπως τα επιχάρτου. Ε, αναφέρομαστε εδώ στις απροστατευμένες διαδικασίες, ειδήσει για μικρά ποσά που ενδιαφέρουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και κανόνες που επιτρέπουν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να <clears throat> δίνουν τον ορισμό ΦΠΑ σε βάση ρευστού. Μειώνονται τα νομικά εμπόδια στη μεταβίβαση και αποθήκευση των ηλεκτρονικών τομολογίων. Επίσης προσπαθεί να καταπολεθεί η απάτη με πιο αυστηρούς κανόνες όσον αφορά την μείωση ΦΠΑ και τις συναλλαγές διακοινωτικά. Η Κομισιόν προτείνει να προσθεθούν οι κανόνες όσον αφορά το ενδοκοινωτικό εμπόριο και να καθορίσει μια ενιαία ημερομηνία κατά την οποία ε, θα πρέπει να επιβάλλεται ο φόρος αυτός δηλαδή επιτρέπουν το τιμολόγιο να αποσταλεί στις 15 του μηνός και να απομένει το κύριο έγγραφο που θα καθορίζει τις συναλλαγές αυτές ενδοκοινωνικά. οι κανόνες τροποποιούνται για να είναι σύμφωνοι μεταξύ τους σε όλους τους τομείς. Η πρόταση ε, αναφέρεται στο δικαίωμα α, απαλλαγής ή έκπτωσης ανάλογα εάν υπάρχει στα χέρια του δικαιούχου αυτό το τιμολόγιο. Μόνο τότε μπορεί να ασκήσει το δικαίωμά του για να εκπέσει ο φόρος. Υπάρχει κάποια αμφιβολία κατά πόσον αυτή τη στιγμή εφαρμόζονται οι κανόνες αυτοί σε κάποια κράτη-μέλη και αυτό οδηγεί σε μια σύγχυση για τις επιχειρήσεις. Ένα άτομο υπόχρεο σε φόρο που αγοράζει κάτι σε μια άλλη χώρα θα πρέπει να πληρεί τους κανόνες για τα τιμολόγια στο άλλο κράτος μέλος και αυτό είναι δύσκολο βέβαια για τη χώρα μέλος στην οποία αυτό το άτομο είναι εγκαταστημένο. Η λύση είναι να υπάρχουν μια σειρά εναρμονισμένων κανόνων για τις συναλλαγές από επιχείρηση σε επιχείρηση. Ούτως ώστε ο υπόχρεος φόρο να ξέρει ότι το τιμολόγιο του αυτό ισχύει σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταρχήν υπάρχει η πρόβλεψη για τον πλήρη φόρο για τις συναλλαγές αυτές από επιχείρηση σε επιχείρηση και κατόπιν η δυνατότητα του υποχρέου να ασκήσει το δικαίωμά του για έκπτωση του φόρου αυτού. Όσον αφορά το τιμολόγιο το πλήρη ΦΠΑ, υπάρχουν τρεις αλλαγές στα άρθρα 2 ε, 6 της οδηγίας ΦΠΑ. Το πρώτο είναι να αναφέρεται ο αριθμός ΦΠΑ του ε, πελάτη. Δεύτερον, η ημερομηνία που αναφέρεται πρέπει να είναι η ημερομηνία κατά την οποία ε, πρέπει να καταβληθεί ο φόρος. Και τρίτον, αναφέρεται το δικαίωμα του πελάτη από αυτή την ημερομηνία και μετά να ζητήσει την έκπτωση. Επίσης υπάρχει το θέμα της αντιστρόφου, του αντιστρόφου συστήματος εάν ε, η αγορά γίνεται σε ένα άλλο κράτος μέλος. Και αναφέρεται το, η επίσημη ισοτιμία στην οποία υπολογίζεται το, ο ΦΠΑ ε, ανάλογα με τη χώρα στην οποία έχουν λάβει ε, χώρα οι αγορές ή οι προσφορές υπηρεσιών. Και αυτή είναι η ισοτιμία που καθορίζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Η Κομισιόν προτείνει επίσης όπως σας είπα ε, τιμολόγια επιχάρτου και ηλεκτρονικά να τεθούν επίσης όρις. Αναφέρεται ε, η, επίσης η διάρκεια δια, ε, τήρησης των ε, τιμολογίων αυτών να είναι έξι χρόνια. Έξι χρόνια πρέπει να τηρούνται. Εγώ έχω γενικά μια θετική αντιμετώπιση της πρότασης, αλλά έχω και κάποιες παρατηρήσεις να κάνω όσον αφορά το πώς θα μειωθεί η αβεβαιότητα κατά πόσον το γεγονός το οποίο είναι υπόχρεος το φόρο θα εξετάζεται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση με τον ίδιο τρόπο. Η Κομισιόν αυτό λέει την ομιλότητα των οποίων πραγματικά οι υπηρεσίες αυτές ή τα αγαθά έχουν ε, δοθεί στον δικαιούχο. Από εκεί και πέρα. Ε, δεν θα έχουμε πια την αβεβαιότητα που οδηγεί σε στρεβλώσεις. Μία δυνατή λύση θα ήταν να συσχετιστεί αυτό το γεγονός ...στη στιγμή κατά την οποία το τιμολόγιο εκδίδεται. Γιατί λέμε ότι πρέπει να υπάρχει στα χέρια του δικαιούχου ένα έγκαιρο τιμολόγιο για να μπορέσει να ζητήσει έκπτωση. Αυτό θα οδηγήσει σε προβλήματα ίσως εάν κάποιες επιχειρήσεις παίρνουν οι αγαθά υπηρεσίες από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί οι χώρες, στις χώρες αυτές δεν γνωρίζουν τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. θα πρέπει να ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή δεν προβλέπονται τα τιμολόγια όταν εκπίπτουν τα αγαθά του φόρου και θα χρειαστούν πολύ ε, χρονοβόρες και ακριβές διαδικασίες για να μετατραπούν τα συστήματα των εν λόγω χωρών. Επίσης όταν η, το είναι σε άλλο νόμισμα από εκείνο της χώρας στην οποία ε, εκδίδεται υπάρχουν επίσης προβλήματα. Όσον αφορά την απέτηση που λέει για τις εγχώριες ε, προς ε, παροχές να υπάρχει ο αριθμός ΦΠΑ στο τιμολόγιο, αυτό θα οδηγούσε σε ε, συμπληρωματική επιβάρυνση, γιατί αυτή τη στιγμή πολλά κράτη-μέλη δεν ζητούν τον αριθμό ΦΠΑ του πελάτη. Επίσης, είναι σημαντικό κατά τη γνώμη μου η καλή λειτουργία του συστήματος αυτού να υποστηριχτεί συμπληρωματικά μέσα στο ενό συμπληρωματικού φορολογικού συστήματος ή άλλων δυνατοτήτων. Γι' αυτό χαιρετίζω τις προτάσεις της Κομισιόν σαν ένα θετικό βήμα για ε, νομική βεβαιότητα και διαφάνεια και για τους ε, πελάτες και για την διοίκηση και μια συμπληρωματική δυνατότητα καταπολέμησης της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ. Θα ήθελα να ακούσω τους κοιότες εισηγητές. Είχαμε ήδη κάποιες συναντήσεις μεταξύ μας, καθώς επίσης και με τους συναδέλφους στην Επιτροπή αυτή. Και ίσως θα μπορούσαμε να έχουμε μια συζήτηση βάσει των προτάσεων που σας υπέβαλα και όταν προετοιμάσω το σχέδιο γνωμοδότησής μου θα μπορούσαμε να συζητήσουμε περαιτέρω. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Um, α, μία τελευταία παρατήρηση που την ξέχασα, Πρόεδρε. Συγγνώμη, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι η παρουσία μου του πρώτου σχεδίου θα γίνει σε 11, Μαρτίου, σε 11 Ιανουαρίου και 19 Ιανουαρίου θα είναι η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών. Ευχαριστώ. Σας διέκοψα για να δώσω μία πληροφορία, αλλά η γραμματεία με αντικατέστηση επαξίως. Ισκιώδης τώρα με πρώτο τον κύριο Τάλερ. Σα Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Σιγητά, αγαπητοί συνάδελφοι, γνωρίζουμε όλοι τη σημασία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την οικονομική ανάπτυξη και θα πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε το επιχειρησιακό περιβάλλον τους ώστε να υπάρχουν περισσότερες επιτυχίες, ιδέες και αγαθά. Συνήθως ε, οι επιχειρήσεις αυτές θεωρούν ότι τα διοικητικά εμπόδια είναι το κύριο ε, μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουν. Ένα κοινό σύστημα στον τομέα του φόρου προστασμένης αξίας όσον αφορά την τιμολόγηση είναι βέβαια καλόδεκτο. δεκτό. Από την άλλη μεριά όμως ε, δίνεται εντύπωση ότι ασχολούμεθα με μάλλον τεχνικά και όχι με πολιτικά θέματα. Αλλά θα πρέπει κανένας να παραδεχθεί ότι οι επιπτώσεις των ε, αλλαγών αυτών θα είναι σημαντικές. Η πρόθεση και χρήση των νέων τεχνολογιών και αναφέρομαι εδώ στα ηλεκτρονικά τιμολόγιας μειώνουν την γραφειοκρατία, την επιβάρυνση των επιχειρήσεων και αυτό θα δώσει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε άλλες επιχειρήσεις την ευκαιρία να μειώσουν το κόστος τους και να κερδίσουν ανταγωνιστικότητα. Απ' την άλλη μεριά, η χρήση των ε, ε τιμολογίων αυτών μέσα στα πλαίσια της οδηγίας ΦΠΑ μειώνονταν στις διαφορές μεταξύ των ηλεκτρονικών ε, ε, και των επιχάρτου τιμολογίων θα καταστήσουν τις φορολογικές αρχές πιο αποτελεσματικές. Πιο αποτελεσματικές για να αντιμετωπίσουν την πραγματική φορολογική απάτη και να μπορέσουν επίσης να μειώσουν το λειτουργικό τους κόστος. Παρόλο που γενικά συμφωνούμε με τις προτιμονόμενες τροπολογίες, παραμένουν κάποιες ερωτήσεις. Παραδείγματο χάρη η αποδίκευση των στοιχείων αυτών των τιμολογίων ή το όριο του ποσού για τις απλουστευμένες διαδικασίες θα πρέπει να αυξηθεί. Ως και ο δεσηγητής προσβλέπω να βρεθούν οι λύσεις για αυτά και άλλα παρόμοια ερωτήματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ κυρία Τάλερ. Παρακαλώ, πριν δώσω το λόγο στην Κομισιόν υπάρχει κάποια παρέμβαση. Όχι. Δεν ζητεί κανείς το λόγο. Οπότε τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Thank Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Σκάζα και τον σκιώδη συγγητή για την υποστήριξή τους. Σφαιρική υποστήριξη δική μα πρωτοβουλία από ό,τι κατάλαβα. Αυτή τη στιγμή δεν θα ήθελα παρά να τονίσω ότι η πρόταση αυτή είναι μια σημαντική πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με στόχο την μείωση του διοικητικού κόστους των επιχειρήσεων, προώθηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αύξηση όπως ακούσαμε την χρήση των ηλεκτρονικών τιμολογίων και επίσης ενίσχυση των κρατών μελών για να αντιμετωπίσουν την απάτη στον τομέα του ΦΠΑ. Είναι τμήμα δηλαδή μιας ευρύτερη στρατηγικής της Κομισιόν. Αξίζει επίση να σημειωθεί ότι το τμήμα που αφορά την ε, τα ηλεκτρονικά τιμολόγια, όπως αναφέρθηκε ιδίω και από την ενότατη ομάδα για τη μείωση του διοικητικού άχθους, που διοικήθηκε από τον κύριο Παρόζο και τις οποίες εδρεύει ο ο Σέβερ, την χάνει έντονης υποστήριξης και από την επιχειρησιακή κοινότητα. Η πρόταση αυτή λοιπόν συμπεριλαμβάνει πολλά τεχνικά στοιχεία, παρόλα αυτά τα ηλεκτρονικά ε, τιμολόγια είναι ένα σημαντικό στοιχείο και πολιτικά. Και χαίρομαι για την υποστήριξη που εκφράστηκε ήδη αυτή τη στιγμή από τον εισηγητή και τον σκιώδη εισηγητή. Σημειώνω τα διάφορα σχόλια που έγιναν για τεχνικό επίπεδο όσον αφορά του κανόνες που χρησιμοποιούν τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τις ισοτιμίες των νομισμάτων, την υποχρέωση των ε, πελατών να δίνουν τον αριθμό τους ΦΠΑ, το θέμα της διάρκειας αποθήκευσης των στοιχείων. Είμαι σίγουρο ότι θα μπορέσουμε μελλοντικά να επανέλθουμε σε αυτά τα πιο τεχνικά στοιχεία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κάζα για να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα βεβαίως να ευχαριστήσω τον Σκιώδη εισηγητή και τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο βασικός στόχος της νέας προτάσεως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να βοηθήσει τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις με την μείωση του διοικητικού άχθους να τις καταστήσει πλέον αποτελεσματικές και βεβαίως επίσης να καταπολεμήσει την φορολογική απάτη που ανέρχεται σε ύψος εκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται λοιπόν για μία πρόταση που θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις μας. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι για το σεβασμό και την ε, συμμόρφωση με αυτή την πρόταση θα πρέπει να επιβάλλουμε περισσότερα κανονιστικά μέτρα. Μέχρι την Ολομέλεια θα πρέπει να εξεύρουμε λοιπόν μια ισορροπία μεταξύ αυτού που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αυτού που εμείς θα επιθυμούσαμε ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και βεβαίως ε, να ικανοποιήσουμε και τα θεμητά αιτήματα του κλάδου τον, μέχρι τον Ιανουάριο θα, έχω, θα θέσω στη διάθεσή σας το πρώτο σχέδιο εκθέσεως το οποίο ε, θα συζητήσουμε και ελπίζω ότι έτσι θα μπορέσουμε να συμφωνήσουμε. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Έχει ανακοινωθεί το πρόγραμμα 8 Δεκεμβρίου είναι η καταληκτική προθεσμία για τροπολογίες. ¿Sabe Ε, δυστυχώς εδώ έχω κάποιο πρόβλημα. Κύριε Κάζα, ξέρετε το χρονοδιάγραμμα. Ναι, Πρόεδρε. 11 Ιανουαρίου θα παρουσιαστεί το σχέδιο έκθεσης. 19 Ιανουαρίου καταληκτή προθεσμία για τροπολογία που θα συζητηθούν 23 ε, Φεβρουαρίου και η ψηφοφορία 17 Μαρτίου στην Επιτροπή και ολομέλεια κάποια στιγμή αργότερα. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ για την πολύτιμη βοήθειά σας. Εδώ τα χάσαμε κάπως μέσα στη χαρτούρα που είχαμε. Τέλος πάντων. Συνέπειες της οικονομικής και δημοσιονομικής κρίσης στις αναπτυσσόμενες χώρες. Ο κύριος Κλούτε είναι ο εισηγητής. Έχετε το λόγο. Καλημέρα σας και ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς, κοιτάξτε, είμαστε σχολιαστές ε, στην έκθεση, γιατί η έκθεση ε, είναι στις ε, αρμοδιότητες Επιτροπής Ανάπτυξης. Ως εκ τούτου, απλά εγώ εκλήθη να τοποθετηθώ σύντομα ε, όσον αφορά την έκθεση αυτή τη επιτροπή Ανάπτυξης, δεν ξέρω ποια είναι η εξέλιξή τη. Η Επιτροπή Ανάπτυξης έθεσε το θέμα αυτό στην ημερήσια διάταξη λόγω του γεγονότο ότι η οικονομική κρίση έχει βέβαια επιπτώσει στις αναπτυσσόμενες χώρες. Και στις αναπτυσσόμενες χώρες αυξάνεται η ανεργία, διαπιστώνονται ε, αρνητικέ επιπτώσει στις εμπορικέ συναλλαγές και επίση προκύπτει το φαινόμενο πάρα πολύ εργαζόμενοι στις αναπτυγμένες χώρες ε, να ε, προσπαθούν να βοηθήσουν τις ε, πατρίδες τους με εμβάσματα αλλά και εκεί διαπιστώνεται σημαντική μείωση. Άρα δηλαδή βλέπουμε ότι υπάρχουν ουσιαστικές επιπτώσεις της ε, χρηματοπιστωτικής κρίσης και στις αναπτυσσόμενες χώρες. Και για τον λόγο αυτό η Επιτροπή Ανάπτυξης θέλησε να καταρτήσει αυτή, να συντάξει αυτή την έκθεση. Εγώ μία σελίδα είναι η δική μου έκθεση. Οι γνωμοδοτήσεις είναι αρκετά σύντομες. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες. Απλά θα ήθελα να σας πω ποια είναι τα κριτήρια τα οποία με οδήγησαν στο να ε, διατυπώσω αυτήν την την πρότασή μου. Νομίζω όλοι συμφωνούμε ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες δεν είναι οι κύριοι υπέτη αυτής της κρίσης, είναι θύματα της κρίσης αυτής. Γι' Ε, γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να δούμε ε, τι ακριβώς θα κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις χώρες αυτές. Εδώ θα πρέπει να ισχύει η αρχή της υπετιότητας και με βάση αυτή την αρχή να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα. Με άλλα λόγια δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση, τουλάχιστον αυτή είναι η δική μου άποψη και πρόταση, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι υποχρεωμένη να επιδείξει κάποια αλληλεγγύη απέναντι στις χώρες εκείνες οι οποίες χωρίς να φταίνε αντιμετωπίζουν μια κατάσταση που καλούνται να την διαχειριστούν αποτελεσματικά. Οι στόχοι και οι πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να στοχεύουν έχοντας κατά νου ότι υπάρχουν χώρες που έχουν σημειώσει πρόοδο, αναπτυσσόμενες χώρες που παρουσίασαν οικονομική ανάπτυξη. Γι' αυτό λοιπόν οι πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους ότι αυτή η πρόοδος πρέπει να σταθεροποιηθεί, οι χώρες αυτές ε, δεν πρέπει να υποστούν οπισθοχώρηση ε, και αυτό που θέλω επίση να πω είναι ότι να ληφθούν ιδιαίτερα υπόψη οι λιγότερο αναπτυγμένες χώρες. Αυτές με τα μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να στηριχθούν, να σταθεροποιηθούν έτσι ώστε να μην διολυστήσουν σε ακόμα πιο βαθιά κρίση. Αυτά νομίζω ότι είναι τα βασικά στοιχεία της ε, έκθεσή και τα βασικά στοιχεία που θα πρέπει να καθορίσουν τι πράξεις τη Ευρωπαϊκής Ένωση. Επιτρέψτε μου σύντομα να αναφερθώ στο σημείο υπαριθμών 5. Τη Δευτέρα είχαμε μία ανταλλαγή απόψεων σε ανοιχτή συνεδρίαση συντονιστών με τον κύριο Μάιστατ, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της ΕΙΜΠ, της ε, Τράπεζα, Εγώ ε, στο σημείο υπαριθμό 5 αναφέρομαι στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Ο κύριος Μάιστατ ε, και αυτός ε, τοποθετήθηκε. Εγώ λέω ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων δεν πρέπει να καταφεύγει σε φορολογικούς ε, παραδείσους. Ο κ. Μάιστερ τοποθετηκε και αυτός και γι' αυτό έχει κατεθεί μια τροπολογία που λαμβάνει αυτά που είπε ο πρόεδρος ε, της ΕΤΕ που είπε ότι η ΕΤΕ πράγματι θα λάβει υπόψη σε αυτές τις εξελίξεις. Υπάρχει λοιπόν μια συγκεκριμένη πρόταση που σας καλώ να την υποστηρίξετε κατά άλλα. Θέλω να σας πω ότι ο κύριος Μάιστατ χαιρέτησε ανεπιφύλακτα το γεγονός ότι σε αυτό το σχέδιο ε, συμπεριλαμβάνουμε τα κριτήρια της Διεθνούς ε, Οργάνωσης Εργασίας και η Κομισιόν έχει τοποθετηθεί. Γίνεται λόγος για μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας που πρέπει να λάβουν χώρα κυρίως αναπτυσσόμενες χώρες οι οποίες χρειάζονται την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ συνειδητά τα αναφέρω αυτά. Από πλευρά ε, Διεθνού Οργάνωση Εργασία υπάρχει ένα πρόγραμμα το οποίο ξεκίνησε ε, πριν από 10 χρόνια. Ε, φέρει την επικεφαλίδα Decent Work. Κατ' ουσίαν εδώ πρόκειται για αξιοπρεπεί συνθήκε εργασία και νομίζω ότι το πρόγραμμα αυτό θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την χορήγηση κονδυλίων. Θα πρέπει μάλιστα να είναι το καθοριστικό κριτήριο. Και αυτό το υποστήριξε και ο κ. Μάιστατ. Ήθελα και εγώ να σα το αναφέρω σήμερα εδώ. Δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Κατά τα άλλα, προ τα παρόν, ε, ολοκληρώνω και θα δούμε. Περιμένω τι παιδικέ παρατηρήσει. Ο κύριος Λάγκεν έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ θα ήθελα να σας επισημάνω ότι η ανακοίνωση της Κομισιόν της ε, είναι της 8ης Απριλίου του 2009, δηλαδή ε, παρουσιάστηκε αμέσως μετά την πρόταση του πρώτου πακέτου της δέσμης μέτρων για την αντιμετώπιση της χρηματοπιστωτικής κρίσης. Αυτή είναι η πρώτη μου παρατήρηση. Οι αναπτυσσόμενες χώρες βεβαίως και δεν προκάλεσαν τη χρηματοπιστωτική κρίση, βεβαίως και υποφέρουν από αυτή, δεν υπάρχει αμφιβολία από αυτού, αλλά το πιο κρίσιμο είναι πώς θα ξεπεραστεί η κρίση αυτή. Τούτο λοιπόν αναφέρεται και πρέπει να αναφέρεται ε, στην έκθεση του κυρίου Κλούτε, στη συμπληρωματική του έκθεση. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι το εξή. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι έχοντας μπροστά μας αυτή την ε, εκτεταμένη τοποθέτηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχουμε ουσιαστικά στα χέρια μας ε, πάρα πολλές απόψεις αλλά στη τελική ανάλυση αυτό που προτείνει η Κομισιόν είναι πάρα πολύ μετριοπαθές. Αναφέρονται πάρα πολλά σημεία αλλά τα μέτρα που προτείνει κατ' ουσίαν τι λένε. Λένε μόνο ότι τα κονδύλια που υπάρχουν να ε, εκταμιευθούν νωρίτερα ή τα ήδη υπάρχοντα προγράμματα να αυξηθούν. Αυτό δεν είναι καμιά ιδιαίτερη πολιτική, είναι απλά κάποια ενίσχυση των μέτρων που ήδη έχουν ληφθεί. Κατόπιν, αυτό που θέλω να πω και δεν μου αρέσει ιδιαίτερα είναι ότι ε, εστιάζεται η έκθεση σε δημοσιονομική βοήθεια. Όλοι μας γνωρίζουμε ότι πρέπει να τεθεί το θέμα της διαφθοράς και στις αναπτυσσόμενες χώρες ε, πρέπει να ισχύουν συνθήκες πλαίσιο για να τους ε, χορηγηθούν τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα τύχουν σωστής και αποτελεσματικής χρήσης. Εγώ λοιπόν δεν χαίρομαι πάρα πολύ για το γεγονός ότι άλλοι παράγοντες όπως η Διεθνής Εμπορική εμπορική πολιτική ή τα διαρθρωτικά προβλήματα των αψωμένων χωρών, ναι μεν θίγονται αλλά δεν προτείνονται συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπιση της κρίσης. Ως εκ τούτου, οι προτάσεις της Κομισιόν, κατά τη δική μου τουλάχιστον άποψη, παραμένουν προσκολλημένες ε, στα στερεότυπα, ότι δηλαδή λύνονται τα προβλήματα μόνο αυξάνοντας τα κονδύλια. Δεύτερον, η ε, αξιολόγηση των μέτρων ως προς την αποτελεσματικότητά τους, κατά πόσο αυτά συμβάλλουν στην ανάπτυξη και στην μείωση της ένδυας, αυτό το στοιχείο δεν αναφέρεται στην έκθεση της Κομισιόν. Τα δομικά, τα διαρθρωτικά προβλήματα των αναπτυσσομένων χωρών, όπως και τα συμφέροντα ε, των ε, δωρητών, αυτά ε, δεν είναι συντονισμένα και ως εκ τούτου δεν αντιμετωπίζονται συγκεκριμένα και δεν αποδίδουν ιδιαίτερα. Αν θέλετε με άλλα λόγια, είναι ο απολογισμός καλή είναι η διάγνωση, όμως η θεραπεία κατά τη γνώμη μου ε, δεν είναι αποτελεσματική και ως εκ τούτου η δική μας η έκθεση ε, θα πρέπει να καθιστά σαφή αυτή την άποψη, κάτι που δεν καθιστά σαφές η έκθεση του κυρίου Κλούτε. Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι θα πρέπει να αποδώσουμε ιδιαίτερη σημασία στην ε, ταχύτατη αντιμετώπιση της κρίσης, να καλέσουμε παράλληλα τα κράτη-μέλη να κάνουν και αυτά μία προσπάθεια, να μην ε, ε, πέφτουν σε ένα είδο ε, νοσταλγίας γιατί στη τελική ανάλυση για να του δοθούν κονδύλια πρέπει να πληρούνται και ορισμένε προϋποθέσεις. Ω εκ τούτου εγώ θα υποβάλω ε, τροπολογίες εκ μέρου της δικής μου πολιτικής ομάδας γιατί όσο ωραία και αν είναι η έκθεση λυπάμαι ε, όπως και όλες οι γνωμοδοτήσεις ε, υποφέρει καταρχήν από ότι είναι πολύ σύντομη και κατόπιν τούτου με τροπολογίες εμείς θέλουμε να συμπληρώσουμε αυτό το σχέδιο έκθεσης. Θα καταθέσουμε λοιπόν τροπολογίες οι οποίες θα καθιστούν σαφές ότι η διεθνοποίηση στο σύνολό της τελική ανάλυση περισσότερο ωφέλησε και δεν ζημίωσε τις αναπτυσσόμενες χώρες. Ναι, μεν θίγονται από τη χρηματοψηφική κρίση τα αναπτυσσόμενα κράτη, αλλά σε τελική ανάλυση η κρίση έπληξε περισσότερο τις ε, μεγάλες ε, χώρες και οι φτωχότερες χώρες παρόλα αυτά επιδεικνύουν ένα κάποιο ποσοστό ανάπτυξης. Παρότι θίγονται δεν είναι αλήθεια ότι η αναπτυξιακή πολιτική δεν έχει αποφέρει καρπούς. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Λάγκεν. Η κυρία Χούμπνερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Πρέπει να αποφύγουμε να δώσουμε την εντύπωση με την ανακοίνωση αυτή και με την αντίδρασή μας ότι η κρίση προέρχεται από το διεθνές ε, οικονομικό περιβάλλον και τις αναπτυγμένες χώρες. Γιατί αυτό θα έχει πολύ κακές συνέπειες στις αναπτυσσόμενες χώρες. Θα πρέπει να είμαστε απόλυτα σαφείς ότι θα πρέπει να έχουμε ρεαλιστική <clears throat> προσέγγιση να βελτιώσουμε την νομοθεσία και σε εθνικό και σε διεθνές επίπεδο, ούτως ώστε να αποφύγουμε προβλήματα που αφορούν που προέρχονται από τον προστατευτισμό ή τη, φορολογική, τη φοροδιαφυγή ή τη φορολογική απάτη. Και βεβαίως θα πρέπει να είμαστε αποτελεσματικοί και στο, διεθνή, στο διεθνές προσκήνιο. Υπάρχει συνένεση σε πολλές από αυτές τις χώρες, ε, εξαιρετικά ευάλωτη και εύθραυστη όμως, που τώρα λόγω της ε, κρίσεως μπορεί να καταρρεύσει. Γι' αυτό θα πρέπει να αναφέρουμε τα πράγματα ως έχουν, γιατί αλλιώς αν εθελοτυφλήσουμε οι αρνητικές συνέπειες στις αναπτυσσόμενες χώρες θα είναι τραγικές. Το δεύτερο μου σχόλιο το διεθνές ε, σύστημα θα πρέπει να προστατεύσει ε, τους ευάλωτους, ε, τα ευάλωτα κομμάτια του πληθυσμού, τις ευάλωτες χώρες. Αλλιώς αυτοί θα αποκλειστούν από την θετική πτυχή του συστήματος. Θα πρέπει λοιπόν να αναλάβουμε μια δέσμευση μια αποφασιστικότητα εναντί των ευάλωτων αναπτυσσομένων χωρών. Και το τρίτο, δεν λέμε τίποτα για τι αναπτυσσόμενες χώρε και τα χρηματοοικονομικά συστήματα σε αυτές τις χώρε θα πρέπει να αναφέρουμε πώς θέλουμε να είναι ο τομέας στις αναπτυσσόμενες χώρες. Στα πλαίσια της μεταρρύθμισης του παγκοσμίου δημοσιονομικού και χρηματοοικονομικού συστήματος, πριν την κρίση στην Ασία, λέγαμε στις αναπτυσσόμενες χώρες ότι το σύστημα του θα πρέπει να είναι σαν το δικό μας. Μετά την κρίση, σταδιακά αρχίσαμε να λέμε ότι εντάξει, ενδεχομένως ή σιγά σιγά σταδιακά θα πρέπει να είναι σαν τα δικά μας ε, τα συστήματά τους, σαν το δικό μας. Είναι θέμα αξιοπιστία λοιπόν. Η εικόνα που θέλουμε να περάσουμε στις αναπτυσσόμενες χώρες δεν είναι τόσο ε, μονοσήμαντη, δεν είναι τόσο σαφής. Είναι πιο πολύποκα τα πράγματα και μιλάμε για ένα μείγμα νομοθεσίας και κρατικής παρέμβασης. Αλλά να σιωπήσουμε δεν μπορούμε γιατί πρέπει οι αναψώμενες χώρες να ενσκύψουν από αυτών των θεμάτων αν θέλουν να αποφύγουν ε, τις μακροπρόθεσμες ε, παρενέργειες της κρίσεως. Αφήστε που και για μας αυτό θα είναι πιο επώδυνο, πιο δύσκολο. Τώρα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα θέματα αυτά, διότι όσο πιο πολύ καθυστερούμε, το πιο δύσκολο θα είναι να τα αντιμετωπίσουμε. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Τσικλούνα, Γκίκο και Περέιρα από τους οποίους ε, ζητώ μεγάλη συντομία. Ο κύριος Τσικλούνα. Ευχαριστώ. Ξέρω ότι η ανάπτυξη είναι πολύ πλοκό ζήτημα. Δεν μπορούμε όμως να αγνοήσουμε την εκπαίδευση και το εμπόριο. Δεν αναφέρεται η απασχόληση, η ανεργία, το ίδιο και η μετανάστευση, η παράνομη μετανάστευση αλλά και η μετανάστευση για λόγους εργασίας. Στη Μεσόγειο το πρόβλημα είναι οξύ και δαπανηρό. Όταν μιλάμε λοιπόν για βοήθεια προς τις αναπτυσσόμενες χώρες θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και το θέμα της μετανάστευσης. Για τη διαφθορά. Πιστεύω ότι θα πρέπει να το τονίσουμε περισσότερο το ζήτημα αυτό. Η χρηστή διαχείριση, η χρηστή διακυβέρνηση ή η έλλειψη αυτής είναι λόγος υπανάπτυξης και θα πρέπει να το πούμε. Και τέλος, για την παράγραφο 6. Δεν χωρά καμία αμφιβολία ότι αυτή είναι η ιδανική λύση. Όσο πιο ψηλά στοχεύουμε όμως, τόσο πιο δύσκολα είναι τα πράγματα. Θα πρέπει να είμαστε λιγότερο φιλόδοξοι, πιο προσγειωμένοι ούτω ώστε να μιλάμε για μεταρρυθμίσεις και αλλαγέ που στο ε, άμεσο μέλλον θα μπορέσουν να εφαρμοστούν. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Γκίγκο, παρακαλώ και εσείς σύντομα, όπω ο προλαλή σα. Συμφωνώ με όσα ελέγχθησαν. Δεν χρειάζεται να τα επαναλάβουμε. Νομίζω λοιπόν ότι όλη αυτή η μερίσια διάταξη περί συνοχής είναι πολύ σημαντική και είναι πολύ κοντά σε αυτά που είπε ο κ. Λάγκε. Και πιστεύω ότι θα πρέπει να το υπογραμμίσουμε αυτό όταν μιλάμε για εμπόριο ή για άλλες πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετανάστευση πρέπει να το τονίσουμε. Πέρα από αυτό θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι από ό,τι Πιστώσα. η έκθεση είναι σωστή. Εγώ συμφωνώ με αυτήν. Υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να προσθέσουμε. Αυτό που πρέπει να το πούμε με μεγαλύτερη σαφήνεια είναι το εξή. Αν δούμε ένα σημείο όπου πράγματι υπάρχει κάποια ευθύνη των ε, αναδυόμενων οικονομιών, εκεί είναι στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το παγκόσμιο νομισματικό οικονομικό σύστημα. Και εδώ υπάρχουν δύο πτυχές του νομίσματος. Από τη μια πλευρά έχουμε μεγάλο έλλειμμα των ΗΠΑ και από την άλλη υπάρχουν πλεονάσματα. Το θέμα λοιπόν ότι μια χώρα που είναι ε, φτωχή, που έχει προβλήματα σταθερότητας, το ε, προσπαθεί αυτή να βρει μια καλή ισοτιμία, αυτό είναι κατανοητό. Από την άλλη όμως η ανισορροπία είναι πάρα πολύ μεγάλη. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να επισημανθεί ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει ένα παγκόσμιο νομισματικό σύστημα που θα ε, καταπολεμά αυτά τα υπερβολικά ελλείμματα και τα υπερβολικά πλεονάσματα. Τέλος, και αυτό το λέω σε σχέση με αυτά που είπε ο συνάδελφός μου από την πατρίδα μου, ο κύριος Λάγκεν. Ε, νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να αποφύγουμε να ξαναρχίσουμε το ίδιο θέμα, ε, την ίδια διαμάχη κατά πόσον η παγκοσμιοποίηση είναι καλή ή όχι για τις αναπτυσσόμενες χώρες. Κοιτάξτε, η πραγματικότητα είναι πολύ πιο περίπλοκη. Στις ε, αναπτυσσόμενες χώρες υπάρχουν και νικητές και οι Το ίδιο ισχύει και για τις αναπτυγμένες. Αν δούμε παραδείγματο χάρη τις εξαγωγέ, έχουμε του ιτημένους και ε, στις αναπτυσσόμενες χώρες έχουμε αυτούς που έχασαν τη δυνατότητα να ζουν σε ένα υγιές περιβάλλον. Από την άλλη βέβαια υπάρχουν πολλές αναπτυσσόμενες οικονομίες που βελτιώθηκαν, ε, δημιουργήθηκε βιομηχανικός ε, κλάδος, έχουμε γυναίκες που εργάζονται, υπάρχουν και θετικές εξελίξεις. Ω εκ τούτου με τις τροπολογίες ε, που θα καταθέσετε μην πείτε μόνο ότι το ε, παγκόσμιο εμπόριο είναι καλό ή κακό. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Είναι πολύ πιο περίπλοκα. Ευχαριστούμε πολύ. Ε, κοιτάξτε, δεν θα αρχίσουμε φιλοσοφική συζήτηση. Κάθε πολιτική ομάδα μπορεί βεβαίως να καταθέσει τις δικές της τις τροπολογίες. Πριν δώσουμε το λόγο στον εισηγητή, θα ήθελα να δώσω το λόγο πρώτα στο σκιώδη εισηγητή. Θα ήθελα να πω ότι είναι πολύ θετική η πρόταση του εισηγητή μας ε, την οποία στις αδρές της ε, γραμμές ε, συμμερίζομαι απόλυτα. Θα ήθελα απλώς να συμπληρώσω επί κάποιων πτυχών για την οικονομική ανάλυση, τη μακροοικονομική συνεργασία, τα θέματα ισορροπίας, στεθερότητας, τα δημόσια οικονομικά και τη διεθνή φορολόγηση. Από πλευράς οικονομικής ανάλυσης είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι η διάσταση και η πολυπλοκότητα της κρίσεως ε, οφείλεται στο χάσμα μεταξύ της, ε, των χρηματοπιστωτικών και χρηματοοικονομικών αγορών και της πραγματικής οικονομίας. Στο Πίτσμπουργκ αυτό ελέγχθηκε ότι θα πρέπει να μειωθεί το χάσμα και για να μειωθεί το χάσμα η ανάπτυξη μπορεί να είναι μια πολύ σημαντική κινητήρια δύναμη από τρεις λόγους ε, προέκυψε η κρίση. Οι πιστώσεις, οι χρηματοοικονομικές αγορές και η παγκοσμιοποίηση Αυτή είναι οι τρεις διάβλοι και από αυτών των τριών διάβλων ε, θα πρέπει να κάνουμε προτάσεις και σε διεθνές επίπεδο επ' αυτού θα επιμείνουμε. Μακροοικονομική συνεργασία G20 ΟΗΕ και μεταρρύθμιση των διεθνών δημοσιονομικών φορέων. Είναι θέμα και της καλύτερης επίσης λειτουργίας του διεθνούς εμπορικού συστήματος. Και βεβαίως ε, θα πρέπει να έχουμε ε, πολυμερείς ε, κανόνες στον τομέα των εμπορικών συναλλαγών αλλά και τον χρηματοοικονομικό μετά, στην μετά Bretton Woods εποχή σε συνεργασία με τις ΗΠΑ και τις αναψώμενες χώρες των ΟΗΕ ε, και θα πρέπει να επιμείνουμε επί δύο θεμάτων που είναι επικαιρότητα. Το G20 μίλησε για μεταρρύθμιση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που θα πρέπει να αξιολογήσει ε, το άχθος ε, που προκύπτει από το φορολογικό άχθος που ε, προκύπτει ε, από την σημερινή κατάσταση. Όχι μόνο για τις αναπτυγμένες αλλά και για τις αναπτυσσόμενες χώρες. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο λοιπόν θα πρέπει να ασχοληθεί με αυτό το θέμα. Και δεύτερον, αφορά τον φόρο για τις διεθνείς χρηματοοικονομικές συναλλαγές. Θα πρέπει να το συζητήσουμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να δούμε ποιοι είναι οι στόχοι, δηλαδή οι στόχοι της χιλιετίας, η κάλυψη των διεθνών ανισορροπιών και η συνεισφορά μας στην αηφόρο ανάπτυξη. Ευχαριστώ κύριε Σάντσεθ Πρεσέδο. Ελπίζω ότι ο εισηγητής κύριος Κλούτε σημείωσε τα λεγόμενα όλων των συναδέρφων παρατηρήσεις που θα μετασχηματιστούν σε τροπολογίες που θα έχουμε τη δυνατότητα να μελετήσουμε εφόσον υποβληθούν μέχρι την καταληκτική προθεσμία που είναι η 8η Δεκεμβρίου. Κύριε Λάγκεν, εγώ προεδρεύω. Θα σας δώσω το λόγο όταν το θεωρήσω σκόπιμο. Λοιπόν, 11 Ιανουαρίου οι τροπολογίες και η ψηφοφορία αυτών και 25 Ιανουαρίου του 2010 στην Επιτροπή. Τώρα έχετε το λόγο κύριε Λάγκεν. Κοιτάξτε, εγώ προτείνω την ε, επόμενη εβδομάδα να μας τη δώσετε και να μπορούμε να καταθέσουμε τις τροπολογίες μέχρι τις 10. Το έγγραφο αυτό ε, γκρίθηκε τον Απρίλιο με την ε, έγκριση και της κυρίας Χούπνερ ε, πρώην Επιτρόπου. Γι' αυτό λοιπόν αφήστε μας λίγο χρόνο, μας βάλει το μαχαίρι στο λαιμό και να πρέπει να καταθέσουμε τις τροπολογίες μέσα σε τρεις ημέρες. Ο εισηγητής συμφωνεί. Εντάξει, συμφωνεί. Μπράβο κύριε Λάγκεν, έβγε, πέρασε η πρότασή σας, κερδίσατε. Λοιπόν, τέλειωσε αυτό το σημείο της ημερησίας διατάξεως. Ε, παραχωρώ την Προεδρία στον κύριο Τσικλούνα εφόσον εγώ ίδιο θα πρέπει να παρουσιάσω την ε, έκθεση αυτή. Μείνετε στέση σας κύριε Τσικλούνα, δεν χρειάζεται να έρθετε εδώ. Θα γίνει εικονική μεταφορά του προεδρικού θόκου. Η δεύτερη λοιπόν γνωμοδότηση, της οποίας εγώ, ε, έκθεση της οποίας εγώ είμαι εισηγητής, είναι η διοικητική συνεργασία και η καταπολέμηση της απάτης. Αναδιατύπωση των ε, σχετικών οδηγιών. Μιλάμε για 60 με 100 δις το χρόνο που χάνουμε. Τώρα, η, έκθεση προτείνει δύο βασικά στοιχεία. Ένα οπλοστάσιο περισσότερων μέτρων στη διάθεση των κρατών μελών για την καταπολέμηση της απάτης και δεύτερο, μία νομική βάση για τη δημιουργία μιας πιο της δομής εις αφορά τη συνεργασία για την καταπολέμηση της απάτης. Υπάρχουν προηγούμενα και προέρχονται από διάφορους φορείς. Εδώ, στο Κοινοβούλιο, στην προηγούμενη θητεία, εγκρίναμε ε, την έκθεση της κυρίας Μπάουτ, Προέδρου της Επιτροπής, που σωστά είχε πει ότι ναι μεν η καταπολέμηση της απάτης είναι θέμα εθνικό και εθνικής κυριαρχίας αλλά που κανείς δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μόνος του. Όπερ σημαίνει διεθνή συνεργασία. Έχουμε και το ελεγκτικό συνέδριο που το 2007 σε γνωμοδοσή του ζητεί τρία τεινά. Πιο πολύ συνεργασία, πιο πολύ επικοινωνία και βελτίωση των βάσεων δεδομένων που, ε, στις βασιζόμαστε ε, για την ε, φορολογία. Στις αρχές του 2009 η Κομισιόν έκανε μια ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία επισημαίνει κάποια ελλείμματα εις ό,τι αφορά, ελλείψεις ό,τι αφορά την εφαρμογή του κανονισμού. Ας πούμε, οι καθυστερημένες ανταποκρίσεις σε αιτήματα άλλων κρατών μέλων έφτασαν σε επίπεδο απολύτως απαράδεκτο. Ε, επίσης ότι θα πρέπει να βελτιωθεί η αυτόματη πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων για την συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών που εμπλέκονται σε διαμεθοριακές συναλλαγές ότι είναι απαραίτητο να υπάρξει ένα σύστημα μέσω του οποίου το ένα κράτος μέλος να ενημερώνει το άλλο να βελτιωθεί η αξιοπιστία των ε, αριθμών φυρολογικού μητρώου και τέταρτο υπογραμμίζει ότι οι υπάλληλοι που κάνουν έρευνα σε άλλο κράτος μέλος να μην θεωρούνται ε, ότι παρεμβαίνουν στα χωράφια της εθνικής κυριαρχίας και ότι να υπάρχει συνεργασία και υποστήριξη από το κράτος που τους φιλοξενεί. Η πρόταση λοιπόν αυτή παρουσιάζει κάποια στιγμή τα οποία θα ήθελα να σχολιάσω. Πρώτον, ο στόχο έχει η πρόταση της Κομισιόν να οδηγήσει σε μεγαλύτερη κινητοποίηση των κρατών μελών ό,τι αφορά την διοικητική συνεργασία για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, στη συγκεκριμένη περίπτωση για το ΦΠΑ. Ένας από τους στόχους του κανονισμού είναι η διευκόλυνση του υπολογισμού του φόρου και άρα και της εφαρμογής του. Ιδιαίτερα στις ενδοκινοτικές συναλλαγές. Μεγαλύτερη λοιπόν ευθύνη ε, για τα κράτη-μέλη και περισσότερες πληροφορίες. Ο κανονισμός επίσης αναφέρει ως υποχρέωση την συλλογή και διαβίβαση των πληροφοριών που είναι χρήσιμες για άλλο κράτος μέλος. Και αυτό θεωρείται ένα κατάλληλο μέσο που περνάει όμως από τη δημιουργία μιας βάσης, ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων που κατά την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μπορεί να διευκολύνει και να προωθήσει τη διοικητική συνεργασία. Τρίτη πτυχή του κανονισμού. Αύξηση της χρησιμότητας της πληροφορίας που διαβιβάζεται. Κοινοί κανόνες, κοινά πρότυπα σε ό,τι αφορά αυτές τις πληροφορίες. Με ιδιαίτερη προσοχή σε αυτές που αναφέρονται στην συλλογή και διαβίβαση δεδομένων σχετικά με τον αριθμό φορολογικού μητρώου. Και τέταρτο, κοινή αποθήκευση των δεδομένων για πέντε χρόνια στη βάση δεδομένων. Και πέμπτο, διοικητική έρευνα σχετικά με την λεγόμενη αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών με δύο καινοτόμες υποχρεώσεις την λεγόμενη αυθόρμα, αυθόρμητη ανταλλαγή απόψεων και την ανταλλαγή, όχι απόψεων, πληροφοριών και δεύτερον ανταλλαγή πληροφοριών μετά από αίτημα και βεβαίω θα πρέπει να βασιστούμε στην κατάλληλη νομική βάση, ούτως ώστε να δημιουργήσουμε αυτή την κοινή διοικητική δομή, την λεγόμενη Eurofisk, που είναι ε, ουσιαστικά η μετάφραση με νομικούς όρους της ε, Europanet που υπάρχει ήδη ως ε, βάση του συστήματος. ο Ευρωπαίος επόπτης ε, και ε, έστειλε επιστολή στον πρόεδρο Μπούζεκ αναφέροντας ότι ορισμένες πτυχές θα μπορούσαν να βελτιωθούν ούτως ώστε να γίνουν σεβαστοί οι ευρωπαϊκοί κανόνες για την προστασία των δεδομένων. Ορισμένα ερωτήματα προς την Κομισιόν. η αεροφυσική είναι κοινοτική ή διακυβερνητική δομή. Ποιο είναι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα πλαίσια της λειτουργίας του δικτύου Eurofisc εφόσον υπάρχουν μικτές αρμοδιότητες. για την ορθή λειτουργία της διοικητικής συνεργασίας και για την κάλυψη των ελλείψεων που η ίδια η Κομισιόν έχει εντοπίσει. Πώς θεωρείτε, Κομισιόν, ότι μπορούμε να αναλάβουμε μια πραγματική κοινή ευθύνη τα κράτη-μέλη και να έχουμε μια σωστή αναπτυξιακή ε, συνεργασία με τις αναπτυσσόμενες χώρες. Και τελευταίο, καλό θα ήταν η Κομισιόν να μας ενημερώσει για το πού βρίσκεται η πρόταση αυτή σε σχέση με την συνεργασία με το Συμβούλιο. Αυτά από μένα. Ποιος ζήτησε το λόγο. Πήγαινα να πω ότι είναι, ο πρόεδρος είναι ο Τσικλούνα. Δεν μπορώ εγώ να προεδρεύσω. Οπότε δεν μπορώ να δώσω το λόγο σε κανένα. Ε, ωραία, αναλαμβάνω εγώ. Αναλαμβάνω εγώ ούτως ή άλλως για το επόμενο θέμα, οπότε θα αναλάβω από τώρα. Κύριε Στρέτσεκ. Ε, Καλημέρα σας ε, κύριε Πρόεδρε. Προσβλέπω στην συνεργασία με τον κύριο Καρσία Μαγκάλο για την έκθεση αυτή, γιατί τον γνωρίζω σαν ένα πολύ σεβαστό και σόφρον μέλος της Επιτροπής αυτής. Θα ήθελα να τον ευχαριστήσω για την εισαγωγή που καταδείχνει ότι θα χρησιμοποιήσει μία λογική και σταθμισμένη προσέγγιση στο πρόβλημα αυτό. Ε, χαίρομαι ιδιαίτερα με τα όσα μας είπατε εισαγωγικά. Συνεννοούμαστε νομίζω. Για το ΦΠΑ θα αναφέρω αυτό που είπα και χθε. Ε, δεν ήταν βέβαια ιδανικό εάν μπορούσαμε να έχουμε μόνο ένα ε, ποσοστό ΦΠΑ χωρίς όλες αυτές τις εκατοντάδες εξαιρέσεων στα διάφορα κράτη-μέλη. Γιατί ακριβώς αυτές οι εξαιρέσεις είναι εκείνες ε, που οδηγούν στην φοροδιαφυγή και στην απάτη. Συμφωνώντας με τον κύριο Γκαρσία Μαγκάλιο, νομίζω ότι αυτό όμως δεν πρόκειται ποτέ να επιτευχθεί. Αυτό που θέλετε ότι είναι, θεωρώ ότι είναι κάπως λεπτό θέμα είναι η επιλογή της ε, ανταλλαγής πληροφοριών. Στο έγγραφο, και αυτό το ανέφερε και ο κ. Καρσία Μαγκάλο, γίνεται αναφορά στην αυτόματη ανταλλαγή απόψεων ή πληροφοριών. Φοβούμε ότι η αυτόματη αυτή ανταλλαγή απόψεων θα στρεβλώσει τον ανταγωνισμό γιατί αυτόματα η ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά τον ε, φόρο εργασιών των επιχειρήσεων μπορεί να οδηγήσει σε καταχρήσεις. Εμείς δεν θα ήμασταν κατά της ε, εγκαθίδρυσης ενός συστήματος στα πλαίσια του οποίου τα μεμονωμένα κράτη-μέλη θα συλλέξουν πληροφορίες, θα ανταλλάξουν αμοιβαία τις πληροφορίες τους και ούτω καθεξής. Απ' την άλλη μεριά, εμείς υποστηρίζουμε ένα σύστημα μινιμαλιστικό όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών, κυρίως για τα ευαίσθητα τμήματα της πληροφορίας αυτές όπως ε, άφησε να ενωθεί και ο κ. Γκαρσία Μαγκάλιο, ότι τα συστήματα ηλεκτρονικής ανταλλαγής απόψεων και πληροφοριών είναι πολύ επικίνδυνα και υπάρχουν διάφοροι, ξέρετε, που μπορούν να μπουν κάποιοι hackers στα συστήματα άμυνας των ΗΠΑ της Αμερικής. Ε, πόσα παραπάνω σε αυτά τα θέματα που είναι λεπτά όσον αφορά τη φορολογία, όσον αφορά μια επιχείρηση κλπ. Εμείς θα φοβόμαστε ότι θα υπάρχει πραγματικά διαρροή πληροφορών, αλλά ε, φαντάζομαι ότι κάπου θα μπορούσαμε να συνεννοηθούμε. Το ευάλωτο των ηλεκτρονικών συστημάτων ανταλλαγή ε, προβλημάτων είναι το ένα. Η Eurofisc επίσης θα πρέπει να αναφερθεί εδώ. Έχω και εγώ κάποιο πρόβλημα με τον καθορισμό του Eurofisc. Δηλαδή, πώς θα λειτουργήσει, ποια μορφή θα πρέπει να έχει. Θα πρέπει να είναι υπεράνω των εθνικών ε, νομοθεσιών και της εθνικής εκάστοτε δικαιοσύνης. Εγώ προσβλέπω πάντως να ακούσω περαιτέρω τη σύντηση που θα εξελιχθεί. Ευχαριστώ. Η κυρία Κιούρη έχει το λόγο από το ΕΛΚ. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να χαιρετήσω την πρόταση αυτή και να πω ότι θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε μία νομική βάση για τη λειτουργία του Eurofisc. Αυτό ήταν ένα μεγάλο εμπόδιο και παρεμπόδιζε τη συνεργασία των ε, αρχών. Όσον αφορά την αποκάλυψη των απατών ε, ΦΠΑ, δεν είχε λειτουργήσει το σύστημα μέχρι στιγμής. Τώρα όμως ε, υπάρχει ένα νέο σύστημα και με τη βοήθεια αυτού μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις απάτες στον τομέα του ΦΠΑ και τις απάτες αυτές τύπου καρουσέλ. Αυτό είναι εθνικό σπορ θα έλεγα σε ορισμένε χώρες όπως παραδείγματο χάρη στην Ουγγαρία και θα χαρούμε να μειώσουμε. Το έργο τη Eurofisk θα πρέπει να είναι ένα σύστημα έγκυρη προειδοποίηση. όσον αφορά κάποιε ύποπτε συναλλαγέ. θα πρέπει να φροντίσουμε να μπορεί να ελεγχθεί ο αριθμός ε, μητρόφιπη α το που υποβάλλεται εκάστοτε, κατά πόσον ισχύει ή όχι. Αυτό είναι σημαντικό θέμα. Επίσης θα πρέπει να αποφύγουμε τα στοιχεία αυτά βέβαια να φτάσουν στα χέρια εκείνων που δεν δικαιούνται. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Να δώσω το λόγο πάλι στον εισηγητή για να απαντήσει και μετά μπορούμε να κλείσουμε τη συζήτηση. Θα ήθελα απλώς κυρία Πρόεδρε να ευχαριστήσω όλους όσους ε, έλαβαν ε, το λόγο ε, επ' αυτού του θέματος και, θέλουν, και όσους θέλουν να συμμετέσχουν στην τελική μορφή που θα λάβει αυτή η έκθεση. Θα προσπαθήσω να ικανοποιήσω όλες τις ανησυχίες, όλα τα αιτήματα και να διασκεδάσω όλες τις ανησυχίες για τα όσα ακούσαμε. Θα ήθελα να πω ότι συμφωνώ και είμαι σίγουρος ότι θα καταλήξουμε σε συμφωνία. Ευχαριστώ τους συναδέρφους και τον Αδόλφο Μπαρμπέρα Δεροσάλ, τον συμπατριώτη μου για τη συνεργασία του, αλλά και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την οποία είχαμε αγαστή συνεργασία όπως πάντα και ελπίζω ότι εντός του προβλεπωμένου χρονοδιαγράμματος θα καταλήξουμε σε μια ικανοποιητική λύση. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Δεν θέλω να υπενθυμίσω του συναδέλφου ότι εξεταστεί το σχέδιο τη έκθεση στι 11 Ιανουαρίου. Και θα περιμένουμε βέβαια του σκιώδει και του ενδιαφερόμενου να είναι εδώ. Θα περάσω στην έδρα τη Πρόεδρου και μετά θα περάσουμε στο επόμενο θέμα. I've had a temporary promotion, in <laughs> Πήρα μια προσωρινή προαγωγή εδώ για τις επόμενες δύο ώρε. ώρες. Και έχω καλή υποστήριξη της γραμματείας, αυτό είναι σημαντικό. Λοιπόν, ας περάσουμε στο επόμενο θέμα, αγαπητοί συνάδελφοι. Ασφάλεια του φωνδημού σε φυσικό αέριο, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα γενικά για μας, το Κοινοβούλιο. Και η Επιτροπή ε, Βιομηχανίας εξετάζει, αλλά έχουμε εδώ τον ε, εισηγητή μας, ε, τον κύριο Χουντή. Αν δεν θα το προφέρω καλά το όνομά σας, διορθώστε με. Κούντης, είπε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καλά προφέρατε το όνομά μου. Άλλωστε το ενδιαφέρον σε αυτή την περίπτωση δεν είναι το όνομά μου, αλλά το θέμα που καλούμεθα να συζητήσουμε στην προκειμένη περίπτωση και για, την οποία, και για τον οποίο μου δώσατε το λόγο. Αγαπητοί συνάδελφοι, δεν είναι προφανώς η πρόσφατη ρωσο-ουκρανική κρίση αερίου τούτου του Γενάρη η μόνη αιτία που συζητούμε αυτό το θέμα. Ο φόβος ενδεχόμενης επανάληψης πιθανόν να πιέζει να ληφθούν έγκαιρα μέτρα σχεδιασμού και αντιμετώπισης ενδεχομένων τέτοιων καταστάσεων. Βεβαίως οι αιτίες που συζητάμε με βάση την, την πρόταση κανονισμού που εισηγείται η Επιτροπή ούτως ώστε να υπάρξει ένας κανονισμός που θα αντικαταστήσει την ανεπαρκή και κατά την προσωπική μου άποψη οδηγία 2004 του 67 είναι οι λόγοι είναι ότι έτσι κι αλλιώς έχουμε αυξανόμενη εξάρτηση των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το εισαγόμενο αέριο. Υπάρχει αυξανόμενος κίνδυνος από τον εφοδιασμό λόγω του γεγονότος ότι οι αγωγοί διέρχονται μέσω τρίτων χωρών και υπάρχει αυξανόμενη ροή αερίου λόγω και της ανάπτυξης της εσωτερικής ευρωπαϊκής αγοράς. Αυτό οδηγεί στην ανάγκη ενός καλύτερου νέου σχεδιασμού και σε κάθε περίπτωση θέσπισης τέτοιων μέτρων ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η ασφάλεια για τον εφοδιασμό με φυσικό αέριο. Δεν επεκτείνομαι, δεν είναι ρόλος αυτής της ε, γνωμοδότησης να επεκταθεί σε γεωπολιτικές συγκρούσεις γύρω από το ενεργειακό, στην οικονομική κρίση που σίγουρα επηρεάζουν και την ενεργειακή πολιτική και την τροφοδοσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επηρεάζουν και την οικονομική κοινωνική συνοχή. Θα σταθώ μόνο στο αντικείμενο του κανονισμού λέγοντας ότι θεωρώ ότι η προσπάθεια που κάνει η Επιτροπή με αυτό το σχέδιο είναι θετική. Και είναι θετική διότι επαναλαμβάνω ότι η υφιστάμενη οδηγία 2004 του, 67, του, του ε, ε, Παύλα 67 είναι ανεπαρκής για να αντιμετωπίσει τις νέες εξελίξεις έτσι όπως προσπάθησα να τις περιγράψω. Επίσης, θεωρώ θετική την πρόθεση της Επιτροπής να εξασφαλίσει το συντονισμό σε κοινοτικό επίπεδο των ενεργειών για την ασφάλεια της ε, παροχής φυσικού αερίου. Ωστόσο, ωστόσο κατά την άποψή μου, αυτός ο κανονισμός πρέπει να απαιτεί, πρέπει, σε αυτόν τον κανονισμό πρέπει να γίνουν ορισμένες συγκεκριμένες τροπολογίες οι οποίες θα ενισχύσουν την ικανότητα να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη παροχή φυσικού αερίου σε περιόδους κρίσης. Το ποιες είναι αυτές τις τροπολογίες τις έχετε μπροστά στο κείμενο. Κωδικοποιημένα, για να ολοκληρώσω τη δική μου άποψη, τη δική μου παρουσίαση και να ακούσω τις δικές σας παρατηρήσεις, τέσσερα σημεία θα ήθελα να υπογραμμίσω σύντομα, ε, τα οποία υπηρετούν και ενισχύουν τον κανονισμό, κατά την άποψή μου, με βάση τις τροπολογίες. Το πρώτο σημείο. Θεωρώ ότι πρέπει να ενισχυθεί ο ρόλος που θα παίζει η αρμόδια αρχή και ιδιαίτερα στην ασφαλή παροχή φυσικού αερίου και ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσης. Αυτές, αυτή η πρόθεση ενισχύεται από τις τροπολογίες 3 και 7 για κάποιον που παρακολουθεί σχολαστικά το κείμενο. Η δεύτερη παρατήρηση. Νομίζω ότι πρέπει να θωρακίσουμε, να ενισχύσουμε τον κανονισμό και να θωρακίσουμε όλο αυτό το σύστημα από τυχόν κερδοσκοπικά παιχνίδια από την πλευρά των ιδιωτικών εταιριών παροχής φυσικού αερίου με τις τιμολογιακές τους πολιτικές, ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσης. Αυτή τη λειτουργία, αυτή την πλευρά νομίζω ότι την ενισχύουν οι τροπολογίες 1 και τροπολογίες 6. Τρίτη παρατήρηση, και σας παρακαλώ την προσοχή σας, θεωρώ ότι η τροπολογία μας που πρέπει να διορθώσει τον κανονισμό πρέπει να παραδέχεται και να αναγορεύει ως προτεραιότητα το δημόσιο και κοινωνικό συμφέρον, ιδιαίτερα σε περίοδους κρίσης, έναντι της έμφαση που δίνει σήμερα ο κανονισμός στο να μην διαστρεβλωθεί ο ελεύθερος ανταγωνισμός και η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Επιτρέπετε μου ένα πρόσθετο σχόλιο εδώ. Δεν πρόκειται περί του ιδεολογικού ζητήματο ανταγωνισμό, αγορά, σχεδιασμού και ούτε καθεξή. Εδώ είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο το θέμα. Σε περιόδου κρίση, την οποία έζησαν οι Ευρωπαίοι πολίτε, νομίζω ότι η προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στο κοινωνικό και στο δημόσιο συμφέρον. Δηλαδή, να μην σταματήσει η τροφοδοσία επειδή ενδεχομένως θα υπάρξουν και έκτακτα μέτρα εξασφάλισης αυτής της τροφοδοσίας έναντι της αρχής να μην στρεβλώσει η αγορά. Ως προς αυτή τη λειτουργία λειτουργούν, ενισχύουν οι τροπολογίες 4, 5 και 6. Και το τέταρτο και τελευταίο σημείο είναι ότι κατά την άποψή μου στον σχεδιασμό στην αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων εκτός από την, ε, ε, τους κρατικούς φορείς, τις βιομηχανίες, τις εταιρείε, εταιρείες, νομίζω ότι πρέπει να μπει ο, ο παράγων πελάτης, ο παράγων καταναλωτής. Επομένως, οι τροπολογίες 3 και οι τροπολογίες 10 απαιτούν, ζητούν τη συμμετοχή οργανώσεων πιθανών καταναλωτών σε τέτοιες καταστάσεις, στο σχεδιασμό και στο συντονισμό. Σας ευχαριστώ πολύ και θα ήθελα να ακούσω με προσοχή τις παρατηρήσεις σας. Ήταν ε, πολύ καλή παρουσίαση τη θέση αυτή για την Επιτροπολογία. Οι σκιώδει ηγητέ τώρα, ο κ. Φέρμπερ, εξ ονόματο του ΕΛΚΑ. Ναι, σα ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν βέβαια να ευχαριστήσω τον συνάδελφο για την έκθεση που υπέβαλε. Τα ελληνικά μου δεν είναι πολύ καλά και αυτό δεν τολμάω να προφέρω καν το όνομά σας. Είναι πράγματι αληθές και σημαντικό ότι πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για αυτό που ζήσαμε τρεις φορές από την αρχή του χρόνου. Μια, δύο φορές με το φυσικό αέριο, μία φορά με το πετρέλαιο. Είναι ένα πρόβλημα στην τροφοδότηση με ενέργεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι επειδή κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν τήρησαν τις υποχρεώσεις τους, αλλά στην ε, συγκεκριμένη περίπτωση πρόκειται για μια χώρα τράνζιτ, για και θα πρέπει να έχουμε μια λύση και είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων που η Κομισιόν πραγματικά δέχθηκε την εντολή αυτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και προετοίμασε τις σχετικές προτάσεις. Θεωρώ όμως ότι θα πρέπει να έχουμε μηχανισμούς οι οποίοι αναφέρονται συγκεκριμένε συγκεκριμένες περιόδους κρίσης. Και η περίοδη κρίσης είναι ακριβώς όταν διακοπή ή τροφοδότηση με φυσικό αέριο από μία από τις κύριες χώρες ε, από τις οποίες αγοράζει η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να εξασφαλιστεί, λέω. Και γι' αυτό δεν ξέρω αν θα πρέπει να έχουμε τόσο πολύπλοκο σύστημα ε, διακανονισμού που δίνει την εντύπωση ότι η κρίση είναι η φυσιολογική ε, περίπτωση. Η κρίση θα πρέπει να παραμείνει κρίση. Να έχουμε δηλαδή κάποια μέσα για την Περίοδος στην οποία θα παρουσιαστεί η κρίση. Εάν θεωρήσουμε ότι η κρίση είναι φυσιολογική, ε, καταστρέφει πολλά πράγματα σε μια αγορά η οποία έχει δημιουργηθεί εδώ και πολλά χρόνια και από οικονομικούς λόγους ή τουλάχιστον θα διασφιβητεί όλα αυτά τα στοιχεία της εν λόγω αγοράς. Και γι' αυτό έχω κάποιες παρατηρήσεις να κάνω όταν αναφέρω το θέμα της ενδυνάμωσης ε, του ρόλου των αρχών. Αυτό θέλουμε. Θέλουμε δηλαδή μέσω των αρχών αυτών να παρέμβουμε και στον καθορισμό των τιμών. Έχω κάποια προβλήματα εδώ κατανόησης γιατί η εμπειρία μου των αρχών του έτους ήταν ότι ακριβώς εκείνες οι χώρες στην οποία υπήρχε δυνατότητα αποθήκευση φυσικού αερίου μπόρεσε να γίνει μια τροφοδότηση εκείνων των χωρών που είχαν πληγεί ιδιαίτερα από το γεγονό ότι από τη Ρωσία δεν μπορούσαν να πάρουν τίποτα. Υπάρχουν κάποια τεχνικά προβλήματα γιατί η αγωγή αυτή του φυσικού αερίου μπορούσαν να μεταφέρουν μόνο προς τη μία κατεύθυνση, θα πρέπει να μετατραπούν ή να μπορούν να μεταφέρουν και στους δύο κατευθύνσεις. Δεν είναι λοιπόν θέμα αρχών, είναι θέμα τεχνικών προβλημάτων. Δεύτερον, δεν επιτρέπεται οι χώρες οι οποίες αγοράζουν σε τιμή αγορά το φυσικό αέριο για την εξασφάλιση των δικών τους υποχρεώσεων σε ένα χειμώνα, χωρίς κρίση δηλαδή φυσικά, αναγκάζονται να πουλήσουν αυτό το φυσικό αέριο σε άλλες τιμές, χαμηλότερες τιμές δηλαδή. Αυτό δεν είναι προς όφελος και συμφέρον εκείνων που είχαν αγοράσει το φυσικό αέριο στην τιμή αγοράς. Και αυτό λοιπόν είναι ένα θέμα που θα πρέπει να εξετάσουμε λεπτομερώς. Και το άλλο θέμα που θέλω να θίξω έτσι στα γρήγορα είναι το θέμα της ομάδας των προστατευομένων πελατών. Ο εισηγητής μας διευρύνει τον κύκλο των προστατευομένων αυτών πελατών και δεν ξέρω αν έχουμε ε, συμφέρον να, είμαστε όλοι, να είναι όλοι προστατευόμενοι. Έτσι κατάλαβα εγώ την πρόταση αμενοι, όλοι προστατευόμενοι ε, πελάτες δεν χρειάζομαστε μια πραγματική αγορά φυσικού αερίου θα λύσουμε το πρόβλημα διαφορετικά Βέβαια θα συμφωνούσα, πρέπει να σας το πω και αυτό. Λοιπόν, η συζήτηση στην Επιτροπή ε, βιομηχανίας που είναι επί της αρμόδια είναι κάπως διαφορετική και θα χαιρόμουν να συμφωνήσουμε εδώ στην Οικονομική Επιτροπή σε μια λύση που να τονίζει ακριβώς αυτές τις οικονομικές πτυχές γιατί θα είναι καλό να χρησιμοποιήσουμε και μέσα της ε, οργάνωσης αγοράς ούτως ώστε να μπορούμε να βρούμε μια λύση. Δηλαδή δεν χρειαζόμαστε αρχές, δεν χρειαζόμαστε διακανονισμούς. Η αγορά μόνη της θα μπορέσει να το διακανονίσει και θα πρέπει να είμαστε αρκετά κοντά σε αυτό που συζητιέται στην Επιτροπή Βιομηχανίας και σε αυτό που πρότεινε η Κομισιόν. Έτσι θα μπορέσουμε νομίζω να κινηθούμε περαιτέρω. Ευχαριστώ πολύ. Uh, thank Ευχαριστούμε πολύ κύριε Φέμπερ. Ο κύριος Κούτσας ε, εκ μέρους των ε, σοσιαλιστών. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα επιτρέψτε μου να πω ότι η έκθεση αυτή αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός, προς την ε, ασφάλεια εφοδιασμού αερίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή η ασφάλεια είναι καθοριστική σημασίας για την εύρυθμη λειτουργία της ευρωπαϊκής οικονομίας ε, εδώ και πολύ καιρό. Ε, πάνω από 20% της παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος προέρχεται από αέριο και το 60% του αερίου που καταναλώνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση εισάγεται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν μάλιστα χώρες που εξαρτώνται πλήρως από την εισαγωγή αερίου. Αυτός λοιπόν ο κανονισμός ε, προβλέπει δύο πράγματα. Πρώτον, την πρόληψη κρίσεων και δεύτερον, τη διαχείριση κρίσεων. Ε, τη διαχείριση έκτακτων ε, περιπτώσεων. Θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Χουντή για την έκθεσή του. Εγώ συμφωνώ με την προσέγγιση του και με την άποψή του γιατί είναι πολύ σημαντικό το να ελέγχει κανείς τις ε, τιμολογιακές πολιτικές και είναι και πολύ σημαντικό να ελέγχει κανείς τις πληθωριστικές τιμές. Εξάλλου, οι εταιρείες παραγωγής αερίου διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ευρωπαϊκή αγορά. Ένα άλλο σημαντικό θέμα είναι ε, σχετικά με τις δαπάνες, ε, ε, τον επιμερισμό δαπανών για την κατασκευή νέων υποδομών. Είναι λοιπόν σημαντικό κατά την άποψή μου να ενθαρρύνουμε τις επενδύσεις για τη δημιουργία υποδομών και τις επενδύσεις για τη δημιουργία νέου δυναμικού εφοδιασμού. Η ασφάλεια προέρχεται προφανώς και από τη δημιουργία νέων υποδομών, ευρύτερων υποδομών που προσφέρουν και άλλες εναλλακτικέ λύσεις πέρα από το ρωσικό αέριο. Μία τέτοια δυνατότητα επιλογής είναι ο γογός Ναμπούκο. Εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι να μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε προγράμματα, ε, παραδείγματο χάρη με επιστώσεις από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Να σας πω εξάλλου ότι ε, προβλέπονται ε, διαφορετικές απαιτήσεις απέναντι στους προμηθευτές. Αυτό όμως πρέπει να τροποποιηθεί, γιατί εγώ πιστεύω ότι όλοι οι παίκτες εισαγωγικά πρέπει να είναι προετοιμασμένοι σωστά, έτσι ώστε να έχουμε μια νέα και καλύτερη υποδομή. Ο κύριος Λάμπερτς ε, από τους Πράσινους ε, και ο ε, δεν θέλετε τίποτα να πείτε. Πάρα πολύ ωραία. Άρα δηλαδή μπορούμε και εμείς να κρατήσουμε το χρόνο μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Άλλος παρακαλώ επιθυμεί κάποιος άλλος το λόγο. Η κυρία Γκυρή παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό να, το ότι μπορούμε και συζητάμε αυτή την πρόταση. Η ασφάλεια εφοδιασμού με αέριο για μας είναι πολύ σημαντική. Από χθε, από την 1η Δεκεμβρίου, μην ξεχνάτε ότι έχουμε αποκτήσει και περισσότερες αρμοδιότητες λόγω της θέσης ισχύ της συνθήκης Λισαβόνας. Έχουμε περισσότερες αρμοδιότητες για ενεργειακά θέματα. Άρα δηλαδή υπάρχει νομική βάση. Η συνθήκη της Λισαβόνας αναφέρει παραδείγματο της λισαβονας αναφερει παραδειγματος χαρη ότι τα κράτη-μέλη οφείλουν να επιδεικνύουν φιλαλληλία, αλληλεγγύη αν θέλετε, ανάμεσά τους και να μην εκτίθενται σε ακραίες καταστάσεις. Εγώ λοιπόν θα ήθελα να κάνω τρεις παρατηρήσεις για αυτή την πρόταση του κυρίου Χουντή. Πρώτον, ε, αυτή είναι τεχνικής φύσεως η πρώτη μου παρατήρηση. Ο κύριος Φέρμπερ ήδη αναφέρθηκε ε, στο τι μπορούν να κάνουν οι αγωγοί και τι όχι. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν όλοι οι αγωγοί να μπορούν να προσφέρουν τα πάντα. Αυτό δεν γίνεται. Δεν μπορεί ένας αγωγός να κατευθύνεται την ίδια στιγμή σε διαφορετικές κατευθύνσεις. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό το ότι η αγωγοί δεν θα πρέπει να έχουν μόνο κατεύθυνση από Ανατολάς προς Δυσμάς, αλλά και από Βορρά προς Νότο. Και το βρίσκω πολύ καλό το ότι η Κομισιόν δίνει αυτή τη δυνατότητα και στο μέλλον αυτή η δυνατότητα πρέπει να τονιστεί περαιτέρω. Δεύτερη παρατήρηση, σημαντική κατά την άποψή μου, σχετικά με περιόδους κρίσης. Κοιτάξτε, εγώ συμφωνώ με την Επιτροπή ότι στην περίπτωση κατά την οποία ε, χάσουμε το 10% των εισαγωγών αριού, αυτομάτως προκύπτει κρίση. Εγώ άκουσα μερικούς που λένε ότι όχι, κρίση ε, προκύπτει στο 20%. Τούτο όμως, αυτή η αύξηση του ποσοστού, αντιφάσκει με την αρχή της ε, φιλαλληλίας. Υπάρχουν λοιπόν ορισμένα κρατημέλη όπου ακόμα και αν λείπει αυτό το 10% ε, αντιμετωπίζουν τεράστιο πρόβλημα. Τρίτη μου παρατήρηση. Εγώ δεν βλέπω στο κείμενο που έχει, καταθέσει, έχει κατατεθεί καμία απάντηση στο ποιος πρέπει να λάβει μέτρα για την εξασφάλιση της ε, τροφοδοσίας. Ποιος είναι ο ρόλος των κοινοτικών θεσμών, ποιος είναι ο ρόλος των κρατών μελών. Κατά αυτό το θέμα πρέπει να εξετάσουμε περισσότερο σε βάθος. Κύριε Πρόεδρε, εγώ θα ξεκινήσω λιγάκι με ανορθόδοξο τρόπο, αν μου επιτρέπετε. Κοιτάξτε, στην ε, πολιτική, κατά κανόνα δεν λέει κανείς ότι έχει πολλούς φίλους. Όμως, ο πρώην Υπουργός Ενέργειας και Εμπορίου της ε, χώρας μου της, της Τσεχίας ήταν φίλος μου, ήταν φίλος μου και νομίζω ότι ήταν ένας από αυτούς τους τρεις ή τέσσερις που στις αρχές αυτού του έτους αγωνίστηκαν για την ε, επαναλειτουργία ε, των προμηθειών ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση από την Ουκρανία. Και επειδή είναι φίλος μου, ξέρω τι έγινε στο παρασκήνιο. Ξέρω τι διαδραματίστηκε. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα κι εγώ τι ε, πληροφορίε που έχω συγκεντρώσει να σα ανακοινώσω να καταλάβουμε λιγάκι περί τίνο πρόκειται. Κοιτάξτε, η κρίση προέκυψε διότι κατέρευσαν οι προσωπικέ οι εσωτερικές σχέσεις ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία. Ό,τι κανονισμό και ε, αν είχαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τίποτε θα μπορούσε να βοηθήσει εκεί στι σχέσει ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία. Αυτό ήταν το πρώτο βασικό πρόβλημα. Το δεύτερο ήταν το εξή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση απλά δεν έχει ε, επάρκεια σε πλουτοπαραγωγικές πηγές. Δηλαδή, ό,τι και να κάνουμε, ό,τι και κανονισμό και αν ε, εκπονήσουμε, θα μπορέσουμε να παράγουμε φυσικό αέριο. Απλά δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα στον τομέα αυτό. Και στο μέλλον, ούτε και στο μέλλον θα μπορούμε να επηρεάζουμε τις σχέσεις ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία. Μα ό,τι συνθήκη Λισαβόνας ή οποιαδήποτε άλλη και αν έχουμε, Τίποτα δεν θα βοηθήσει αυτό. Τώρα λοιπόν, αφού τελείωσα με αυτά, θα σας πω και εγώ τα δικά μου τα επιχειρήματα. Εγώ συμφωνώ με αυτά που είπε ο κύριος Φέμπερ και ο εισηγητής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να διαφοροποιήσει τις πηγές της ή αν θέλετε να διαφοροποιήσει τα συστήματά της τα οποία μας προσφέρουν την ε, τροφοδοσία. Πρέπει λοιπόν στην Ευρωπαϊκή Ένωση να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον όχι με πάρα πολλές ρυθμίσεις, όπου οι επενδυτές θα μπορούν να επενδύουν ελεύθερα και σε νέα συστήματα που θα ε, προσφέρουν τη διασύνδεση των ε, συστημάτων αερίου. Στην περίπτωση όμως αυτή δεν μπορούμε να μιλάμε για τιμές γιατί αν η τιμή της αγοράς ε, δεν θεωρείται το καθοριστικό στοιχείο ε, που ορίζει την ε, τιμή και τη ζήτηση, αν εμείς θέλουμε να ορίσουμε τις τιμές με κάποιο διοικητικό τρόπο, ε, τότε και εμείς εμποδίζουμε τις εταιρείε να προσποριστούν κέρδος. Μα δεν είναι κακό το κέρδος, γιατί το βλέπετε κακό. Άμα υπάρχει κέρδος, μπορεί κανείς να επενδύσει και στη σύγχρονη τεχνολογία. Γι' αυτό λοιπόν εγώ προσωπικά πιστεύω ότι δεν πρέπει να εκπονούμε υπερβολικές ρυθμίσεις για τα ε, εμπορεύματα, για αυτά τα αγαθά. Να μην ακολουθήσουμε αυτό το δρόμο. Ε, εμείς θα καταθέσουμε σχετική τροπολογία, έχουμε ακόμα χρόνο μέχρι τις αρχές Ιανουαρίου, όμως εγώ θεωρώ ότι υπάρχουν τρία αντιφατικά, επίμαχα θέματα εμείς θα τα αντιμετωπίσουμε αυτά με πολύ μεγάλη σύνεση. Καταρχήν, όλες τις τροπολογίες για τις οποίες μιλάμε ε, αναφέρονται στην αποκαλούμενη δίκαιη τιμή. Εμείς δεν το στηρίζουμε αυτό, μα δεν υπάρχει αυτό δίκαιη τιμή. Δεν υπάρχει δίκαιη τιμή στην αγορά, fair price. Εξάλλου, θα είμαστε πολύ προσεκτικοί αναφερόμενοι στον ρόλο των ε, οργανώσεων πελατών ή καταναλωτών. Ε, θα είμαστε πολύ προσεκτικοί στο κατά πόσο αυτοί μπορούν να έχουν λόγο στην ε, διαμόρφωση τη τιμή αγορά. Και ένα τρίτο μου επιχείρημα, συμφωνώ εδώ με τον κύριο Πέρμπερ, πολύ προσεκτικοί θα είμαστε επίση κρίνοντας αυτή την ομάδα των προστατευμένων καταναλωτών. Γιατί εμείς πιστεύουμε ότι αυτή η ομάδα είναι ιδιαίτερα ευρία και εκτεταμένη και εδώ θέλουμε να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Επανέρχομαι στον εισηγητή, μήπω ε, θέλει να σχολιάσει κάποια θέματα, κυρίως ε, ίσως αυτά που έχουν σχέση με την αγορά. Και τι πρέπει να κάνουμε όταν αποτυγχάνει η αγορά. Είμαι σίγουρη ότι θέλετε να κάνετε κάποια σχόλια. Κύριε Χουντή, έχετε το λόγο. Θέλω να ευχαριστήσω, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για τις παρατηρήσεις, τις αντιρρήσεις που διατύπωσαν ε, δεν ξέρω ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα. Νομίζω ότι οι τροπολογίε, αν είμαι καλά ενημερωμένο, μπορούν να κατατεθούν μέχρι τι 10 12 το ας πει το Προεδρείο, η Γραμματεία της Επιτροπής, μέχρι πότε είναι η προθεσμία για να δουλέψουμε. Αν είναι έτσι, Προφανώ πρέπει να συνεχίσουμε και εγώ να δουλεύω και οι συνάδελφοι για να καταθέσουν τι δικέ του τροπολογίε. Δύο σχόλια, ένα σχόλιο στην αρχή. Προφανώ αν θέλει κανεί να μελετήσει σε βάθο αυτό το θέμα και πρέπει να έχει γνώση και τεχνικών προβλήματων. Ε, θα σας έλεγα δεν στερούμε τέτοιων γνώσεων, είμαι μηχανικός, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα τώρα. Και δεύτερο, ε, όσο είναι δυνατόν να μην επεκταθεί, να μην επεκταθεί, δεν ξέρω αν είμαστε συνάδελφοι, να μην επεκταθεί το θέμα σε μια γενικότερη συζήτηση που είναι ανοιχτή σχετικά με την πολλαπλότητα των πηγών τροφοδοσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις πιέσεις που ασκούνται και τα πολιτικά παιχνίδια, που και αυτά επηρεάζουν όλο αυτό το κλίμα που κάνουμε. Όμως είμαστε, είμαστε υποχρεωμένοι να περιουστούμε στο αντικείμενο λαμβανωμένο υπόψη ε, συζητώντας σε άλλα επίπεδα αυτή τη συζήτηση, αυτό το θέμα. Αυτό είναι το πρώτο σχόλιο. Το δεύτερο, όπως ε, είπατε κυρία Πρόεδρε, υπάρχει το θέμα της αγοράς. Δεν μπορεί κατά την προσωπική μου άποψη να αφήσουμε την αγορά να ρυθμίσει τέτοια θέματα και να λειτουργήσει ε, ομολογώ απρόσκοπτα σε συνθήκες κρίσης. Δεν μιλώ για το θεμητό, παραδεκτό, αποδεκτό κέρδος. Μιλώ για κερδοσκοπικά παιχνίδια που εξελίσσονται σε τέτοιες περιόδους και υποθέτω, δεν ξέρω αν είναι εκπρόσωπος της Επιτροπής εδώ, ότι και το σχέδιο κανονισμού έχει μια τέτοια επιφύλαξη να τα αφήσει στην αγορά. Επομένως, ε, εδώ πρέπει να το δούμε ότι πρέπει να υπάρξει ε, η παρέμβαση, ο ρόλος αναβαθμισμένος της αρμόδιας αρχής Τη ομάδα συντονισμού που να τα προλαβαίνει αυτά. Και ξαναλέω, όχι να μην υπάρχει κέρδος, αλλά να μην υπάρχει αυτό το κερδοσκοπικό παιχνίδι που πολύ φοβούμαι εξελίσσεται σε τέτοιες ε, περιπτώσεις. Και το τελευταίο σχόλιο για τους προστατευόμενους πελάτες. Ε, κοιτάξτε ε, αγαπητοί συνάδελφοι, εκεί δεν μπορεί να μην πάρεις υπόψη σου και στο θέμα ότι οι προστατευόμενοι πελάτες με αποφασιστική γνώμη πρέπει να έχουν και μικρομεσαίε μικρομεσαίες νοσοκομεία, σχολεία, εφόσον έχουν και με τον τρόπο έκφραση εφόσον έχουν συνδεθεί με το αέριο και στο συντονισμό ε, οι ομάδε καταναλωτών. Αρκετοί συνάδελφοι, ίσω να μην είναι στη δική, μου, στη ρητορική, ισχυρίζονται ότι η συνθήκη τη Λισαβόνα δίνει περισσότερα δικαιώματα στου πολίτε και να παρεμβαίνουν να... στη λήψη αποφάσεων. Θα παρακαλούσα να σκεφτούν και από αυτή την οπτική, μήπω είναι μια ευκαιρία να δώσουμε τέτοια δικαιώματα έτσι περαιτέρω. Σα ευχαριστώ πολύ. Um, uh, Ευχαριστούμε πολύ κύριε Χούντι. Ε, κοιτάξτε συνάδελφοι, θα ήθελα να σας λιγάκι το θέμα του χρονοδιαγράμματος πράγματι μέχρι 10 Δεκεμβρίου ε, μπορούμε να καταθέσουμε τροπολογίες. Τον Ιανουάριο θα τις εξετάσουμε και θα ψηφίσουμε πίσω τον Ιανουάριο. Άρα δηλαδή το χρονοδιάγραμμα είναι αρκετά σφιχτό. Κύριε Φέρμπερ, παρακαλώ. Κοιτάξτε, μία ερώτηση έτσι κάπως περίεργη. Από ό,τι άκουσα υποτίθεται από τις 11 Ιανουαρίου θα έχουμε εδώ ακροάσεις επιτρόπων. Τι θα γίνει με τη δική μας την επιτροπή, θα συνεδριάσουμε εμείς, ε, τι θα κάνουμε εμεί, ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή επεξεργαζόμεθα το δικό μα το χρονοδιάγραμμα γιατί δεν έχουν επιβεβαιωθεί οι ακροάσει των επιτρόπων. Μόλι επιβεβαιωθούν θα σα ενημερώσουμε γιατί είναι πολύ δύσκολο για μας να προβλέψουμε τι θα γίνει. Α κάνουμε το δικό μα το χρονοδιάγραμμα, α το τηρήσουμε και βλέπουμε μετά, θα το προσαρμόσουμε. Σα ευχαριστούμε πολύ συνάδελφοι, ευχαριστούμε πολύ για τι παρεμβάσει σα στη συζήτηση. Πάμε τώρα στο επόμενο θέμα τη ημερησία διάταξη έχουμε την ε, έκθεση για την πρόθεση της χρηστής ε, διακυβέρνησης στο φορολογικό τομέα. Ο εισηγητής, ο κύριος Ντομένιτσι, θα μας κάνει την παρουσίαση. Ευχαριστώ. 59 τροπολογίες υπευλήθησαν 12 από μένα, από τον εισηγητή και οι υπόλοιπες 38 από τους συναδέλφους. Κάναμε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων με την παρουσίαση της εκθέσεως ε, στις 10 Νοεμβρίου. Η δε ψηφοφορία στην Επιτροπή προβλέπεται για τις 11 Ιανουαρίου και η ψηφοφορία στην Ολομέλεια ε, τον Φεβρουάριο. Σας ευχαριστώ για τη συμβολή σας και το ενδιαφέρον που δείξατε εναντί αυτής της εκθέσεως. Πιστεύω ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις, ε, υπάρχουν συνθήκες για μια καλή συνεργασία και την εξέβρεση σύγκλησης και συμβιβασμών όχι για όλα αλλά για σχεδόν όλα τα θέματα που θίγουν οι τροπολογίες. Πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε και συγχώνευση κάποιων τροπολογιών από τις 26 που έχουν υποβληθεί ας πούμε ε, από τον συνάδελφο Ζωρή τον οποίο ευχαριστώ για την συμβολή του και πιστεύω ότι είναι σημαντικό να διατηρήσουμε μια ισορροπία στην έκθεση. Ισορροπία μεταξύ, όπως λέω στην έκθεση, του εσωτερικού επίπεδου και του διεθνούς επίπεδου για τη χρηστή διαχείριση και διακυβέρνηση. Αυτό θα πρέπει να το έχουμε κατά νου και κατά την συζήτηση των τροπολογιών. Ελπίζω ότι μέχρι τις 11 Ιανουαρίου θα μπορέσουμε να εργαστούμε συμβιβαστικά, επικοδομητικά, με ενωτικό τρόπο, χωρίς βεβαίως να αποποιηθούμε των βασικών αρχών που διέπουν αυτήν την έκθεση και την εμπνέουν. Ευχαριστώ. 59 λοιπόν οι τροπολογίε που έχουν κατευθεί και θα ήθελα μετά να ζητήσω από τον Ισκέδη Συγητή να παρέμβει. Πρώτα, κυρία Κιόρ. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω εκ βάθου βάθου καρδία τον εισηγητή μα για την θαυμάσια δουλειά που έχει κάνει. Είναι σαφέ ότι μπορέσαμε τελικά να συνεργαστούμε άριστα μαζί του. Νομίζω λοιπόν ότι θα μπορούσαμε τελικά να καταλήξουμε σε μια συμφωνία για όλα τα θέματα. Έχουμε λοιπόν εδώ ένα θέμα ε, που έχει ήδη συζητηθεί παλαιότερα αναφέρθηκε ότι έχει διασπανιστεί, διασπαθιστεί, με συγχωρείτε, πολύ χρήμα. Ε, και αυτό λόγω των δημοσιονομικών των κρατομέλων δεν είναι επιτρεπτό. Η πρόταση λοιπόν δεν έχει ως ε, στόχο το που ακριβώς επιθυμούμε να εμβαθύνουμε τη συνεργασία για τα φορολογικά θέματα, αλλά η όλη συζήτηση είναι κατά πόσον θέλουμε να διαφυλάξουμε αυτό που υπάρχει και τι θα κάνουμε με τις ε, offshore εταιρείες. Εγώ τις δικές της τροπολογίες ε, τις ε, έχω εξηγήσει επανειλημμένα στην Επιτροπή μας. Εγώ ε, προσπάθησα σε συγκεκριμένα προβλήματα να διατυπώσω συγκεκριμένες απαντήσεις. Εκείνο το οποίο κατά την άποψή μου είναι ιδιαίτερα σημαντικό είναι το ότι οτιδήποτε αποφάσισαν οι G20 πράγματι αυτό πρέπει να υλοποιηθεί γιατί σε τελική ανάλυση αντιμετωπίζουμε μια κατάσταση όπου έχουμε θαυμάσια και μεγαλοπίβολα σχέδια. Όμως τώρα φτάνουμε στο διατάφτα. Αυτά πρέπει να εφαρμοστούν. Ε, είναι λοιπόν σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να ε, παίξει πρωτοπόρο ρόλο για μας, για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είναι πολύ σημαντικό το ότι εδώ πρόκειται για ένα τομέα όπου ναι μεν τα κράτη-μέλη δεν συμφωνούν πάντοτε, όμως οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τις περισσότερες τουλάχιστον φορές, στηρίζονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γι' αυτό λοιπόν ε, στον τομέα της ε, χρηστής ε, διακυβέρνησης συμφωνούμε με τα περισσότερα που περιλαμβάνονται στην ανακοίνωση της Κομισιόν. Τώρα, όσον αφορά τον εισηγητή, τον κύριο Ντομένιτσι, έχουμε συζητήσει επανειλημμένα μαζί του και νομίζω ότι οι περισσότερες τροπολογίες θα τη στηρίξει, θα τις δεχθεί, τις δικές μας εννοώ. Δηλαδή, ένα σύστημα κινήτρων, αυτό θα πρέπει να εισαχθεί και αυτό το σύστημα θα οδηγήσει στο ότι οι φόροι που έχουν εισπραχθεί από άλλο κράτος μέλος να υπάρχει κάποια ε, συμμετοχή σε αυτό και οι αρχές του ΟΣΑ που λένε ότι αν μια χώρα έχει συνάψει συμφωνίες διαφορολογικά θέματα με 12 χώρες, αυτή η χώρα είναι, χαρακτηρίζεται ως συνεργαζόμενη. Αυτό όμως δεν αρκεί γιατί υπάρχουν εκατοντάδες χώρες ολόκληρου τον κόσμο. Μετά υπάρχει ε, ένα θέμα όπου ο κύριος ε, Ντομένιτσι ε, αναφέρεται στο CCDT αυτό είναι ένα πολύ ε, λεπτό θέμα τόσο στο Κοινοβούλιο όσο και στο Συμβούλιο. Η δική μου λοιπόν η τροπολογία έχει ως στόχο το συμβασμό. Περί τι πρόκειται. Ο κύριος Ντομένιτσι επιθυμεί να έχει σαφέστατη διατύπωση για το CCDT. Άλλοι πάλι θέλουν να διαγράψουν αυτή την αναφορά. Συμβιβαστικά λοιπόν εγώ λέω το εξής. Να διευκρινίσουμε τι είναι αυτό το CCDT και να αναφερόμεθα μόνο στις ε, τιμές ε, μεταφοράς. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το σύστημα του συγκρίσιμου κέρδους θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και τα κέρδη των θηγατρικών. Γιατί αν η κερδοφορία της θηγατρικής είναι πολύ κάτω από το μέσο όρο του τομέα, τότε ελοχεύει ο κίνδυνος. Αυτή η θηγατρική να ε, μεταφέρει τα κέρδη της σε φορολογικό παράδεισο. Ε, αυτό λοιπόν θα μπορούσε να είναι επικίνδυνο για το CCTV. Κοιτάξτε, κοιτάξτε υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Ε, η υποχρέωση των ε, συναδέλφων που έχουν εγκατασταθεί ε, σε offshore εταιρείε και έχουν την υποχρέωση να δηλώνονται. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σκιώδη ε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να μου επιτρέψετε να σχολιάσω τις ε, τρεις τροπολογίες ε, τις οποίες κατέθεσα εγώ. Η πρώτη μου τροπολογία έχει να κάνει με τις αναπτυσσόμενες χώρες. Κατά την άποψή μου τουλάχιστον. Αναφέρομαι στην παράγραφο υπαριθμών 16. Εγώ στηρίζω ανεπιφύλακτα τη δουλειά που έχει γίνει για να προάγουμε τη χρηστή διακυβέρνηση και τη δουλειά του εισηγητή. Στο άρθρο 16 εδώ προτείνεται η Ευρωπαϊκή Ένωση να εξτάσει το ενδεχόμενο ε, σε ειδικού φόρου για ε, οργανισμούς, οντότητες που δεν επιδεικνύουν πνεύμα εργασίες. Τι είναι όμως αυτό, αυτό δεν έχει οριστεί. Αυτά τα συσυντητή που λέγαμε προηγουμένως. Αυτό όμως ε, μπορεί να αφορά, τουλάχιστον αφορούσε κατά το παρελθόν, τις ιδιαίτερα φτωχές χώρες. Γι' αυτό λοιπόν εγώ δεν συμφωνώ αυτομάτως να τους επιβάλλουμε κάποιο πρόστιμο ή ε, κάποια ειδική εισφορά και να αφορά αυτό ανθρώπους που έρχονται εδώ για να μαζέψουν κάποια χρήματα να τα στείλουν στην πατρίδα τους. Ίσως λοιπόν θα πρέπει πριν καθορίσουμε στο φόρο ή στο πρόστιμο να δούμε τι άλλες επιλογές έχουμε στη διάθεσή μας. Γι' αυτό λοιπόν ε, προτείνω να διαγράψουμε αυτό το ειδικό Ευρωπαϊκή επιβάρυνση και να πούμε καλύτερα η Ευρωπαϊκή Ένωση να εξετάσει τη βεντάλια επιλογών που έχει στη διάθεσή της. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Κιούρη, την ε, οποία και άκουσα προηγουμένως, ε, το θέμα ε, της φορολογικής βάσης Common Consolidated Tax Base. Αυτό που ενδιαφέρει είναι ότι τελικά όλοι μας συμφωνούμε ότι θέλουμε να αντιμετωπίσουμε τη φορολογική απάτη και την φοροδιαφυγή. Από τη στιγμή λοιπόν που αρχίζουμε να θέλουμε να εισάγουμε αυτό το πολύ αμφιλεγόμενο που είπατε προηγουμένως ότι θα πρέπει να περάσουμε σε μια κοινή ε, φορολογική βάση αυτομάτως δημιουργούνται αντιφάσεις και διαμάχες ανάμεσα στα κράτη-μέλη που υπονομεύουν αυτή την έκθεση που στη τελική ανάλυση έχει ως στόχο να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τη φοροδιαφυγή και την φοροαποφυγή. Γι' αυτό εγώ λοιπόν λέω ας το αφήσουμε αυτό, ας το διαγράψουμε και ας επικεντρωθούμε στο βασικό στόχο αυτής της έκθεσης. Το τρίτο που θέλω να πω αφορά την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών. Γνωρίζω βέβαια ότι εδώ πρόκειται για ένα ιδιαίτερα λεπτό θέμα, αλλά θα ήθελα να καταλάβετε κι εσείς γιατί το θέμα αυτό είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο στην, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η κυβέρνηση του Ηνωμένου ε, δεν έχει να επιδείξει ε, καλό ιστορικό ε, σχετικά με τα φορολογικά πολλών ατόμων. Υπήρξαν πολλές περιπτώσεις όπου χάθηκαν πληροφορίες και η χειρότερη περίπτωση ήταν πριν από τρία χρόνια περίπου όταν η κυβέρνηση έχασε δύο σκληρούς δίσκους ηλεκτρονικού υπολογιστή που περιείχαν φορολογικές πληροφορίες. Το όνομά μου, τη διεύθυνσή μου ε, τον τραπεζικό μου λογαριασμό και αυτό αφορούσε 25 εκατομμύρια, 25 εκατομμύρια ανθρώπους. Ε, ήταν εκεί το όνομα το δικό μου, της κυρίας Σουίνμπας, της κυρίας Στάλης και είμαι σίγουρο, ε, Αιλίν, και εσύ ε, θα είχε οικογένεια και γνωστούς που επηρεάστηκαν από αυτό. Άρα δηλαδή, αν θέλετε, το Ηνωμένο Βασίλειο δεν έχει να επιδείξει καλή φήμη στο πώς χειρίζεται τις πληροφορίες για τους φορολογούμενους. Δυστυχώ. Αυτό είναι ένα από τα θέματα όπου το Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να καταβάλει προσπάθεια. Του χρόνου ε, θα έχουμε ευτυχώ αλλαγή κυβέρνηση, αλλά εντωμεταξύ άλλα κρατημέλη, οποτεδήποτε σκέπτονται την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών, να το σκεφτούν δυο φορέ. Να ε, σκεφτούν ότι μπορεί οι ειδικέ του οι δικοί του, οι τραπεζικοί λογαριασμοί <laughs> να ενδοθούν ω πληροφορίε στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και θα σα έλεγα να προσέξετε πάρα πολύ και μακριά τα χέρια από αυτό. Ο κύριος Χουντής παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ναι, ναι. Έχω το λόγο, μπορώ να συνεχίσω. Εκ μέρους της ΚΟΕ, ως σκιώδης συγητής θα ήθελα, ναι, θα ήθελα να πω πολύ λίγα σύντομα λόγια για να μπορέσουν να μιλήσουν και άλλοι συνάδελφοι. Καταρχήν ε, θεωρώ ανάγκη και υποχρέωση να ευχαριστήσουμε τον εισηγητή τον ε, συνάδελφο τον κύριο Ντομένιτσι, διότι έχει κάνει μια πάρα πολύ σοβαρή και επίπονη δουλειά από ό,τι φαίνεται, την οποία πρέπει να προσεγγίσει κανείς με πολύ προσοχή, σεβασμό, προκειμένου να συμφωνήσει ή να μην συμφωνήσει μαζί του. Η δική μας η άποψη είναι ότι ε, η έκθεση, το σχέδιο που καταθέτει ο κύριος συνάδελφος είναι σε θετική κατεύθυνση και την υποστηρίζουμε. Είναι γεγονός ότι το θέμα της φορολογικής απάτης και καταπολέμησή του δεν είναι εύκολο ζήτημα το ψήφισμα που κατατίθεται εξοραίζει τα πράγματα, ενώ η έκθεση του κυρίου συναδέλφου και οι τροπολογίες που καταθέτει νομίζω ότι βελτιώνουν προς το θετικότερο προφανώς την κατάσταση εφόσον γίνουν αποδεκτές. Επειδή δεν είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε πιο αναλυτική συνεργασία με τον κύριο συνάδελφο και εφόσον υπάρχουν νομίζω τα περιθώρια, εγώ απλώς θα ήθελα να πω ότι ενώ συμφωνούμε με τις τροπολογίες, υπάρχουν ορισμένες τροπολογίες, θα αναφέρω τους αριθμούς για την ατζέτα μας για να μην κουράζω τους συναδέλφους, τις οποίες θα θέλαμε να γίνει μια συζήτηση, να δούμε αν συμφωνούμε, αν ακριβώς καταλάβαμε αυτό που θέλει να πει ο κύριος συνάδελφος. Είναι τροπολογίες 17, 41, 42, 45, 46, 52, 53 και 56 κύριε συνάδελφε. Σε αυτές τις τροπολογίες για τις οποίες έχουμε ερωτήματα και καταρχήν επιφυλάξεις, θα σας παρακαλούσα στο μέτρο που έχουν δυνατόν να κάνουμε μια συζήτηση προκειμένου να, βρει, μια, να βρεθεί μια κοινή λύση εφόσον συμφωνούμε. Κατά τα άλλα, συμφωνούμε και υποστηρίζουμε την ε, έκθεση του κυρίου συναδέλφου και για άλλη μια φορά το συγχαίρω για την επίπονη υπογραμμίζω δουλειά που φαίνεται ότι έχει κάνει για να μας φέρει την έκθεση στην Επιτροπή. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, πρώτα απ' όλα θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή τον κύριο Ντομένιτσι για το ότι έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά και επίση συμφωνώ και με αυτό που ελέγχθη προηγουμένως ότι πράγματι υπάρχει μεγάλο περιθώριο ε, σύγκληση απόψεων ανάμεσα σε διάφορες πολιτικές ομάδες. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη γιατί η κυρία Ζολή ε, έχει πάει στην Αφρική και μου ζήτησε να μιλήσω εγώ εξ ονομάτό τη. Ε, τώρα, δεν θα παρουσιάσω όλε τι 26 τροπολογίε που έχουμε καταθέσει, απλά θα ήθελα να σχολιάσω ορισμένε ε, που έχουν κατατεθεί από άλλου, για να ξεκινήσει η συζήτηση. Πρώτα απ' όλα, αυτά που είπε η κύριο Κυρί, ελπίζω και εγώ ε, να μην ε, κακοποιώ το όνομά σας. Ε, κοιτάξτε, ε, εντυπωσιάζομαι, αλλά διαπιστώνω όλο και πιστώ ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε σε πολλά πράγματα. Κυρίως στις τροπολογίες αυτές που κάνατε εκ μέρου του ΕΛΚ. Εκεί όμω που διαφωνούμε είναι όσον αφορά αυτή την κοινή φορολογική βάση. αυτό τελικά αν γίνει και αν υπάρχει και κάθε έκθεση για κάθε ένα κράτος μέλος, ίσως να υπάρξει διαφάνεια. Για όσους εξημών ε, θέλουν τον ανταγωνισμό, εμείς πιστεύουμε ότι αν υπάρχει διαφάνεια θα υπάρχει και μεγαλύτερος ε, φορολογικός ε, ανταγωνισμός. Και αυτό τελικά θα ωφελήσει όλους. Το θέμα που τίθηκε πάλι είναι η διαφάνεια. Κοιτάξτε, εγώ θα έλεγα ότι η αναδυόμενες χώρες και στην Ευρώπη γενικά, αυτό όταν έχουμε κοινή φορολογική βάση, δεν σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε τον ίδιο φορολογικό συντελεστή. Ε, σαφώς και θα πρέπει να υπάρχουν διαφοροποιήσεις, καθότι πρόκειται και ε, διαφορετικό βαθμό ανάπτυξης ε, στα κράτη-μέλη. Ας πούμε, η Ουγγαρία ε, δεν θα πρέπει να βρεθεί σε δύσκολη θέση γιατί ε, θα ήταν αναγκασμένη να υποστεί ένα τέτοιο φορολογικό συντελεστή που δεν θα μπορούσε να τον δεχθεί η οικονομία της. Κατόπιν, σε σχέση με αυτά που είπατε, ε, που επικρίνατε τον ΩΣΑ, εγώ χτες είπα ότι ο ΩΣΑ δεν είναι ο χρυσός κανόνας ε, σε σχέση με τα φορολογικά. Και εσείς αναφέρατε, είπατε ότι οι 12 χώρες αν έχουν συναυθεί 12 συμφωνίες με ένα κράτος ότι αυτό είναι αρκετό. Για μένα δεν είναι ο που παίζει ρόλο. Το θέμα είναι ότι μπορεί κανεί να συνάψει οποιαδήποτε συμφωνία επιθυμία. Ας πούμε, αν η δική μου η χώρα, το Βέλγιο, συμφωνούσε με τη δική σας τη χώρα να τρώνε μαζί δύο φορές το χρόνο, αυτό είναι συμφωνία και είναι εντάξει. Αυτό όμως τι είναι αυτό, τίποτα δεν είναι, δεν λέει τίποτα για το περιεχόμενο της συμφωνίας. Βεβαίως ο ΣΑ την ανταλλαγή ε, των ε, πληροφοριών ε, μετά από έτοιμα την καθιστά κανόνα και εμείς δεν συμφωνούμε. Ε, πάω τώρα στις ε, τροπολογίες ε, που στήριξε η προλαλήσασα. Κοιτάξτε, συμφωνώ με τις επιφυλάξεις για την διαφύλαξη της ιδιωτικής σφαίρας. Κανείς μας δεν θέλει τα προσωπικά του στοιχεία να εκτίθενται στην κοινή γνώμη. Και η Βρετανική κυβέρνηση επέδειξε επιπολαιότητα με το να αφήνει να διαρρεύσουν αυτά τα στοιχεία. Αλλά και πάλι αυτό δεν αποκαλεί, αποτελεί λόγο για μας ότι επειδή η κυβέρνησή σας είναι ανίκανη εμείς να μην μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το μόνο εργαλείο που στη τελική ανάλυση είναι αποτελεσματικό, δηλαδή την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών. Επιτρέψτε μου να προχωρήσω και πιο πέρα. Ε, όταν θα πάρετε την κυβέρνηση διορθώστε τα. Η δική σα, η Βρετανική κυβέρνηση, εξ όσων γνωρίζω, είναι σε θέση να προστατεύει τα μυστικά για το που βρίσκεται το πυρηνικό σα υποβρύχιο όλο το χρόνο. Ε, φαντάζομαι ότι με τον ίδιο τρόπο θα μπορεί να προστατεύσει και τα φορολογικά μυστικά. Δεν υπάρχει τεχνικής φύσεως κόλλημα. ω εκ τούτου, μην το χρησιμοποιείτε κι εσεί ω πρόφαση για να παρεμποδίζετε την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών. Αυτά είχα να πω. Ε, ο κύριος ε, Σμιτ δεν είναι παρόν. Κατά τα άλλα, εμείς στηρίζουμε τις ε, τροπολογίες του. Ελπίζω να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση έγκαιρα για να διαφυλάξουμε και το κύριο μας απέναντι στην Κομισιόν και το Συμβούλιο σε θέματα φορολογικά. Κύριε Λάμπερτς, λέει η Πρόεδρος, όλοι μπορούμε ε, να κατηγορούμε μια κυβέρνηση ότι είναι ικανή, ανίκανη ή όχι, αλλά αυτά που ακούσαμε προηγουμένως έχουν ε, περισσότερο σχέση με την επιθυμία της κυρίας ε, να, της συναδέλφου να έρθει η δική της, το δικό της ακόμα στην κυβέρνηση. Ας περάσουμε λοιπόν στην κυρία Λούλινγκ, η οποία επίσης έχει καταθέσει τροπολογίες. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ο προλαλής σας δεν με έπεισε προφανώς. Για κανένα από τα ζητήματα που ανέφερε, ούτε βέβαια και για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών. Τέλος πάντων, χτες που συζητήσαμε τη διοικητική συνεργασία στο φορολογικό τομέα, τα είπα τα βασικά, οπότε τώρα θα περιοριστώ σε κάποια πιο συγκεκριμένα πράγματα σχετικά με τις τροπολογίες που έχω υποβάλει με την κυρία Φόρντα, με την οποία συμφωνώ βεβαίως πλήρως, για την ανταλλαγή πληροφοριών. Η θέση μου είναι εξή. Θα πρέπει να εφαρμοστεί το πρότυπο του ΩΣΑ με ομοιόμορφο τρόπο. Αυτό θα ήταν μια πραγματική πρόοδος. Γι' αυτό είμαι κατά της αυτόματης ανταλλαγής ε, πληροφοριών αδιάκριτα. Ή Τροπολογία 46, ξέρω αυτό το νόημα έχει. Ομοίω. δύο λόγια για το τραπεζικό απόρριτο. Είναι πολιτικό, πολιτικός μη ορθό και είναι αδίκως η πηγή κάθε κακού. Θα παραθέσω κάτι στη γερμανική. Το γεγονός ε, ότι το πρέπει να διαφυλάσετε το απόρριτο των πελατών των τραπεζών. Εδώ δεν γίνεται λόγος για το απόρριτο των τραπεζών, αλλά των πελατών. Και αυτό είναι θεμελιώδης δικαίωμα, ε, το δικαίωμα της ιδιωτικής σφαίρας. Ως εκ τούτου θα πρέπει να αναγνωρίζεται το δικαίωμα αυτό και για άλλους τομείς. Και κοιτάξτε, οι αριστεροί είναι εκείνοι που ε, κατεβαίνουν στους δρόμους ε, οποτεδήποτε μιλάμε για την ε, διαφύλαξη αυτών των ε, στοιχείων και για την ασφάλεια που πρέπει να επικρατεί. Αυτές οι σκέψεις αντικατοπτρίζουν ένα φιλελευθερισμό, η ελευθερία του ατόμου υπέρκειται της αυταρχικότητας των κρατών. Μία κοινωνία η οποία παρετείται επιπόλαια από την προστασία των ιδιωτικών στοιχείων του ε, πολίτη, η κυβέρνηση αυτή μπορεί κάλλιστα να διολυστήσει στον αυταρχισμό. Η άρση του απορρίτου θα πρέπει να λαμβάνει χώρα μόνο διακυβεύονται πολλά και σημαντικά θέματα ως ε, εκ τούτου αυτό είναι ένα στοιχείο που το ξεχνάνε πάρα πολλές φορολογικές αρχές. Είναι θέμα θεμελιώδους ελευθερίας λοιπόν. Το τραπεζικό απόρριτο είναι θεμελιώδης ελευθερία που δεν θα πρέπει να αμφισβητηθεί λόγω κάποιων καταχρήσεων. Δεν υποστηρίζω την φιλοσοφία που διέπει την έκθεση Ντομενίτσι. Πρέπει να μιλήσουμε εξάλλου για αυτό το θέμα και στην ε, πολιτική μου ομάδα, κάτι το οποίο δεν έχουμε κάνει. Ω εκ τούτου θα απόσχω από λεπτομερέστερες ε, προτάσεις για άλλε τροπολογίε και σχόλια. Κύριος Μπούλμαν. Ε, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι ο κύριος Ντομένιτσι μας παρουσίασε μια ιδιαίτερα ισόρροπη έκθεση, όμως δεν θέλω να μακρηγορήσω και θα ήθελα να παρακαλέσω τους συναδέλφους ότι όταν πρόκειται για φορολογικά θέματα να προσπαθούμε να επιδεικνύουμε συνένεση. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί κοιτάξτε, το κοινοβούλιο αυτό αγωνίζεται μεταξύ άλλων στο να μπορούμε να δίνουμε καλές συμβουλές εκεί όπου δεν έχουμε νομοθετικές αρμοδιότητες. Γιατί σε τελική ανάλυση η οικονομία αντιμετωπίζει τόσα πολλά προβλήματα που αν δεν βοηθήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν θα γίνει τίποτα. Αυτή είναι η δουλειά μας κατά κύριο λόγο. Κυρία Λούλινγκ, θέλω για άλλη μια φορά να σας πω, επειδή εδώ έγινε λόγος ε, για τα δικαιώματα ελευθερίας και τη σημασία του ατόμου από τη Γαλλική Επανάσταση. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, δεν πρόκειται εδώ για την απαλωτρίωση του τραπεζικού λογαριασμού. Πρόκειται για το γεγονό ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρχει απάτη και αποφυγή καταβολής φόρων δισεκατομμυρίων που δεν καταβάλλονται στον ε, εκάστοτε κρατικό κορβανά για να κάνουν τα κράτη-μέλη τη δουλειά τους. Αυτός είναι ο στόχος της ε, φορολογικής πολιτικής. Εμείς προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικότερα την φοροδιαφυγή. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να παρακαλέσω το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα να σκεφτεί και εκείνο κατά πόσον θα μπορούσε να δώσει κάποιες ε, σοφές συμβουλές στον εισηγητή τις οποίες και αυτό θα μπορούσε να δεχθεί. Κοιτάξτε, ε, θα σε έδινα το λόγο κύριε Λάμπερτ, αλλά δεν θέλω να ξεκινήσουμε τώρα τη συζήτηση για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών, γιατί την κάναμε χθε την κουβέντα σε τέσσερα δευτερόλεπτα. Κυρία Λούλινγκ, ήθελα απλώ να σα πω ότι είμαι και εγώ υπέρ τη ελευθερία, που θα πρέπει όμω να, είναι, ε, να πηγαίνει χέρι-χέρι με την ευθύνη. Ξέρω ότι και τα δύο είναι κοντά ε, στις αρχές σας και στο μέρος της καρδιάς. Ελευθερία λοιπόν με ευθύνη, με υπευθυνότητα. Ευχαριστώ που ήσασταν σύντομος. Κύριε Ντομένιτσι. Uh, και η ψηφοφορία για τις αρπολογίες θα είναι 11 Ιανουαρίου νομίζω. Θέλετε να σχολιάσει η Κομισιόν. Από εσά εξαρτάται, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο να σχολιάσει η Κομισιόν. Παρακαλώ, Κομισιόν. Έχουν υποβληθεί 59 τροπολογίε. Σας ακούμε. Ευχαριστώ. Και τι 59 δύσκολα θα μπορέσω να τις σχολιάσω. Κάποια σύντομα σχόλια παρόλα αυτά. Είναι επίμαχο το ζήτημα βέβαια και δημιουργεί δυσκολίε. Και είναι πολύ σημαντικό να μας υποστηρίξετε στην γενική άγουσα που έχουμε λάβει. Διότι η ανακοίνωση για τη χρηστή διαχείριση είναι μια γενική πολιτική. Και όπως είπαν ορισμένα μέλη, έχετε κοιτάξει άλλα στοιχεία του όλου πακέτου. Ας πούμε πρόταση για την αμοιβαία συνδρομή. κυρία Γκιόρη νομίζω ότι έχει δίκιο. Θα πρέπει να ακολουθήσουμε μια πρακτική θεώρηση των πραγμάτων. Γι' αυτό λέμε προς το Συμβούλιο ότι θα πρέπει να έχει μια σαφή και συντονισμένη πολιτική και εσωτερικά και εξωτερικά. Οι τροπολογίες που πηγαίνουν προς αυτή την κατεύθυνση είναι σαφώς ε, σωστές και εμείς θα τις υποστηρίξουμε. Υπάρχει σήμερα μια δοκιμασία του Συμβουλίου. Το ΕΚΟΦΗΝ καλείται να εγκρίνει να εξετάσει και να εγκρίνει κάποιες ε, προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα δούμε σε ποιο βαθμό το Συμβούλιο μπορεί να επιδείξει αραγές μέτωπο και συνενετικό πνεύμα. για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και των καταχρηστικών πρακτικών δεν θα πρέπει να μιλάμε γενικά. Δηλαδή, ένα πράγμα είναι τα μέτρα καταπολέμηση τη απάτης και άλλο πράγμα είναι οι συστημικές αλλαγέ που θα πρέπει να επιφέρουμε. Και τις στρατηγικέ εξόδου που θα πρέπει να διαθέτουν τα κράτη-μέλη. Παραλαμβάνω, δεν μπορώ να σχολιάσω όλες τις τροπολογίες. Χαίρομαι όμως από το γεγονός ότι επιδεικνύουν ε, τα μέλη τόσο μεγάλο ενδιαφέρον για τα θέματα αυτά. Και αυτό χρειαζόμαστε. Όχι μόνο γενικές κρίσεις και γενικές πολιτικές, αλλά και θέματα πρακτικά. Ευχαριστώ. Κύριε Ντομένιτση. Πέντε λεφτά, τα θέλετε, τα έχετε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ όλους όσους ομίλησαν και ιδιαίτερα αυτούς που ομίλησαν καλά για την έκθεσή μου. Θα ήθελα να σχολιάσω κάτι που είπε ο συνάδελφος Μπούλμαν. Κατά το έργο αυτό που αναλάβαμε, επαναλαμβάνουμε και επανεπιβεβαιώνουμε τη σημασία του ρόλου του Κοινοβουλίου σε ένα θέμα όπου δεν είμαστε ακόμα συνομοθέτες. Αυτό που είπε λοιπόν επ' αυτού ο κύριος Μπούλμαν για τη συνένεση είναι πολύ σημαντικό. Και συμφωνώ. Δύο παρατηρήσεις. Πρώτον, αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών. Και μιλήσαμε και χθες με αφορμή την έκθεση Άλβαρεθ. Ήδη λειτουργεί το μέτρο αυτό θετικά, με θετικό τρόπο μεταξύ των κρατών μελών. Απλώς μιλάμε εδώ για κάποια θέματα που αφορούν την προστασία των δεδομένων και ορισμένους κανόνες απορρίτου Υπάρχουν όμως ήδη αυτά. Υπάρχουν κάποιοι κανόνες περί αυτών. Ευχαριστώ τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής γιατί και εγώ αυτό το στόχο έχω με την έκθεση. Να προωθήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών όχι με στόχο να ελέγξουμε τους πολίτες αλλά να καταπολεμήσουμε καταχρηστικές, παράνομες πρακτικές. Αυτός είναι ο στόχος. Διότι αλλιώς θα δημιουργήσουμε μεγάλο πρόβλημα, πληγή. Ο συνάδελφος Φο, ή συνάδελφος Φόρντ, την οποία ευχαριστώ για αυτά που είπε, δεν ε, ε, έχει δίκιο. Διότι η περίπτωση που ανέφερε δεν αφορά την αυτόματη ανταλλαγή μεταξύ κρατών μελών. Έτσι. Αφορά άλλη περίπτωση. Τώρα για το corporate tax. Το κοινοβούλιο για τον φόρο επί των συναλλαγών. Ε, έχει εκφραστεί ήδη από αυτό και ιδιαίτερα το 2005 μέσω μιας εκθέσεως του συναδέλφου Μπερτσάνη εγώ συμφωνώ με αυτά που είπε ο συνάδελφος ε, Λάμπερτς. Ο στόχος είναι να έχουμε μία μέθοδο κοινή φορολόγησης των επιχειρήσεων που είναι κατεστημένες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και που έχουν διασυνοριακές δραστηριότητες. Όχι για να δημιουργήσουμε μειονέκτημα, αλλά για να δημιουργήσουμε πλέον έκτημα για αυτέ τι επιχειρήσει Και αυτό ε, που δεν, αμφισβητεί την ανεξαρτησία, την αυτονομία, την κυριαρχία των κρατομελών στα φορολογικά θέματα που συνεχίζουν να είναι τα μόνα αρμόδια για την έγκριση τέτοιων μέτρων. Υπενθυμίζω ότι από το 2005 στο 2008 εργάστηκε μια τεχνική ομάδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που καθυστέρησε λόγω του αρνητικού αποτελέσματος του πρώτου Ιρλανδικού δημοψηφίσματος και πολιτικά λοιπόν πιστεύω ότι σήμερα έχουν αλλάξει τα πράγματα και ότι θα πρέπει να επανενσκύψουμε επί του θέματος αυτό. Παρόλο που, και αυτές είναι οι τελευταίες μου δύο παρατηρήσεις, παρόλο που για το CCCTB θα μπορούσαμε να εισαγάγουμε ένα σταδιακό στοιχείο. Δηλαδή, οι επιχειρήσεις να έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν αυτό το καθεστώς σε μια πρώτη χρονική περίοδο. Και βεβαίως θα μπορούσαμε να προβλέψουμε την δυνατότητα της ενδυναμωμένης, της ενισχυμένης συνεργασίας. Κάτι το οποίο δημιουργεί ε, μια διαφορετική κατάσταση σε ό,τι αφορά τις σχέσεις μεταξύ των κρατών μελών. Σας καλώ να το σκεφτείτε. Σας ευχαριστώ εκ νέου για τη συνεισφορά σας και ελπίζω ότι με τον ίδιο θετικό τρόπο θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε και στο μέλλον. Και ευχαριστώ πολύ και τη συνάδελφο Γκέρι και τη συγχαίρω για τα καταπληκτικά Ιταλικά της. Καλώς. Σα ευχαριστώ. Κατά πάσα πιθανότητα θα ψηφίσουμε καν Ιανουαρίου. Ένα λόγο αν θα έχουμε τι ε, ακροάσει των επιτρόπων αυτό. Έχουμε πάντω προ το παρόν στην ημερησία διάταξη. Περνάμε τώρα στο επόμενο θέμα τη ημερησία διάταξη. Αλλά βλέπω ότι η ζωή δεν έχει φτάσει ακόμα. Ξέρει κανένα πότε θα έρθει. Να του δώσουμε καν δύο λεπτά. Γιατί έπρεπε να αρχίσουμε στις 11. This is the report on the 2009 annual... Αυτή είναι η τέτοια δήλωση για τη ζώνη του ευρώ 2009 και τα δημόσια οικονομικά. Πολύ σημαντικό θέμα για τις εργασίες της Επιτροπής μας και χθες είδατε το θέμα οι συντονιστές και το Προεδρείο, ξέρετε, ίσως συναντήθηκαν με την Τρόικα της Εκοφή. Ε, μια συνάντηση που πραγματικά εξέτασε το θέμα των δημοσίων οικονομικών και είμαι σίγουρη ο κύριος Γκίγκολ θα είναι πλήρως ενήμερος. Λοιπόν, συνάδελφοι. We restart the committee, our... Συνεχίζουμε τις εργασίες μας. Έφτασε ο εισηγητής. Θέλετε κανένα δύο λεπτά για να οργανωθείτε, κύριε ή Είσαστε έτοιμος. Επανάρχισουμε τη συζήτηση. Ο εισηγητής μας είναι εδώ, κ. Γκίκουλ, για την έκθεση για την ετήθεια σε δήλωση τη ζώνη του ευρώ 2009 και τα δημόσια οικονομικά. Κύριε Γκίγκουλ, έχετε το λόγο. Καταρχήν θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη για την καθυστέρηση γιατί εκ παραλλήλου λαμβάνει η χώρα η συνεδρία της αντιπροσωπείας ε, <clears throat> για τις Άνδρες και ο κύριος ε, Μαγκάλιο είναι ο πρόεδρος εκεί έχουν τους πρέσβες από την Κολομβία και το Περού που παρουσιάζουν ένα νέο, μια νέα συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών με τη ΣΥΠΑ πρόκειται για το θέμα ε, της καταβάσης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κλπ. Και εγώ έτσι πήγαινε ρόχομαι ανάμεσα στα δύο αυτά θέματα. Είναι τα προβλήματα αυτά των οργανωμένων συνεδριάσεων στην, ε, στο κοινοβούλιο γενικά. Δεν θα σα επαναλάβω όλα αυτά που έχω γράψει. Το πρόβλημα που έχουμε είναι ότι πρόκειται για ένα τεράστιο θέμα και πρέπει να αναφερθούμε με δύο λόγια σε αυτό. Και γι' αυτό χαίρομαι για τις μελλοντικέ σίγουρα τροπολογίες στην έκθεση όσο έχει σήμερα. Θα αναφέρω ορισμένα κεντρικά σημεία. Αυτό που αξίζει ιδιαίτερα να τονιστεί στην πρόταση Κομισιόν για την κατάσταση του Ευρωχώρου είναι ότι η Κομισιόν θεωρεί ιδιαίτερα σημαντικό το θέμα των ανισορροπιών. Δεν αναφέρεται αυτό παντού όταν συζητιέται αυτό το θέμα και γι' αυτό ε, όσα λέει η έκθεση και οι προτάσεις δικές μου αναφέρονται συγκεκριμένα σε αυτό το τομέα. Χαίρομαι γι' αυτό για τις περαιτέρω συζητήσει των προτάσεων και εδώ στην Επιτροπή μας και με την Κομισιόν και ίσως κάποια στιγμή και με το Συμβούλιο. Μία κεντρική πρόταση στην οποία θα ήθελα να αναφερθώ είναι τα μέσα του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης που θα πρέπει να τα εκμεταλλευτούμε για να αποφύγουμε υπερβολικά ελλείμματα ή και πλεονάσματα από τα κράτη-μέλη. Και με αυτόν τον τρόπο να μπορούμε να φτάσουμε σε μια πιο ομοιόμορφη εξέλιξη μέσα στα πλαίσια της Ευρωζώνης. Äh, äh, Κατά τη γνώμη μου, ένα θέμα πολύ κεντρικό εδώ είναι ότι μια αιτία για τις ανισορροπίες που είδαμε στις απλήσεις για τις κρίσεις ήταν η αύξηση των ε, κόστων ε, ε, περιουσιών. Πρέπει να εξετάσουμε το θέμα. Πολύ καλά θα έκανε η Κομισιόν για να σταθεροποιηθεί η οικονομική ανάπτυξη και για ενδυνάμωση της στρατηγικής εξόδου να ε, ακολουθήσει μία πολύ απαιτητική στρατηγική που θα προσπαθεί να περιοριστεί η εξάρτηση από ε, πόρους που πρόκειται να λήξουν για να απευθυνθούν έτσι και οι κερδοσκοπικές δραστηριότητες στον τομέα. Και έτσι θα δημιουργηθούν περαιτέρω θέσεις απασχόλησης και αηφόροι μελλοντικές βιομηχανίες. Όσον αφορά τον τομέα των δημόσιων οικονομικών, η βασική θέση θα πρέπει να υποστηριχτεί. Αυτό που αναφέρεται μέσα στα πλαίσια των υπερβολικών δραστηριοτήτων, ότι έχει κάνει η Κομισιόν μέσα στα πλαίσια του Συμφώνου Ανάπτυξης και Σταθερότητας, θα πρέπει εμείς να πούμε όμως ότι όλα αυτά δεν αρκούν. Ότι μετά από την έκθεση που υποβάλλει η Κομισιόν, όσον αφορά την κατάσταση των δημοσίων οικονομικών, είναι σαφέστατο ότι κάποια κράτη-μέλη μπορούν να έχουν τεράστιες δυσκολίες να αντιμετωπίσουν την κατάσταση με τα μέσα που τους δίνει όλο το σύστημα της Ευρωζώνης. Θα πρέπει λοιπόν εμείς να προσπαθήσουμε να βρούμε κάποιες λύσεις σε αυτό το τομέα. Αυτό είναι κάτι που προσπαθώ με τη δική μου πρόταση. Και έχω να πω ότι εδώ έχουμε ένα πρόβλημα για τα κράτη-μέλη και υπό την πίεση οικονομικών ανισιοτήτων. Και όσον αφορά τους περιορισμούς στον τομέα της φορολογικής συνεργασίας, να προσπαθήσουν να εξισώσουν, να εξορροπήσουν τους προϋπολογισμούς τους. Εκτός αυτού παρατηρούμε κάτι στην Ευρωζώνη που δεν θα πρέπει να υπάρχει σε μια νομισματική ένωση. Ότι δηλαδή τα διάφορα κράτη-μέλη έχουν διαφορετικά επιτόκια για την χρηματοδότηση του δημοσίου χρέους. Και εν ώψη αυτού η αρχή της ε, αλληλεγγύης μέσα στα πλαίσια της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης θα έπρεπε να μας οδηγήσει να μην έχουν κάποια συγκεκριμένα κρατημέλη τόσο μεγάλη επιβάρυνση στα δημόσια τους οικονομικά. Αυτό είναι και ένα πολιτικό θέμα, δηλαδή μια δυνατότητα ε, εξισορρόπησης των συμφερόντων. Αφενός υπάρχει ενδιαφέρον για καλύτερη φορολογική συνεργασία για να αποφευχθεί υπερβολική φορολογική, υπερβολικός φορολογικός ανταγωνισμός. Απ' την άλλη μεριά, ορισμένα δεν έχουν να αναλάβουν τόσο υψηλό κόστος και, κίνδυνο για τη χρηματοδότηση των ε, δημοσίων ελλημάτων. Εδώ λοιπόν θα μπορούσαμε να κάνουμε κάποια συμφωνία, ένα deal αν θέλετε, δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σας επ' αυτού. Θα ήθελα να σας πω και κάτι που δεν αναφέρεται. Δηλαδή το θέμα της διεύρυνσης της Ευρωζώνης σε περαιτέρω κράτη-μέλη. Ήδη στην πρώτη ανταλλαγή απόψεων είχα πει ότι κατά γνώμη αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Εγώ δεν το ανέφερα γιατί υπάρχει περιορισμό των σελίδων που μπορώ να γράψω, αλλά νομίζω ότι θα ήταν καλό, παραδείγματο χάρη, οι σκιώδεις συζητητές να μα πούνε κάτι από τη σκοπιά των δικών του ομάδων, πολιτικών ομάδων. Είναι δύσκολο το θέμα, περίπλοκο είμαι σίγουρο ότι θα υπάρχει μια ενιαία αντιμετώπιση. Αλλά η αρχή τη αλληλεγγύη θα απαιτούσε εμεί ω Κοινοβούλιο να είμαστε ανοιχτοί για το θέμα αυτό. Από την άλλη μεριά υπάρχουν σοβαρά οικονομικές δυσκολίες, δηλαδή κατά πόσο μια χώρα η οποία δεν έχει ακόμα σταθεροποιηθεί στην οικονομική της εξέλιξη, που μπορεί να περιμένει υψηλότερα ε, πληθωρισμό στο μέλλον, κατά πόσο θα πρέπει να ταχθεί επίσης με τους άλλους. Θα ήταν καλό λοιπόν αυτό το θέμα να το συζητήσουμε ανοιχτά και να δούμε ενδεχομένω πώς μπορούμε να θέσουμε κατά μέρο δυσκολίες και διαφορές των πολιτικών ομάδων για να συζητήσουμε το θέμα εις βάθος, γιατί αυτό αφορά μια βασική αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις αιτήσει των χωρών αυτών για ένταξη στην Ευρωζώνη. Αυτά προς το παρόν. Περιμένω να ακούσω τις παρατηρήσεις σας και ελπίζω μετά σε μια ανοιχτή συζήτηση συνενετικά να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να βελτιώσουμε την έκθεση. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, εγώ σας ευχαριστώ. Κύριε Γκέγκουλ, οι σκιώδες τώρα. Η κυρία Μπριάρντα Κούν. Ναι, σας ευχαριστώ πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι. Καταρχήν θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή, τον κύριο Google, για την ποιότητα της εργασίας του. Τον ευχαριστώ και προσωπικά, γιατί όταν είχαμε συναντηθεί είχε την ευγένεια να μιλήσει στα γαλλικά. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα. Τον ευχαριστώ επίσης γιατί έλαβε υπόψη κάποιες από τι παρατηρήσει μου, συμφωνήσει πάνω σε αυτή την έκθεση τώρα έχω να κάνω κάποιες παρατηρήσεις για θέματα στα οποία θα πρέπει να επανέλθουμε, ιδίως όσον αφορά την νομισματική πολιτική. όπου υπήρχαν κάποιες ενδιαφέρουσες προτάσεις. Εγώ όμως θα ήθελα να υπάρχει περισσότερη ε, μετριοπάθεια όσον αφορά την ε, μισθολογική ε, μέση οδό, η οποία σε ορισμένες χώρες οδήγησε σε αύξηση της ανεγνωστικότητας. Όσον αφορά την ε, νομισματική πολιτική της Κεντρικής Τράπεζας, εγώ συμφωνώ με τον ε, εισηγητή όσον αφορά την ε, σοφία της ε, Κεντρικής Τράπεζας, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο θα πρέπει να ξαναορίσουμε το τι εννοούμε με σταθερότητα των τιμών και ούτε κατά πόσο θα πρέπει να αναφερθούμε σε συγκεκριμένες πτυχές όπως την αναύξηση των ενεργών τιμών. Για τα δημόσια οικονομικά απορώ με την πρόταση του εισηγητή όσον αφορά ένα όριο που θα πρέπει να οριστεί στα υπερβολικά πλεονάσματα. Γιατί αυτό είναι δύσκολο μου φαίνεται να εφαρμοστεί και είναι και πάρα πολύ υπερβολικό. Από την άλλη μεριά όσον αφορά τα υπερβολικά πλεονάσματα και το υπερβολικό ε, δημόσιο χρέος Συμμερίζομαι απόλυτα την άποψή του εισηγητή κ. Γκούγκολ και την ε, αίτησή του για επαγρύπνηση. Κατόπιν, εγώ συμφωνώ για μια ενδυναμωμένη ευρωπαϊκή συνεργασία, αλλά το πρόβλημά μας παραμένει πάντα η ομοφωνία στο Συμβούλιο. Θα πρέπει όμως να προχωρήσουμε όσον αφορά την ε, εισαγωγή μιας ε, νομικής βάσης ο παγιωμένης για την φορολογήση των επιχειρήσεων. Χρειαζόμαστε νομίζω όπως προτείνει και ο κ. Γκέγκολ, μια ανοιχτή υψηλής ποιότητας συζήτηση και θα πρέπει βέβαια να συμφωνήσουμε και τι σημαίνουν τα ευρωχρεόγραφα γιατί αυτά είναι χρεόγραφα υπογράφουν, που εκδίδουν τα θεσμικά όργανα, πράγμα που δεν επιτρέπεται από τη συνθήκη. Από την άλλη μεριά έχουμε δάνεια σε ευρώ, που συνάπτουν διάφορα κράτη-μέλη. Αυτή η ιδέα θα μπορούσε να ήταν ενδιαφέρουσα. Θα πρέπει όμως να εξεταστεί πολύ προσεκτικά και να εξεταστεί πολύ καλύτερα στις ομάδες μας. Και ομολογώ ότι στην ομάδα μου στο ΕΛΚ δεν εξετάσουμε ακόμα το θέμα και μου φαίνεται ότι θα ήταν σημαντικό να το κάνουμε προσεχώς. Και θα ήθελα να έχω και την άποψη από τους παρόντες βουλευτές ε, όσον αφορά αυτό το θέμα που ξαναεπανέρχεται συνεχώς και μου φαίνεται πάρα πολύ ενδιαφέρον. Τέλος, όσον αφορά την εξωτερική εκπροσώπηση της ζώνης του ευρώ, συμμερίζομαι τις προσανατολισμούς του εισηγητή. Πραγματικά έχει έρθει το πλήρωμα του χρόνου η εκπροσώπηση της ζώνης ευρώ να ενωθεί, να διευκρινιστεί, να ενδυναμωθεί σε διεθνές επίπεδο. Αυτή είναι μια αιτήσια έκθεση που θα συζητήσουμε οπωσδήποτε στην ομάδα μου. Αλλά τα πρώτα στοιχεία από τις συζητήσεις είναι ακριβώς συγχαρητήρια για την πολύ καλή εργασία του κ. Γκίγκολτ. Ευχαριστώ. Πρώτα, εγώ σας ευχαριστώ. Ο κύριος ε, Φανγκόγκ. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Γκίγκολτ για την ποιότητα της εργασίας του, γιατί πρόκειται για μια πολύ φιλόδοξη έκθεση που αφορά όλες τις πτυχές της μακροοικονομικής πολιτικής της Ευρώπης, νομισματικής, ε, συναλλαγματικής ή ε, ε, εκείνη που αφορά τους προϋπολογισμούς ε, για τις ε, ε, ισοτιμίες θα πρέπει ίσως να το εξτάσουμε το θέμα έναντι του δολαρίου που ε, καταραίει και προβληματίζει πολλές από τις ευρωπαϊκές οικονομίες. Ακόμα και η Γερμανία έχει ένα πρόβλημα. Και θα ήταν λοιπόν καλό να καλέσουμε εμείς τη διεθνή κοινότητα να ξαναεξεταστεί το θέμα των ισοτιμιών μεταξύ των διεθνών νομισμάτων. Όσον αφορά την νομισματική πολιτική, όπως και ο κύριος Κίκουλτ, έτσι και εγώ είμαι πολύ ικανοποιημένος με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, που ήταν αντικυκλική, πραγματικά, δεν τη συζητάμε ίσως, αλλά ήταν αντικυκλική, ενώ των χιλιάδων δισεκατομμύριων ευρώ που πέρασαν σε τραπεζικά συστήματα για να αντιμετωπιστούν οι κρίσεις. Εγώ πιστεύω και ενδιαφέροντα από την σας ένας κίνδυνος να παρατηθεί η μισθολογική μετροπέδα στην Ευρώπη, γιατί πιστεύω πραγματικά ότι εν μέρει έτσι κατέρευσε η εσωτερική ζήτηση στην Ευρώπη. Η Γερμανία, παραδείγματο χάρη, αυτή τη στιγμή εξαρτάται μόνο από τις εξαγωγές της. Όσον αφορά τις αιτίε του πληθωρισμού, συμφωνώ στο αυτό που λέει η ότι ξεχάσαμε το θέμα του πληθωρισμού μέσω του κόστους γιατί ο πληθυσμός από τη ζήτηση δεν υπάρχει γιατί δεν υπάρχει επαρκής απασχόληση αυτή τη στιγμή υπάρχει πολλή ενεργεία και έτσι έχουμε πληθωρισμό μέσω του κόστους ε, δηλαδή του κόστου των πρώτων υλών κατά κατόπιν όσον αφορά τα δημοσιονομικά Εκεί κάποιες ε, πρέπει να διευκρινιστούν, αλλά θα το κάνω εγώ προσωπικά. Γιατί εγώ ε, ε, προετοιμάζω την έκθεση για τη μακροπρόθεσμη ε, εφορία των ε, δημόσιων οικονομικών. Έχω εντύπωση ότι τώρα μερικέ ε, δεν είναι σαφείς, γιατί η έκθεση του κυρίου Γκουγκόλ καλεί να υπάρχει μια νομισματική πολιτική αντικυκλική, από την άλλη μεριά όμως τονίζει και σε, περίπτωση, σε περίοδο οικονομικής ύφεσης τον απαράδεκτο χαρακτήρα του δημοσίου χρέους. Από την μεριά δεν πρέπει να ξέρουμε ότι τα δημόσια οικονομικά εξετάζονται μακροπρόθεσμα. Υπάρχουν περίοδοι δηλαδή, που υπάρχουν πλεονέσματα, υπάρχουν περίοδοι που υπάρχουν ελλείμματα. Και μου φαίνεται αντιφατικό να τονιστεί η αναγκαιότητα επιβολής κυρώσεων στις χώρες που σήμερα οδηγούν σε μια ανάκαμψη ήρθουν αυτά τα μέτρα ανάκαμψης πολύ νωρίς η ανάκαμψη και η αύξηση θα ε, σταματήσει και θα σταματήσουν και τα έλλειμματα. Γιατί αυτό είναι ο μόνο τρόπο για να μειωθούν, ο καλύτερο τρόπο για να μειωθούν τα έλλειμματα. Θα πρέπει λοιπόν να προσέξουμε τα μέτρα ανάκαμψη να μην αποσυρθούν πολύ συχνά. Εγώ δεν είμαι υπέρ του χρέους. Όχι, μην ε, με παρεξηγήσετε. Νομίζω ότι σε ε, περίοδο πλήρης απασχόλησης θα πρέπει πραγματικά να υπάρχει μείωση του χρέους, αλλά σήμερα υπάρχουν χώρες που ασκούν αυτό που λέγεται κακό χρέος, συλλέγουν κακό χρέος και είναι σημαντικό η Κομισιόν να αξιολογήσει την ποιότητα του χρέους. Το πόσο πρέπει για καλό χρέο ή για κακό χρέο. Και αυτό είναι ένα από τα σημεία στα οποία θα υποβάλουμε προτάσει, αλλά οπωσδήποτε πάνω προωθώντα την αντικυκλική αντιμετώπιση. Δηλαδή, όπω προβλέπει και το Σύμφωνο σταθερότητα του 2005, όταν υπάρχουν εξαιρετικές ε, περιστάσεις, να μην τηρήσουμε το 3% και το 60%. Και τώρα έχουμε πραγματικά εξαιρετικές ε, περιστάσεις γιατί έχουμε φέτος ένα μείον 4, μείον 5% στην Ευρώπη. Αυτές ήταν κάποιες ε, παρατηρήσεις που θα οδηγήσουν στις ε, τροπολογίες που θα υποβάλουμε. Πάντως εδώ βρίσκουμε πραγματικά πολύ επικοδηματικό πνεύμα έναντι της έκθεσης αυτής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριος Τρεμόζα, εκ μέρους του, των Φιλελευθέρων. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή τον κύριο Γκίγκαουλτ με τον οποίο κουβεντιάσαμε αρκετές φορές, ανταλλάξαμε απόψεις, συμφωνήσαμε επί πολλών, αλλά έχουμε και διαστάσεις απόψεων. Εμείς θα υποβάλουμε τροπολογίες, σίγουρα πριν το τέλη της εβδομάδας, γιατί ανησυχούμε για τα υπερβολικά, ας πούμε, δημόσια ελλείμματα εδώ θα πρέπει να δούμε σε τι χρησιμεύουν αυτά τα χρήματα. Δεν είναι το ίδιο να ξοδεύονται χρήματα που διονγκώνουν το δημόσιο έλλειμμα. Δεν είναι το ίδιο λέγω να πηγαίνουν για το εκπαιδευτικό σύστημα όπως κάνει η Γερμανία ή για να φτιάχνουμε πεζοδρόμια όπως γίνεται στην Ισπανία. Θα πρέπει λοιπόν να μας απασχολήσει αυτό. Πού διοχετεύονται αυτά τα χρήματα που δημιουργούν δημόσιο έλλειμμα. Και βεβαίως θα πρέπει να αποφύγουμε να γίνει φούσκα που θα σκάσει λόγω του δημοσίου έλλειμματος. Συμφωνούμε με τον εισηγητή ότι θα πρέπει η σταθερότητα των τιμών να επανοριστεί και να συμπεριλάβει και μια σκέψη το όλο θέμα για το τι γίνεται με τα περιουσιακά στοιχεία των ε, συναλλασσομένων στα πλαίσια της κρίσης. Η αύξηση των πιστώσεων θα πρέπει να βάλουμε ένα φρένο 20% το χρόνο αυξανόταν στην Ισπανία τα τελευταία πέντε χρόνια το, το επίπεδο των πιστώσεων. Η ισπανική φούσκα λοιπόν ε, είχε τραγικές συνέπειες ε, στον τομέα των ακινήτων αλλά ε, και στην Ευρώπη γενικά. Για τα Eurobonds θα πρέπει να μιλήσουμε επίσης. είναι δυνατή μια πραγματική ευρωπαϊκή πολιτική στον τομέα αυτό χωρίς ευρωπαϊκό ταμείο. Σύμφωνα με το αμερικανικό μοντέλο. Εγώ πιστεύω ότι η κοινή νομισματική πολιτική θα πρέπει να συνοδεύεται από, μια, από ένα μέτρο που θα ιδρύσει ή θα εδραιώσει μια εποπτική ενιαία αρχή. Τώρα, για τα ελλείμματα των τρεχόντων λογαριασμών. Και εδώ έχουμε αλλά δεν βλέπω πώς θα μπορούσαμε να περιορίσουμε ε, τις παρενέργειες. Η οικονομική βιβλιογραφία μας λέγει ότι ένα πρώτο βήμα για την έξοδο από την κρίση είναι η αύξηση των εξαγωγών. Οπότε δεν θεωρούμε ότι θα πρέπει να μπουν προστατευτικά φρένα και εμπόδια στις εξαγωγές. Δεδομένου ότι είναι απαραίτητες εξαγωγές για την διέξοδο από την κρίση. Κύριε Γκίγκαουντ, θα ήθελα να διαβάσετε το τελευταίο άρθρο του κυρίου Γκλούκμαν που επικρίνει την κινέζικη κυβέρνηση για τις παρεμβάσεις εις ό,τι αφορά την συναλλαγματική ισοτιμία του Ουάν στην ελεύθερη αγορά το συνάλλαγμα, η συνάγματική ισοτιμία είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο. Έχουμε πρόβλημα λοιπόν με χώρες που δεν σέβονται τις αρχές που θα έπρεπε να γίνονται σεβαστές για το θέμα αυτό. Το ανέφερε και ο τρόπος Αλμούνια σε ό,τι αφορά την υποτίμηση του One. Θα υποβάλουμε τροπολογίες και για άλλο λόγο. Ναι, λέμε στην φορολογική συνεργασία, αλλά έχουμε κάποια σχόλια για την φορολογική ανταγωνιστικότητα, για τον φορολογικό ανταγωνισμό καλύτερα. Ναι, λέμε ε, στην, ε, στον φορολογικό ανταγωνισμό. Δηλαδή, αυτό το οποίο ισχύει για τις επιχειρήσεις, ισχύει και για το δημόσιο, για τις δημόσιες αρχές και κυβερνήσεις. Ο ανταγωνισμός λοιπόν είναι φόλης της ύλη θετικός. Ο φορολογικός ανταγωνισμός εμπίπτει σε αυτήν την ε, κατηγορία. Μπορώ να σας δώσω κύριε Γκυγκάουλ την βιβλιογραφία από αυτού. Στις Ηνωμένε Πολιτείε οι περισσότερες επιχειρήσεις που είναι εισηγμένες στο Dow Jones βρίσκονται στο Delaware που έχει το υψηλότερο συντελεστή φορολόγησης των επιχειρήσεων. Τους χαμηλότερους ίσως να εννοεί ο, ο μιλητής συντελεστές φορολόγησης και όχι στη Φλόριδα όπου είναι εξαιρετικά υψηλή. Οι επιχειρήσεις λοιπόν βάζουν την φορολογική τους έδρα όχι μόνο με κριτήριο τον ε, συντελεστή αλλά και άλλα στοιχεία. Τέλος πάντων, όλα αυτά θα τα συζητήσουμε ξανά με τον εισηγητή με τον οποίο συνεργαστήκαμε ε, και θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε επικοδομητικά, είμαι σίγουρος. Ευχαριστώ. Ο κύριος ε, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον ε, εισηγητή για την έκθεσή του. Περιέχει πάρα πολλά και ενδιαφέροντα στοιχεία και συμφωνώ μαζί του ε, με τον ισχυρισμό του ότι στην Ευρωζώνη υπάρχει μια εσωτερική ανισορροπία η οποία μακροπρόθεσμα μπορεί να δημιουργήσει περαιτέρω προβλήματα. Η Ευρωζώνη είναι εκτεταμένη, είναι διαφορετικές οι οικονομίες μέσα στη ζώνη αυτή, ε, σε διαφορετική κατάσταση οι οικονομίες αυτές, το ενιαίο όμως νόμισμα δεν μπορεί να υπάρξει υποτίμηση ή οποιοδήποτε άλλο μέτρο θα μπορούσε να ληφθεί. <coughs> Βεβαίως και το ευρώ είχε θετικές ε, επιπτώσεις. Παρ' όλα αυτά όμως ε, εξακολουθεί να λοχεύει ο κίνδυνος ε, της ανισορροπίας και πρέπει να προσέξουμε. Όσον αφορά τώρα τη συγκράτηση των μισθών. Εδώ συμφωνώ με την εκπρόσωπο του ΕΛΚ. Η συγκράτηση των μισθών είναι ένα σημαντικό στοιχείο όταν μιλάμε για την οικονομική ανάκαμψη. Νομίζω λοιπόν ότι θα ήταν πολύ επικίνδυνο να εγκαταλείψουμε αυτήν την ιδέα και να αρχίσουμε να μιλάμε για αυξήσεις μισθών, οι οποίες όμως θα υποσκάψουν την ανταγωνιστικότητά μας. Στο σημείο υπαριθμών 15 ε, εκεί ε, θεωρώ ότι υπάρχει ε, κάποια αντιφατικότητα. Δηλαδή από τη μια γίνεται έκκληση για την προαγωγή των θέσεων εργασίας. Από την άλλη όμως αναφέρεται ότι θα πρέπει να εγκαταλείψουμε την ιδέα της συγκράτησης των μισθών και να καθοριστεί ένα κατώτατο μισθολογικό όριο και παράλληλα επενδύσεις και παράλληλα να λαμβάνεται υπόψη και το σύμφωνο τη ε, σταθερότητα και ανάπτυξη. Υπάρχουν λοιπόν τόσα διαφορετικά και αντιφατικά στοιχεία σε μία και μόνο παράγραφο που διερωτώ με αυτά είναι υπερβολικά. Είναι πάρα πολλά, είναι αντιφάσεις οι οποίε έχουν συμπεριληφθεί όλες ε, σε μία παράγραφο. Υπάρχουν και κάποια άλλα θέματα που θέλω να φέρω. Είπατε ότι ο ευρωπαϊκός προπολογισμό είναι πολύ περιορισμένος. Εγώ βρίσκω ότι είναι καλός, αρκετά μεγάλος και δείχνει και αυξητική τάση για το μέλλον. Αν όμως σε ευρωπαϊκό επίπεδο θέλετε να χαράξετε μακροοικονομική πολιτική, τότε πραγματικά χρειάζεται ένα τεράστιο προπολογισμό και πώς ε, πιστεύετε ότι θα τον ε, χρηματοδοτήσετε μέσα από ένα φόρο για την Ευρώπη, όπως το ζητάει εδώ και καιρό ο κ. Φερχόφστατ. Είναι ο κ. Φερχόφστατ ένας από αυτούς που το ζητεί αυτό εδώ και αρκετό καιρό. Και κάτι άλλο, πρόκειται για το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Εσείς λέτε ότι πρέπει να αναθεωρηθεί. Εγώ δεν νομίζω ότι πρέπει να αναθεωρηθεί, Απλά πρέπει να αναθεωρήσουμε λιγάκι τη στάση μας. Όταν λέμε ότι θα τον καταργήσουμε και θα ε, καταλήξουμε σε μια άλλη συμφωνία που θα είναι προσαρμοσμένη στις νέες συνθήκες, αυτό είναι λάθος. Το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης είναι καλό και εγώ είπα ότι θα πρέπει να αναλογιστούμε την κατάσταση, πράγματι ε, τα ελλείμματα των προπολογισμών ε, τα δημοσιονομικά ελλείμματα πρέπει να περιοριστούν. Όσον αφορά τώρα τα ευρωομόλογα, εγώ δεν είμαι πέρα αυτού γιατί κάτι τέτοιο θα σήμαινε την ε, ε, νέα μορφή χρέους και τα κράτη-μέλη είναι ήδη υπερχρεωμένα. Τώρα εσείς μιλάτε και για χρέη του συνόλου της Ευρώπης με τα ευρωομόλογα. Δεν συμφωνώ με αυτό. Θεωρώ λοιπόν ότι κατ' ουσίαν εδώ καλούμεθα να άρουμε ένα εμπόδιο το οποίο όμως μόνοι μας δημιουργήσαμε. Εγώ θεωρώ ότι δεν πρέπει η Ευρώπη να σκέπτεται το, την πιθανότητα των ευρωμολόγων. Εγώ είμαι οπαδός ε, της ε, πολιτικής του Φρίτμαν, ε, της, του δόγματος του Σικάγο. Έτσι λοιπόν ο συγητής θεωρώ ότι θα πρέπει να είναι λιγάκι πιο προσεκτικός, κυρίως όσον αφορά αυτό το θέμα της ε, συγκράτησης ε, των μισθών. Να προσέξετε λιγάκι αυτό, γιατί ε, θα προκληθεί περαιτέρω ανεργία, κάτι που δεν θα εξυπηρετήσει κανένα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Και εγώ ευχαριστώ τον κύριο Γκίγκολτ για μια ιδιαίτερα φιλόδοξη έκθεση. Δεν είναι εύκολο ε, σε ένα τόσο δύσκολο θέμα να εξετάσει κανείς ε, όλες τις πτυχές ε, που υπάρχουν. Αυτό για να το πράξει είναι κάτι πολύ φιλόδοξο. Έχω κάποια σχόλια που θέλω να κάνω. Καταρχήν στην παράγραφο, παράγραφο παριθμών 2 για την νομισματική πολιτική. και εμείς εγκρίνουμε την ε, νομισματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ε, βέβαια, εγώ θέλω να σας πω ότι η συγκατάθεσή μου ήταν και υπό κάποιες αιρέσεις, γιατί υπήρξαν πράγματι εποχές ε, όπου η τράπεζα δεν έλαβε παρακώς υπόψη στα στοιχεία της κρίσης και ως εκ τούτου θα μπορούσε ε, κανείς να δώσει την έγκρισή του, αλλά όπως είπα κάτω από κάποιες προϋποθέσεις. Όσον αφορά την παράγραφο υπαριθμών 5, εκεί θα πρέπει να αναφέρουμε και τους Κινέζους. Να τους συμπεριλάβουμε και αυτό σε αυτήν την εικόνα, την ε, ανταγωνιστικότητα που χάθηκε στην Ευρωζώνη. Αυτό δεν οφείλεται μόνο στο δολάριο, αλλά και στο νόμισμα της Κίνας. Και πρέπει αυτό να αναφέρεται. Παράγραφος 6. Δεν είναι σαφές τι ακριβώς εννοούμε όταν μιλάμε για την σταθερότητα των τιμών η οποία μπορεί να ε, συμπεριλαμβάνει και την έννοια την, το ενδεχόμενο της νέας αύξησης των τιμών ενέργειας και τροφίμων. Κοιτάξτε, αν ε, πρέπει να ληφθεί αυτό υπόψη. Αυτό έχει άμεση σχέση με την αναθεώρηση του προπολογισμού. Αλλά ενδέχεται ο κύριος Γκίγκολ να έχει κάτι άλλο κατά νου που πρέπει να μας το διευκρινίσει. Όσον αφορά τις ε, παραγράφους 11, 12 και 13, Νομίζω εδώ πράγματι δίκαιο έχει με τις ανισορροπίες, αλλά δεν ορίζονται επαρκώς οι ανισορροπίες αυτές. Ε, ως εκ τούτου, αυτές μπορούν να οδηγήσουν ε, σε ασάφεια. Παράγραφος 12, παραδείγματος χάρη, εκεί λέει ότι οι ανισορροπίες έχουν περιοριστεί κατά τη διάρκεια της κρίσης. Κοιτάξτε, τα ελλείμματα που δεν είδαν περιορίστηκαν, βεβαίως ε, ενδέχεται, εάν η έκθεση ορίσει με μεγαλύτερη σαφήνεια τη ανισορροπή, τότε να καταλάβουμε και καλύτερα την παράγραφο υπαριθμών 12. Όσον αφορά τώρα την ε, άρση της ε, πολιτικής ε, μισθολογικών συγκρατήσεων. Κοιτάξτε, η συγκράτηση μισθών, καλό είχε αυτό, είναι θέμα υπευθυνότητας. Το να αναστείλει κανείς κάτι το οποίο όμως είναι ένας υπεύθυνος τρόπος ε, που αντικατοπτρίζει ε, και την ε, παραγωγικότητα, το να θέλει κανείς να το αναστείλει αυτό είναι λιγάκι περίεργο. Ίσως θα έπρεπε να κάνουμε λόγο για την αναστολή των μέτρων και των κινήτρων. Ίσως θα μπορούσε κανείς να πει ότι αν αυτά τα μέτρα έχουν αποδώσει σε κάποιες χώρες τότε να συνεχιστούν αλλά ε, θα πρέπει να ε, αντιμετωπιστεί ιδιαίτερη περίπτωση των χωρών που είναι υπερχρεωμένες. Όσον αφορά την παράγραφο υπαριθμών 20, εδώ δεν είναι απόλυτα σαφές ή τουλάχιστον η έκθεση θα πρέπει να αναφέρει να είναι πιο συγκεκριμένη. Δεν μπορούμε γενικά να λέμε ότι ε, προτείνουμε το υπερβολικό έλλειμμα να διασφαλιστεί ότι τα κράτη-μέλη θα αποφεύγουν υπέρμετρα, ελλήμετρα και πλονοσματικά ισοζύγια. Να λέμε ακριβώς τι επιθυμούμε. Τέλος, πιστεύω ότι στην έκθεση θα πρέπει να αναφέρεται και το ότι στην Ευρωζώνη και τώρα και άλλοτε αλλά και τώρα προχωράει κανείς πάρα πολύ γρήγορα. Δηλαδή υπάρχουν χώρες που είναι περισσότερο πειθαρχημένες από άλλες και η το κομμάτι εκείνο των κρατών μελών που έχουν μεγάλα προβλήματα ε, δεν τα προβάλλουν με σαφήνεια και είναι δύσκολο να αντιμετωπιστούν. Αυτό είναι δύσκολο για το σύνολο της Ευρωζώνης. Άρα δηλαδή θα πρέπει να ε, εξηγηθεί λιγάκι η στρατηγική εξόδου, όπως το είπαμε και χθε. Πώς μπορούμε να συντονίσουμε την δημοσιονομική με την νομισματική πολιτική, κάτι που πρέπει να ζητήσουμε στην έκθεση αυτή, δηλαδή η δημοσιονομική πολιτική να λαμβάνει υπόψη τη ότι γίνεται στην νομισματική πολιτική και ίσως ε, θα πρέπει και να ε, προηγείται της νομισματική, όπω ακριβώ μα συμβουλεύουν οι, οι θύνοντες. Ε, για άλλη μια φορά λοιπόν αυτή είναι μια καλή έκθεση αλλά θεωρώ ότι θα πρέπει να εξεταστούν προσεκτικά τα διάφορα σημεία της έκθεσης. Και εμείς ευχαριστούμε λέει Πρόεδρος. Ε, κύριε Γκίγκολτ, ε, θέλετε να ολοκληρώσετε ένα μισό λεπτό. Μήπως μπορείτε να είστε σύντομοι. Κοιτάξτε, εγώ αισθάνθηκα ότι ο κύριος Γκίγκολτ ε, απευθύνθηκε σε μένα. Βέβαια εδώ αισθάνομαι μοναξιά γιατί εμείς δεν ε, ανήκουμε στην Ευρωζώνη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω αυτή την πρότασή σας ότι είναι σημαντικό να συζητήσουμε και για τις ε, χώρες που είναι εκτός Ευρωζώνης. Είδαμε και μιλήσαμε για το πώς η Ευρωζώνη βοηθάει τις αναπτυσσόμενες χώρες. Δεν μιλάμε όμως αρκετά για τις ε, χώρες εκείνες που δεν ανήκουν στην Ευρωζώνη. Κατά τη διάρκεια της κρίσης οι χώρες αυτές ε, αντιμετώπισαν πολλά προβλήματα. Ευχαριστώ πολύ για την πρότασή σας και εγώ ε, προτείνω η Οικονομική Επιτροπή αυτό το θέμα να το εξετάσει με μεγάλη προσοχή Εξ όσων γνωρίζω, ε, μετά από δύο εβδομάδες στο Στρασβούργο θα συζητήσουμε για το θέμα αυτό. Και έχω και άλλη μία παρατήρηση για αυτήν την έκθεση. Όσον αφορά τη σημασία της ενιαίας εκπροσώπησης της Ευρωζώνης, εδώ θα ήμουν πιο προσεκτική. Με τη συνθήκη της Λισαβόνας έχουμε πλέον την αναγνώριση της, ε, Ευρω, της Eurogroup. Εμείς δεν έχουμε αντίρρηση, αλλά το να αναλάβει, να λάβει μάλλον αυτή η Eurogroup αρμοδιότητες και να εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Ένωση προς τα έξω, αυτό απλά θα ενισχύσει τη διαίρεση που υπάρχει στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με τη συνθήκη της Λισαβόνας κάναμε ένα βήμα προς τα εμπρός και θα δούμε τι ακριβώς ε, θα γίνει με τον ύπατο εκπρόσωπο της εξωτερικής πολιτικής και με τον νέο πρόεδρο Τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα δούμε πώ θα λειτουργήσει αυτό. Πάντως εγώ είμαι σίγουρο ότι όλα αυτά δεν θα συμβάλλουν στη συνοχή. Το 2004 όταν προσεχώρησαν οι νέες χώρες ε, της ε, Κεντρικής και τη Ανατολική Ευρώπης δεσμεύθηκαν κάποια στιγμή να ε, υιοθετήσουν, να εισάγουν το ευρώ. Βεβαίω δεν έχουμε να επιδείξουμε πολλά και θετικά αποτελέσματα στον διάμεσο χρονικό διάστημα. Η δική μου η χώρα ε, τα χρόνια που μεσολάβησαν απλά απομακρύνθηκε από το σοσιαλιστικό μοντέλο διακυβέρνησης. Και είδαμε ότι ε, κατά την κρίση οι χώρες εκτός Ευρωζώνης αντιμετώπισαν περισσότερα προβλήματα. Αν λοιπόν ε, λέμε ότι προς τα έξω η Ευρωζώνη εκπροσωπείται ξεχωριστά, αυτό απλά βλάπτει την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη φήμη της και δεν θα ήθελα να ακολουθήσουμε αυτό το δρόμο. Θέλετε παρακαλώ να ολοκληρώσετε τη συζήτηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα αυτά τα σχόλια και ευχαριστώ και για την ε, θετική απήχηση που είχε η έκθεσή μου θα απαντήσω σε δύο-τρία θέματα. Καταρχήν, στο θέμα των ευρωομολόγων και στον επιμερισμό ε, του κόστους που προκύπτει από τα διαφορετικά επιτόκια. Ίσως ε, θα πρέπει να διευκρινίσω κάτι. Κοιτάξτε, εγώ δεν είπα ότι είμαι υπέρ της αύξησης του χρέους. Όχι, εγώ είπα ότι πρέπει να χρησιμοποιηθούν εργαλεία για τις χώρες εκείνες ε, που έχουν χαμηλότερο κόστος στην εξυπηρέτηση του χρέους, αυτές οι χώρες έχουν περισσότερα χρήματα για να επενδύσουν στην παιδεία, στην αηφορό ανάπτυξη και καθεξής. Δεν πρόκειται δηλαδή, δεν λέω να αυξηθεί περαιτέρω το ήδη υψηλό επίπεδο χρέους. Όταν τοποθετήθηκα θετικά για το Σύμφωνο Ανάπτυξης και Σταθερότητας και συμφωνώ με την Κομισιόν, ως προς το υψηλό επίπεδο του δημοσίου χρέους, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να αποσυρθεί η επεκτατική φορολογική πολιτική. Αυτό δεν αναφέρεται καν στην έκθεση. Κοιτάξτε, εδώ θα πρέπει να είναι σαφής η διαφοροποίηση. Πράγματι, ανησυχεί το επίπεδο του χρέους και ακόμα και για καλό σκοπό δεν μπορεί κανείς να προτείνει να αυξηθεί περαιτέρω το χρέος. Σε ορισμένα κράτη-μέλη δεν μπορεί κανείς να πει ότι ξέρετε επειδή είναι απαραίτητο να υπάρξουν επενδύξεις στην παιδεία γι' αυτό και θα αυξήσουμε περαιτέρω το ε, δημόσιο χρέος μας. Στην κατάσταση που βρισκόμαστε σήμερα δεν μπορούμε να προτείνουμε την άμεση απόσυρση αλλά αυτές οι διαδικασίες περί υπερβολικού ελλείμματος Αυτές έρχονται ε, καθυστερημένα. Το Σύμφωνο Σταθερότητας υπάρχει από το 2005 και επιτρέπουν τη λήψη, επιτρέπει τη λήψη κάποιων μέτρων. Δεν διαφωνούμε. Η Κομισιόν τώρα πρέπει να αντιμετωπίσει τη διαδικασία ελλημάτων για να έχει καλύτερες εξελίξεις στο μέλλον. Στη Γερμανία διαπιστώνω και υποφέρω από αυτό ότι η νέα κυβέρνηση ε, περικόπτει τους φόρους και αυτό μακροπρόθεσμα θα οδηγεί σε αύξηση του χρέους. Γι' αυτό είμαι ικανοποιημένο που έχουμε την Κομισιόν που εξισορροπεί λιγάκι κακές οικονομικές πολιτικές. Όσον αφορά τώρα σε υπερβολικά πλεονάσματα Άκουσα αυτό που είπατε, ότι αυτό που λέμε θα μπορούσε να ήταν ε, ιδιαίτερα ε, παρεμβατικό. Εννοούσε προφανώς. Μάλλον. Κοιτάξτε, ε, μιλάμε μόνο για λίμματα και δεν μιλάμε για πλεονάσματα. Ο κύριος Σικλούνα είπε κάτι το παρεμφερές όταν ανέφερε ότι η συγκράτηση των μισθών είναι κάτι το θετικό σε σχέση με την αύξηση της παραγωγικότητας. Συμφωνώ μαζί σας η εξέλιξη των μισθών θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στην, ε, στον πληθωρισμό και την παραγωγικότητα. Όμως βλέπουμε σε ορισμένες χώρες ότι οι μισθοί, δεν ακολουθούν αυτή την εξέλιξη. Είναι χαμηλότερες οι αυξήσεις επί των μισθών. Γι' αυτό είπα να εγκαταληφθεί η ε, μισθολογική συγκράτηση. Και να συνεχιστεί αυτή η πολιτική σε περίοδο κρίσης υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να εμφανιστούν ε, ενδείξεις αποπληθωρισμού. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να το αντιμετωπίσουμε το θέμα ε, που δεν είναι ο κλασικός τρόπος. Αυτοί που είναι ε, κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, θέλουν αύξηση μισθών και οι άλλοι, μάλλον με συγχωρείτε, αυτοί που είναι κοντά στα συνδικάτα θέλουν αύξηση μισθών και αυτοί που είναι κοντά στους εργοδότες θέλουν μείωση ή συγκράτηση των μισθών. Εγώ πιστεύω ότι εδώ πρέπει να έχουμε μια συζήτηση που ξεπερνάει αυτά τα αστερότυπα και αυτόν τον πόλεμο που κατά την άποψή μου δεν υφίσταται πλέον. Κανεί πλέον δεν μιλάει για υπερβολικές αυξήσεις μισθών, κανείς δεν θέλει αυτό. Από την άλλη όμως δεν θα πρέπει να τασόμεθα υπέρ των αποπληθωριστικών πιέσεων. Εγώ πιστεύω ότι έγιναν αρκετές θετικές παρατηρήσεις. Προφανώς συμφωνώ με αυτό που είπατε για την Κίνα, για την παράγραφο υπαριθμών 5. Επίσης πιστεύω ότι για το 2 μια διαφορετική διατύπωση και για την νομισματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ε, ξέρετε, ακριβώς για αυτόν τον λόγο αναφέρω εδώ μια συγκεκριμένη ημερομηνία. Ε, συμφωνώ μαζί σας, εγώ το λέω έτσι κάπως πιο διπλωματικά. Ε, με αυτό που είπατε πάντως συμφωνώ. Λοιπόν, όσον αφορά τον φορολογικό ανταγωνισμό, κοιτάξτε, ο ανταγωνισμός είναι πιο σκληρός όταν διεξάγεται και αφορά τις επιχειρήσεις και εκεί, από εκεί προκύπτει όφελος. Αλλά στη Γερμανία τουλάχιστον αυτό που μάθαμε από την πολιτική τάξη του Όκιν, του Μίκεν Μάλερ και πάρα πολλών άλλων εκπροσώπων αυτής της πολιτικής λέει ότι αν θέλει κανείς να έχει αγορά και ανταγωνισμό που θα αποφέρει ωφέλη για όλους παράλληλα πρέπει να υπάρχει ένα κράτος που ορίζει, ε, βάζει τα όρια και κατευθύνει. Αν όμως ε, το κράτος μέσα του, μόνο του δημιουργεί ανταγωνισμούς και Ας πάμε στο θέμα της ε, φορολογίας, όπου δεν μπορεί κανείς ε, να ε, εξαπατά απλά μεταφέροντας την έδρα του σε κάποια άλλη χώρα και, να, τη φορολογική του έδρα. Αυτό είναι κατά της αρχής μιας τέτοιας οικονομίας αγοράς η οποία χρειάζεται το κράτος για να ε, καθορίζει εκείνο το πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργεί η αγορά. Τώρα λοιπόν στην Ευρώπη είμαστε σε μια τέτοια φάση όπου ειδικά στον τομέα της φορολογίας έχουμε επιζήμιο ανταγωνισμό φορολογικής φύσεως και αυτό φαίνεται και από τον Hans Werner Zinn, ο οποίος είναι ένας από τους ε, ε, πιο μεγάλος υπέρμαχο ε, του νεοφιλελευθερισμού στη Γερμανία που λέει ότι όλα αυτά είναι υπερβολικά και δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με αυτόν τον τρόπο. Θεωρώ λοιπόν ότι για άλλη μια φορά πρέπει να αποφύγουμε αυτή τη στερεότυπη συζήτηση ανάμεσα σε αυτούς που θέλουν περισσότερους φόρους και τους άλλου που θέλουν λιγότερου ε, φόρου. Πρέπει να υπάρχει η ε, κυριαρχία των λαών που καθορίζει το επίπεδο της φορολογίας και οι ομάδες ε, της αγοράς δεν θα πρέπει να είναι εκείνες που θα καθορίζουν το ρυθμιστικό πλαίσιο. Θα μπορούσαμε να προσθέσουμε εδώ πάρα πολλά άλλα. Ε, ευχαριστώ πολύ για τα σχόλιά σας. Ήταν όλα ιδιαίτερα πολύτιμα και νομίζω ότι τελικά θα έχουμε μια ενδιαφέρουσα έκθεση. Ευχαριστούμε πολύ. Η καταληκτική ημερομηνία κατάθεση τροπολογιών είναι 8 Δεκεμβρίου θα τις εξετάσουμε στις 11 Ιανουαρίου, αν βέβαια συνεδριάσουμε εκείνη την ημέρα και θα ψηφίσουμε στις 26 Ιανουαρίου. Προχωράμε πολύ γρήγορα ε, γιατί έχουμε μόνο μισή ώρα για να εξετάσουμε την επόμενη έκθεση της ε, κυρίας Ιντβελτ. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Θα είμαι και σύντομη και απολύτως πιστική, οπότε δεν χρειάζεται καν να το συζητήσουμε. Εξάλλου είναι μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων μόνο οπότε δεν θα χρειαστεί χρόνος. Η έκθεσή μου είναι η ετήσια έκθεση για τις πολιτικές ανταγωνισμού. Παραδοσιακό αντικείμενο σχολιασμού από το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο κάθε χρόνο. Η φετινή έκθεση βεβαίως ως κεντρικό στοιχείο έχει τα σχέδια ανάκαμψης αλλά καλύπτουμε και κάποια άλλα θέματα εις ό,τι αφορά τα δικαστικά πρώτα. Προετοίμασα ένα πολύ ε, συνεκτικό κείμενο που είναι η βάση, το έναυσμα αν θέλετε, της συζήτησης. Οπότε καλό και τους σκιώδεις με τους οποίους υπάρχει μεγάλος βαθμός ε, για τα θέματα που θα πρέπει να θίξουμε αλλά και τους λοιπούς συναδέλφους να βασιστούν σε αυτό το κείμενο το οποίο που δεν είμαι θεωρείστε οριστικό για να υποβάλουν νέες προτάσεις και τροπολογίες. Ε, το δεύτερο ε, από το οποίο συμφωνήσαμε. Θέλουμε να τονίσουμε τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πολύ περισσότερο στον τομέα ε, αυτών που είναι σχεδόν αποκλειστικότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εμείς όμως ως εκπρόσωποι του λαού θέλουμε να έχουμε ένα λέγιν και για την πολιτική ανταγωνισμού. Δεν έχουμε βεβαίως στη διαθέσή μας κάποια επίσημα μέσα για να το κάνουμε αυτό, αλλά αν μη τι άλλο, αν μη τι άλλο, αναμένουμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ε, αναφερθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το follow-up αυτής της ε, συστάσεως και να μας εξηγήσουν πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα. Αυτό είναι βεβαίως οριζόντιο όπως λέμε ζήτημα. Πάγιο δηλαδή έτοιμά μας. Εις ό,τι αφορά τις κρατικές ενισχύσεις που είναι το βασικό ζήτημα. Οι κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις θα μπορούσε κανείς να πει ότι έχουν χρησιμοποιηθεί ως ένα ισοδύναμο μέτρο του toolkit της εργαλειοθήκης του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ. Δηλαδή, όχι μόνο ένας κουμπαράς που σπάει όταν έχουν οι επιχειρήσεις σε πρόβλημα και από τον οποίο αντλούνται χρήματα για να χρηματοδοτήσουν τις επιχειρήσεις που έχουν προβλήματα, αλλά και ως ένα πλαίσιο, ως μια γενική διαδικασία. Φαντάζομαι θα συμφωνείτε ότι τα τελευταία χρόνια ήταν απαραίτητη και επίγουσα κρατική παρέμβαση. Ε, φαντάζομαι από αυτού συμφωνούμε όλοι τώρα για το βαθμό παρέμβασης. Αυτό, ναι, ε, μπορεί να μην μας βρίσκει όλους σύμφωνους. Ότι όμως κάτι έπρεπε να γίνει αυτό ήταν σαφές. Δεδομένων των ποσών για τα οποία μιλάμε και των δημόσιων, του δημόσιου χρέους του δημόσιου ελλείμματος ε, που απέρευσε από αυτή την κατάσταση και πρόλαβα το τέλος της συζήτησης από αυτού του θέματος προηγουμένως καλούμε τους πολίτες να ελέγχουν πολύ προσεκτικά για ποια πράγματα ξοδεύτηκαν τα χρήματα αυτά που οδήγησαν στο δημόσιο χρέος. Την αποτελεσματικότητα αυτών των κονδυλίων, αυτών των πόρων. Την αποτελεσματικότητα και της λεγόμενης πράσινης ανάκαμψης ιδιαίτερα. Διότι πολλές από τις κρατικές ενισχύσεις δικαιολογούνται λόγω αυτής της ανάγκης ε, ριζικής ε, μεταστροφής προς μια πιο βιώσιμη ε, οικονομία, προς ένα πιο βιώσιμο περιβάλλον και προς μια πιο πράσινη οικονομία. Όντως έγινε αυτό, εγώ έχω τα ερωτηματικά μου. Τέλος πάντων μικρό ένα να κινδύνω. Το άλλο θέμα που ήθελα να υπογραμμίσω είναι ότι πρέπει να είμαστε σαφείς ότι είναι, αυτή είναι μια προσωρινή, περαστική κατάσταση. Υπάρχουν ήδη οι πρώτε ενδείξει τη ανάκαμψη. Γνωρίζουμε βεβαίω ότι ο δρόμο μέχρι την ε, εξηγένση είναι πολύ μακρύς. Πρέπει όμως ήδη από τώρα να σκεφτόμαστε κάποιες στρατηγικές εξόδου. Δεν μπορούν να διονυστούν αυτές οι κρατικές ενισχύσεις με την δικαιολογία ότι συνεισφέρουν στην ανάκαμψη. Κάποια στιγμή είναι απαραίτητε, αλλά κάποια στιγμή επίσης θα πρέπει να λήξουν. Τώρα για τις πολιτικές κατά τον τραστ και των μέσων που χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την κύρωση των ε, όσων στραβλώνουν τον ανταγωνισμό και ιδιαίτερα τον καρτέλ πολύ ψηλές κυρώσεις ε, επιβάλλει η Κομισιόν το οποίο έχει όντως αποτρεπτικό χαρακτήρα και αποτέλεσμα αυτό θέλουμε κι εμείς να είμαστε πολύ αυστηροί έναντι των όσων στραβλώνουν τον ανταγωνισμό αλλά θα πρέπει να σκεφτούμε μήπως το πλωστάσιο της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα μπορούσε να είναι έτσι κάπως πιο ε, εξελιγμένο, να μην είναι τόσο πρωτόγονο, δηλαδή να μην αρκείται μόνο στις κυρώσεις. Διότι κάποιες επιχειρήσεις, παρά τις τεράστιες προσπάθειες που έχουν ε, καταβάλει, πολλές φορές κυρώνονται λόγω του αποτελέσματος. Θα πρέπει λοιπόν να ε, θέσουμε αυτό το θέμα της ευθύνης των ατόμων όχι μόνο τη συλλογική ευθύνη τη επιχείρηση. Βέβαια, έχω επίγνωση του γεγονότο ότι είναι εξαιρετικά λεπτό και δύσκολο αυτό το ζήτημα. Και τέλος, για το χρονοδιάγραμμα, το οποίο βεβαίω είναι πολιτικό θέμα, θα πρότεινα θα πρότεινα λέγω να ασκήσουμε κάποια πίεση να εγκριθεί αυτή η έκθεση στην Ολομέλεια του Μαρτίου διότι υπάρχουν α, κάποιες εξελίξεις το Μάιο που θα προκύψουν με τη μορφή εξαιρέσεων για τα οχήματα με κινητήρα και κάποιες άλλες περιπτώσεις. Οπότε ξέρω ότι και άλλες επιτροπές θέλουν να γνωμοδοτήσουν από αυτών των θεμάτων, να συντάξουν εκθέσεις, οπότε καλό θα ήταν να συμφωνήσουμε φαινός χρονοδιαγράμματος, τόσο ώστε όλες οι επιτροπές να μπορέσουν να συμμετάσχουν στη διαδικασία χωρίς ε, συγκρούσεις και προβλήματα με τις ε, τροπολογίες. Αυτά. Ευχαριστώ. ο Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Ιντφέλτ για τη συζήτηση που έλαβε χώρα και πράγματι θέλω να πω ότι συμφωνώ απόλυτα μαζί της ότι η έκθεση αυτή πρωτοβουλίας έχει κάποιο περιορισμό στο χώρο ως εκ τούτου για ορισμένα βασικά θέματα του εσωτερικού δικαίου ε, δεν μπορούμε να αποφανθούμε παρά μόνο ακροθυγώς και πολύ σύντομα. Ε, λυπάμαι πάρα πολύ, όπως είπε και η συγγήτρια, ότι το 2008 ήταν ένα από τα έτη εκείνα κατά τα οποία είχαμε μεγάλες ε, παρεμβάσεις, ε, κρατικές παρεμβάσεις στις επιχορηγήσεις. Ας μην ξεχνάμε ότι από εχθές ισχύει η συνθήκη της Λισαβόνας, η οποία δίνει πλέον στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο περισσότερα δικαιώματα στη συναπόφαση. Και όχι μόνο αυτό, αλλά θα μπορούσαμε και να ξανασυζητήσουμε και την ε, συνθήκη του 81-82. Τέλος πάντων, εγώ θα ήθελα να είμαι σύντομος. Θεωρώ ότι ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από τη στιγμή που ε, κληθήκαμε σε αυτή την έκθεση πρωτοβουλίας να συμπεριλάβουμε ορισμένα θέματα, παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα κράτη-μέλη τους τελευταίους μήνες, ε, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να αντιμετωπίζουμε την πολιτική της Επιτροπής επικοδομητικά, να στηρίζουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε μεμονωμένες περιπτώσεις ίσως θα μπορούσαμε να πούμε ότι και εμείς μπορούμε να ε, βελτιωθούμε. Σε συζητήσεις με τον κύριο Μόσε από την Επιτροπή που σήμερα παρίσταται είδα ότι και η Κομισιόν ε, πρεσβεύει αυτό το πνεύμα. Εγώ έχω καταθέσει τροπολογίες και θα ήθελα να πω το εξής. Αυτά τα οποία έχει ήδη αποφασίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, παραδείγματο χάρη για το σημείο 18 τη έκθεση, εκεί θα πρέπει η διατύπωση να γίνεται με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Αναφέρομαι στην έκθεση Λένε, ε, την έκθεση του κυρίου Σκιώδη Συγητή, επίση, και προτείνω να αναφερθούμε και στο θέμα της συνεργασίας που αναφέρει η συγκήτρια συνεργασία των αρχών ανταγωνισμού. Εκεί να εστιάσουμε την προσοχή μας. Και για αυτό το λόγο, για αυτό το θέμα θα καταθέσω τροπολογίες εκ μέρου της πολιτικής μου ομάδας. Σε όλα τα άλλα θέματα που έθιξε η συγγήτρια, σχετικά με την κρατική πολιτική ε, παρεμβάσεων, σχετικά με τις ε, έρευνες ε, που έχουν ήδη διεξαχθεί ή αυτές που επίκυνται, εγώ προτίθεμαι να στηρίξω την έκθεση. Με τους ε, πράσινους έχουμε καταλήξει σε κοινή γραμμή και νομίζω ότι με την έκθεση αυτή μπορούμε να δείξουμε ε, σε μεγάλο βαθμό συμφωνία. Να δούμε όμως και τι θα γίνει σε σχέση με την Κομισιόν. Εκείνο που μπορώ να σας πω, ως σκιώδης εισηγητής ε, της Επιτροπής Κοινής Αγοράς, μπορούμε να προχωρήσουμε, όπως είπε η εισηγήτρια, με την έκθεση αυτή ε, καλύτερα να εμφανιστούμε προς τα έξω έγκαιρα παρά καθυστερημένα και εκ των υστέρων. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Σφάμπ. Ο κύριος Σάντσεθ. Ευχαριστώ. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για τη δουλειά της και το έγγραφό της που είναι μια πολύ καλή βάση εργασίας να σκεφτούμε και να αξιολογήσουμε την πολιτική ανταγωνισμού του έτος 2008. Η έκθεση θα πρέπει να είναι χρήσιμη σε όσους προσπαθούν να βγάλουν μια άκρη για το τι έγινε πέρσι κατά τη διάρκεια του έτους. Υπάρχουν και ορισμένα θέματα που αφορούν το 2009 και το 2010, τα οποία όμως πιστεύω ότι θα πρέπει να συζητήσουμε σε άλλο πλαίσιο. Και βεβαίως θα πρέπει να αποφύγουμε να παραφορτώνουμε την Κομισιόν με εκθέσεις, ανακοινώσεις κτλ. Υπάρχει μια διαδικασία ετήσιας έκθεσης που αφορά τα πιο συγκεκριμένα και πιο σημαντικά ζητήματα. Βεβαίως και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να έχει μεγαλύτερο, πιο πρωταγωνιστικό ρόλο για λόγους δημοκρατίας, για λόγους διαφάνειας, για λόγους αποτελεσματικότητας. Η πολιτική ανταγωνισμού δεν αφορά άμεσα την ε, εσωτερική αγορά. Άρα συναπόφαση. Αφορά άμεσα τους καταναλωτές. Άρα πάλι συναπόφαση. Οπότε ο ρόλος μας θα πρέπει να ενδυναμωθεί. Όχι μόνο η ανάπτυξη, αλλά και ο ο καθορισμός της πολιτικής ανταγωνισμού θα πρέπει να εμπλέκει πιο ενεργά τη συμμετοχή του Κοινοβουλίου. Ιδιαίτερα που το 2009 ήταν το έτος της δημοσιονομικής και οικονομικής κρίσης. Όχι επειδή έμεινε στο περιθώριο η πολιτική ανταγωνισμού, αλλά επειδή συνεισέφερε στην σταθεροποίηση. Νομίζω ότι αυτό ε, θα πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Όλα τα μέτρα που λαμβάνονται στο πλαίσιο της οικονομικής κρίσης δεν θα πρέπει να θέσουν σε κίνδυνο την σταθεροποίηση, την σταθερότητα που είναι το πρώτο, η πρώτη εκ των ανουκάνευ προϋπόθεση για την ανάκαμψη. Αλλά θέλουμε επίσης να ασχοληθούμε και με το θέμα του moral hazard, όπως το λέμε, του ηθικού κινδύνου. Με τις υπερβολικές αποζημιώσεις ή τη μη συμμόρφωση με τις ήδη λιμένες δεσμεύσεις που έχουν λάβει επιχειρήσεις ή άλλες οντότητες. χωρίς βεβαίως να είμαστε επιθετικοί, να είμαστε χρήσιμοι για την εσωτερική αγορά και για τα συμφέροντα των πολιτών μας. Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο αυτής της ε, εκθέσεως είναι ότι για πρώτη φορά αναφέρεται ένα ιδιαίτερο κεφάλαιο για τα καρτέλ και τους καταναλωτές. Είναι σημαντικό αυτό να το τονίσουμε όντως, διότι καταδεικνύει, καταδεικνύει λέγω, ότι υπάρχουν πολλές καταχρήσεις που βεβαίως ζημιώνουν και την εσωτερική αγορά και τους καταναλωτές. Για τη Λευκή Βιβλό θα πρέπει να διατηρήσουμε, να συντηρήσουμε την συνένεση στην οποία καταλήξαμε από τη συζήτηση στην προηγούμενη θητεία απόφαση Και πρέπει να αποφύγουμε τις υπερβολές του βορειοαμερικανικού μοντέλου. Και θα πρέπει να λάβουμε συγκεκριμένα μέτρα για την προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών και των επιχειρήσεων. Υπάρχει κάτι άλλο. Ο διαχωρισμός της πολιτικής ανταγωνισμού με το ενεργειακό πακέτο το λεγόμενο. Αυτό θα πρέπει να μας απασχολήσει. συγκεκριμένα και σε βάθος. Τώρα, για κάποια πιο συγκεκριμένα θέματα. Για τα αυτοκίνητα. Για τα οχήματα με κινητήρα. Υπάρχει μια διαδικασία αναθεώρησης, σε ό,τι αφορά την εξαίρεση. Θα πρέπει και το Κοινοβούλιο να ενσκύψει επί του θέματος. να δούμε πώς μπορούμε να συνεισφέρουμε στην ανάκαμψη του τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας. Για τα πρόστιμα, για τις κυρώσεις, τα πρόστιμα ή κυρώσεις είναι πολύ δύσκολο ζήτημα. Λένε να εφαρμόσουμε την πολιτική του μπαστούνιου και του καρότου. Δηλαδή όταν δεν δουλεύει το καρότο να έρχεται το μπαστούνι. Αλλά με τα πρόστιμα τα υπερβολικά, ε, τα αστρονομικά πολλές φορές ποσά που ζητούνται μπορεί να δημιουργήσουμε το αντίθετο αποτέλεσμα. Εμείς θέλουμε να έχει αποτρεπτικό χαρακτήρα αυτό μεν, αλλά όταν πλήττονται οι ανταγωνιστικές επιχειρήσεις πλήττονται και οι καταναλωτές. Αν για κάποιος για οικονομικούς λόγους έχει περισσότερο κέρδος από ότι μάλλον παρά την, ε, την ε, αθέμητη ανταγωνιστικά συμπεριφορά του και παρά το πρόστιμο που θα πρέπει να καταβάλει υπολογίσει ως επιχείρηση ότι παρόλα αυτά λέω θα βγάλει ακόμα κέρδος ε, δεν θα έχει κανένα πρόβλημα να προβεί σε αυτήν την ε, αθέμητη συμπεριφορά. Πρέπει λοιπόν να το σκεφτούμε περισσότερο με βάση το πρακτικό αποτέλεσμα στο οποίο θέλω να καταλήξουμε χωρίς δειγματισμούς, χωρίς δόγματισμούς επί του θέματος αυτού. Για τις κρατικές ενισχύσεις δεν με απασχολούν ιδιαίτερα. Είναι θέμα κάθε κράτους μέλους. Η γενική τάση μέχρι την ε, κρίση ήταν πτωτική. Δηλαδή μειωνόντουσαν συνέχεια οι κρατικές ενισχύσεις. Τώρα είναι εξαιρετική η κατάσταση. Τέλος, θα ήθελα να πω ότι είμαι στη διάθεση όλων για να συνεργαστώ με τους συναδέλφους Σκιώδης και βεβαίως με την εισηγήτρια. Έχω κάποιες απόψεις, κάποιες ιδέες ε, και νομίζω ότι θα μπορέσουμε με τη συνεργασία όλων να καταλήξουμε σε ε, πολύ καλά αποτελέσματα. Σα ευχαριστώ κύριε Σέντσε. Ο κύριο Φίλιπ Λόμπερ, των Πρασίρων. Ευχαριστώ πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Σοφή για την καλή συνεργασία και για το πνεύμα με το οποίο το συνέταξε. Δηλαδή δεν εξτάζεται μονάχα το παρελθόν, αλλά αναφέρεται ότι θα πρέπει να γίνει στο μέλλον. Μόνο έτσι θα εισακουστούμε εξάλλου. Α αρχίσουμε με αυτό που πρέπει να προηγηθεί. Όταν αναφέρομαι ότι θα πρέπει να μπλακεί περισσότερο το κοινοβούλιο από ό,τι μέχρι τώρα, τώρα έχουμε μια καλή ευκαιρία. Έχουμε τον Ιωακή Μαλμούνια που έχει οριστεί ε, για τη θέση αυτή και θα έρθει εδώ ενώπιον ημών. Θα πρέπει να δράξουμε τις ευκαιρίες για να μας δηλώσει θα αναλάβει δεσμεύσεις και στο παρελθόν ήταν πολύ καλός ε, κατά βάση στη σχέση του με το Κοινοβούλιο και πώς θα μεταφέρει αυτή τη συμπεριφορά στη νέα του ιδιότητα γιατί υπάρχουν διαφορετικές ε, ε, παραδόσεις στις διάφορες ε, γενικές διευθύνσεις ε, της Κομισιόν μέσα στο παρελθόν η αρμόδια αυτή ε, γενική διεύθυνση δεν είχε συνεργαστεί τόσο πολύ μαζί μα, αλλά ο κ. Σαλμούνια φαντάζομαι ότι θα φέρει ένα νέο αέρα να πνεύσει εκεί. Έχω πολλέ παρατηρήσει συγγνώμη Σοφή που τα έχει ακούσει ίσω στο παρελθόν, αλλά δεν τα, κόσουν, δεν τα έχουν ακούσει ίσω όλοι όσον αφορά τι ε, κρατικές ανισχύσεις. Ε, καλό είναι, αλλά δεν θα πρέπει να το αναβάλουμε Φέρουμε πάντα σαν κάτι αρνητικό. Θα πρέπει να γνωρίσουμε ότι βοηθούν να βγούμε από την οικονομική ύφεση. Επίσης πριν από 30 χρόνια πούμε, δημιουργήθηκε το, η εταιρεία Airbus με κρατικές ενισχύσεις. Τώρα όμως είναι ελεύθερο να πετάξει μόνο του. Δεν εξαρτάται. Λοιπόν είναι θέμα μάλλον μορφής και όχι ουσίας. Η στρατηγική εξόδου συμφωνώ θα πρέπει να παρουσιαστεί τώρα. Το μόνο σχόλιο που θέλω να κάνω είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει συντονισμένη προσπάθεια. Δηλαδή οι κυβερνήσει θα πρέπει να αποφασίσουν τι δικέ του ε, πολιτικέ εξόδου, αλλά η προετοιμασία θα πρέπει να γίνει σε συνεργασία και με του κοινωνικού εταίρου τουλάχιστον. Εργοδότε και εργαζόμενοι θα πρέπει να συμμετάσχουν αν θέλουμε να γίνουν αποδεκτέ οι στρατηγικέ αυτέ εξόδου. Ανταγωνισμός και πολιτική κατά τον τραστ. Ναι, εντάξει, για τις καιρώσεις να υπάρχει μεμονωμένα ε, η ευθύνη Δεν υπάρχει τίποτα που είναι 100% σίγουρο βέβαια, αλλά από την άλλη μεριά κατά βάση είναι η δική τους ευθύνη να εξασφαλίσουν οι επιχειρήσεις ότι οι εργαζόμενοι τους εργάζονται όπως πρέπει. Μετά θα πρέπει να δούμε κατά πόσον οι παραβάτες μπορούν να αποκλειστούν από την υποβολή σε δημοσίους διαγωνισμούς. Εγώ ενοχλούμαι από το γεγονό ότι η Microsoft, παραδείγματος χάρη, εξακολουθεί να είναι ένας από εκείνους που συμβάλλει στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρόλο που θεωρείται μία από τις χειρότερες επιχειρήσεις. Άμα δείτε δηλαδή του επέβαλαν ένα πρόσημο ενός δες. Ίσως ε, οικονομικά δεν πλήττονται οι επιχειρήσεις αν δεν μπορούν να υποβάλλουν σε δημόσιους διαγωνισμούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά όμως είναι ε, σαν ε, ένα δείγμα δυσπιστίας πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης, όταν είχαμε αυτή τη συνάντηση μεταξύ των σκιωδών εισηγητών, είχα την εντύπωση ότι αυτό που εμείς θεωρούμε σαν ανταγωνιστική πολιτική ε, δεν μας κάνει να ξεχνάμε ότι θέλουμε να διατηρήσουμε την δυνατότητα επιβίωσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Γιατί οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις πλήττουν περισσότερο από τον κόσμο με τα σκοτώνοντας φυσικά. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι ο κρογονίος λίθος της οικονομία μας. Η ΜΜΕ και θέλουμε να παραμείνει αυτό. Και τέλος, το πιο αντιφατικό θέμα είναι ότι πολλά συζητήσαμε αυτές τις τελευταίες μέρες για το θέμα του φορολογικού ανταγωνισμού και πιστεύω θα πρέπει πραγματικά να εξακολουθούμε να αποφύγουμε αθέμητο και βλαβερό φορολογικό ανταγωνισμό. Όταν συζητήσαμε το προηγούμενο θέμα, εξετάστηκε αυτό το CCTV. Είναι οπωσδήποτε ένα τομέα στο οποίο θα μπορέσουμε να συμφωνήσουμε και πιστεύω θα πρέπει να βρούμε κατά κάποιο τρόπο ώστε να παραμένουμε όλοι ε, ε, στο θέμα αυτό γιατί οδηγεί πραγματικά σε μια στρέβλωση του ανταγωνισμού συμφωνούμε ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να παραμείνουν ανταγωνιστικά και να τα βραβεύουμε όταν ε, πάνε καλά. Και θα πρέπει να ανταγωνιστούν και σε αυτό που έχουν να προσφέρουν. Και να μην έχουμε μια, ένα ανταγωνισμό προς τα κάτω όσον αφορά τη φορολογία. Αυτά είχα να πω αυτή τη στιγμή. Και χαιρετίζω το επικοδηματικό πνεύμα με το οποίο γίνεται αυτή η συζήτηση και θα πάρετε από μένα κάποιες προτάσεις τροπολογίας εν το χρόνο. Ευχαριστώ. Πρώτα ευχαριστώ κύριο Λαμπέρ. Η κυρία Φεράρη έχει το λόγο. Θα ήθελα και να συγχαρώ τον εισηγητή για την ποιότητα της ε, εκθέσης της που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και δεν πρέπει να ξεχνάμε, το θέμα είναι πολύ πολύ πλοκό. Θα ήθελα να τονίσω μόνο κάποια σημεία. Όσον αφορά το σημείο 10, υπάρχει ίσως κάποια υπεραπλούστευση όταν προτείνεται ένα νέο ευρωπαϊκό ταμείο διάσωσης. Θα πρέπει ίσως να το επαναδιατυπώσουμε. Γιατί υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες προτάσεις αυτή τη στιγμή που δείχνουν να είναι ακόμη πιο συγκεκριμένε ίσως σαν ένα τελικό στόχο. Αλλά πέχουμε πάρα πολύ από αυτό και αν το διατυπώσουμε όσο έχει διατυπωθεί, ίσως ε, είναι κάπως αδύναμο και θα προτιμούσα να επαναδιατυπώσω και να ευθυγραμμιστώ καλύτερα με τις προτάσεις ε, της έκθεσης Λαοζιά. Να διευκρινίσουμε δηλαδή καλύτερα τι θέλουμε να πούμε ως κοινοβούλιο. Παράγραφος 12. Έχω κάποιες αμφιβολίες κατά πόσο ξεκάθαρα μπορούμε να πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επίσημα πραγματικά έχει βγει από την ύφεση. Εν μέρη είναι αληθές. Α, απ' την άλλη μεριά όμως ορισμένες χώρες της ε, Ένωσης αντιμετωπίζουν πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα. Και θα ήθελα εδώ να τονίσω τη σημασία να αναφερθούν οι εσωτερικές διαφορές και η πολύ διαφορετική συμπεριφορά που αυξήθηκε κατά τη διάρκεια της κρίσης. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ξανααντιμετωπίσει την δυνατότητα εναρμονισμένης ε, ανάπτυξης και όχι με μεγάλες διαφορές. Υπάρχει και ένα άλλο θέμα που δεν αναφέρεται εδώ, που είχαμε αναφέρει σε προηγούμενες εκθέσεις και που συζήθηκε συχνά μεταξύ βουλευτών ή και μάλιστα μεταξύ πολιτικών κατευθύνσεων και θα πρέπει να το εξετάσουμε στα πλαίσια μιας έκθεσης ιδίας πρωτοβουλίας. Πρόκειται για το θέμα των ασκουμένων που ορισμένε επιχειρήσεις εκμεταλλεύονται τους χρησιμοποιούν δηλαδή για να εργαστούν χωρίς να τους πληρώνουν. Και έχουμε κάποιες εταιρείες στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πραγματικά ανταγωνίζονται οι με τις δε, έχοντας το 80% του εργατικού του δυναμικού ως ασκούμενους, ως προσωπικό δηλαδή που δεν πληρώνουν. Αυτό είναι ένα θέμα που θα πρέπει επίση να αντιμετωπίσουμε, γιατί έχει καταστεί πολύ σύνηθες. Παράγραφος 19. Δεν ξέρω ακριβώς. Τι εννοείται εδώ, γιατί υπάρχουν κανόνες και εκείνοι που δεν ακολουθούν τους κανόνες πρέπει να τιμωρηθούν. Δεν ξέρω, θα πρέπει να δώσουμε ένα βραβείο σε εκείνους που συμπεριφέρονται σωστά. Ναι, η συμπεριφορά μια επιχείρηση μακροπρόθεσμα πρέπει να ληφθεί υπόψη, αλλά η διατύπωσή σας ε, με κάνει να έχω κάποια ερωτηματικά, δηλαδή πώς θα πρέπει να ε, δίνεται, να επιβραβεύει εκείνους οι οποίοι συμπεριφέρονται καλύτερα από του άλλου. Δεν ξέρω, έχω κάποιε αμφιβολίε για διατύπωση. Οικονομικέ κυρώσει και παραβάσει. Συμφωνώ με αυτό που μας εξηγήσατε προφορικά, αλλά έχω την εντύπωση ότι ο τρόπος με τον οποίο έχουν διατυπωθεί οι εν λόγω παράγραφοι οδηγούν σε κάποιες αμφιβολίες. Οι 22 παραδείγματος χάρη. Άμα τη διαβάσει κανένα δεν ξέρει ακριβώς ποιες είναι οι προτάσεις σας. Τονιακές ε, και τονιακές έρευνες. είναι οι τομεί στου οποίου θέλετε να αναφερθείτε. Θα ήταν καλό να κάνουμε μια σύσταση προς την Κομισιόν ότι ο, κάποιοι από αυτοί ε, θα πρέπει να οδηγήσουν σε κάποιες κατευθυντήριες ε, γραμμές ε, γιατί ακόμα και η αυτοβιομηχανία και άλλες βιομηχανίες πέρασαν από μια διαδικασία πολύ παράξενη γιατί η οριζόντια προσέγγιση ήταν τελικά πολύ εθνικιστική εκάστοτε. Και ίσως αυτό διηγηθεί σε πιο διαρθρωμένη σκέψη για τις βιομηχανίες αυτές. Γιατί αυτό το θα μπορούσε να γίνει μόνο όταν έχουν χρησιμοποιηθεί κάποιες εθνικιστικές μέθοδες σαν ένα διορθωτικό μέσο να περάσουμε σε μια ευρωπαϊκή σκέψη και ευρωπαϊκή αξιολόγηση. Εκτός από αυτές τις λεπτομέρειες όμως που σας παρουσίασα, νομίζω ότι η έκθεση σας συμπεριλαμβάνει πάρα πολύ θετικές πτυχές, ιδίως η ενδυνάμωση του ρόλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες πτυχές που αναφέρθηκαν από τους προλαλήσαντες και έτσι βλέπουμε ότι θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση τελικά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Παραδείγματο. Καλό είστε σύντομος. Ναι, ναι, είμαι σύντομος. Πολύ ωραία. Σε γενικέ γραμμέ συμφωνώ με την έκθεση τη κυρία Σινφέλτερ. Είναι πολύ καλό όταν υπάρχει μια ανεξάρτητη έρευνα για την ε, ε, με τον τρόπο με τον οποίο ε, εφαρμόζονται οι εθνικές ενισχύσεις είχαμε το πρόβλημα με την τράπεζα ΚΑΠΕΣΕΙ και άλλες θα πρέπει να δούμε λοιπόν ακριβώς τι γίνεται και γιατί γίνεται όσον αφορά τα Trust και τις κοινοπραξίες νομίζω ότι υπάρχουν ε, προβλήματα αν είναι και ερευνητή και ε, δικαστής ε, και δήμιος ταυτόχρονα η Κομισιόν. Θα πρέπει γι' αυτό να το ξετάσουμε νομίζω. Μετά να δούμε τα μέσα που υπάρχουν στην ανταγωνιστική πολιτική. Κυρώσεις, παραδείγματος χάρη, οικονομικές κυρώσεις που είναι πάρα πολύ ψηλές βλέπουμε ότι υπάρχουν και άλλες δυνατότητες, δηλαδή υπάρχουν μέτρα κατά μεμονωμένων ατόμων που έχουν κάνει αυτές τις ε, συνεννοήσεις. Γιατί η κύρωση επιβάλλεται στο σύνολο της επιχείρησης. Ίσως θα πρέπει να προβλέψουμε κάτι όπως γίνεται και στις ΗΠΑ που έχει σαν στόχο τον εκάστοτε ε, άτομο που έχει σφάλει. Μετά θα πρέπει νομίζω να μην ξεχνάμε και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εγώ 7 χρόνια εργάστηκα στην Εκτελεστική Επιτροπή και ομολογώ ότι η ανταγωνιστική πολιτική ήταν ένα θέμα του αρμοδίου επιτρόπου χωρίς περαιτέρω να συζητείτε στην Εκτελεστική Επιτροπή. Ίσως κάποια φορά τηλεφωνάει μια κυβέρνηση και κάτι πρέπει να γίνει. Αλλά στο συλλογικό σώμα των επιτρόπων δεν εξετάζεται ποτέ το θέμα της αναγνωστικής πολιτικής. Θεωρείται σαν κάτι το αυτονόητο και παραμένει στα χέρια πραγματικά του αρμοδίου επιτρόπου. Από την άλλη μεριά άλλες ε, γενικές διευθύνσεις έχουν πολύ διαφορετικό αντίκτυπο. Αυτή εδώ είχε αρκετό προσωπικό βέβαια και ίσως γι' αυτό δεν γίνεται και καμία συζήτηση στην Κομισιόν. Ίσως θα ήταν δυνατόν την Άνοιξη να οργανώσουμε μια ακρόαση βασική για την ανταγωνιστική πολιτική. Πού βρισκόμαστε, στο που θέλουμε να κινηθούμε κλπ. Πρώτα ευχαριστώ κύριε Επί. Έχουμε περάσει το δεκάμιση. Σας παρακαλώ να είστε πάρα πάρα πολύ σύντομοι. Ναι, ναι, ξέρω, και εγώ βιάζομαι. Γιατί θα έπρεπε να προεδρεύσω αυτή τη στιγμή κάπου αλλού σε μια άλλη συνεδρίαση. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομη. Υπάρχει μεγάλο ποσοστό συνένεσης νομίζω. Θα αναφθώ σε κάποια τα σχόλια που έγιναν. Πράγματι, θεωρώ ότι ένας από τους κύριους στόχους της έκθεσης θα πρέπει να είναι να υπάρχει μια στρατηγική που στρέφεται προς το μέλλον, πώς θα διαμορφωθεί η ανταγωνιστική πολιτική. Θα πρέπει να δώσουμε ένα πιο σημαντικό ρόλο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.